Okay, colleagues. We'll, we'll make a start. Να ξεκινήσουμε, αγαπητοί συνάδελφοι. Παρακαλώ να καθίσετε. Καταρχήν, να, να πω κάτι για τη θερμοκρασία στην αίθουσα. The temperature in the room. It's um, very, very hot. Ε, κάνει πάρα πολύ ζέστη. Από ό,τι φαίνεται στις 12 ήταν 50 ε, βαθμοί εδώ και τώρα έχει κατέβει η θερμοκρασία και τώρα εργάζονται οι τεχνικοί ώστε να είμαστε όλοι πιο άνετα. Και θα μιλήσουμε και για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν κάποιες δυσκολίες. Έτσι ίσως νιώσουμε και εμείς κοντά τους όλοι ελπίζω να μειωθεί η θερμοκρασία όσο προχωρά και η συνεδρίαση. Έχουμε πια κάποια πολύ σημαντικά θέματα σήμερα στην ημερήσια διάταξη. Καθυστερήσαμε λίγο για να αρχίσουμε. Θα ξεκινήσω με το σημείο 1, έγκριση της ημερησίας διάταξης. Υπάρχουν αντιρρήσεις ή σχόλια για την έγκριση της ημερησίας διάταξης. Όχι. Σας ευχαριστώ. Επίσης, έχετε λάβει τα πρακτικά των τελευταίων συνεδριάσεων και των συνεδριάσεων των συντονιστών. έχετε σχόλια για τα σημεία 2 και 3, παρακαλώ να τα γνωστοποιήσετε στην γραμματεία πριν από το τέλος της σημερινής συνεδρίασης. Διαφορετικά θα θεωρούνται εγκεκριμένα. Έχω κάποιες ανακοινώσεις για σας σήμερα το απόγευμα. Καταρχήν την Τετάρτη το πρωί αυτή την εβδομάδα όλα τα μέλη και το προσωπικό προσκαλούνται να συμμετασχούν σε μία ενημέρωση με την οργάνωση Concord για την, πρόκειται για την οργάνωση ομπρέλα όλων των ε, ΜΚΟ ανάπτυξης και θα συναντηθούμε από τις 10 ως τις 12 στο SP5G2. Νομίζω ότι θα σας σταλεί και μια επενθύμηση από τη Γραμματεία για την ενημέρωση αυτή, για την Τετάρτη. Επίσης, θα έχουμε συζητήσει στις Επιτροπές Περιβάλλοντος και Γεωργίας αυτή την εβδομάδα με τον Φρανς Φίλσλερ, πρώην Επίτροπο Γεωργίας. Είναι πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής που προετοιμάζει την κληρονομιά της Παγκόσμιας Έκθεσης 2015 που θα λάβει χώρα στο Μιλάνο και το θέμα είναι ενέργεια για τον πλανήτη και σύντηση του πλανήτη στις 5 Νοεμβρίου στις ε, 10 το πρωί. Και θα ε, είναι πάλι την Τετάρτη στην Επιτροπή Άγκρη στις 4 το απόγευμα. Όσοι θέλουν λοιπόν ε, να ακούσουν τα σχετικά με την παγκόσμια έκθεση, να παραβρεθούν στη συνεδριάσεις της Επιτροπής Ένβη ή Άγκρη. Σήμερα θα επικεντρωθούμε σε ανθρωπιστικές υποθέσεις πέρα από τη συζήτηση για πέρα από το 2015 Απλώς να φυστήσω την προσοχή σας ε, στις εβδομαδιαίες ενημερώσεις που στέλνει η Γραμματεία σε όλους τους βουλευτές για τα ανθρωπιστικά θέματα. Ποια είναι τα μεγάλα ζητήματα και πώς βοηθάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ χρήσιμη σύνοψη για το τι συμβαίνει. Έτσι λοιπόν να ζητάτε από το προσωπικό σας να σας υπογραμμίζετε τα θέματα αυτά κάθε εβδομάδα. Επίση η διάσκεψη των Προεδρών έχει διαλέξει τον νικητή του βραβείου Ζαχάροφ, τον Dr. Ντένις Μακέγγι. Είναι διάσημος γυναικολόγος που έχει βοηθήσει τα θύματα σεξουαλικής ε, βίας ε, στην δημοκρατία του Κογκό. Πολλοί τον έχετε συναντήσει και ξέρω ότι πολλοί έχετε υποστηρίξει το έργο του Δόκτωρ Μακουέγγι. Θα λάβει το βραβείο του 26 Νοεμβρίου στο Στρασβούργο και θα υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μαζί του τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου σε μια κοινή συνεδρίαση ΔΕΒΕ, ΑΦΕΤ και Ντρουά. Θα γίνει αυτό τη Δευτέρα το βράδυ. Αυτό είναι το τέλος των ανακοινώσεών μου. Δεν βλέπω να έχετε ερωτήσεις. Διαφορετικά πάμε στο σημείο 5, ανακοινώσεις της Επιτροπής. Η Κομισιόν έχει ανακοινώσεις. Όχι από ό,τι φαίνεται. Σας ευχαριστώ. Πάμε στο σημείο 6, ώρα των ερωτήσεων. Δεν έχουμε λάβει κάποιες ερωτήσεις από τους συναδέλφους. Να σας μεθυμίσω αν θέλετε να θέσετε κάποια ερώτηση στην Κομισιόν μπορείτε να το κάνετε αν στείλετε την ερώτηση τρει μέρες πριν από τη συνεδρίαση, τρει εργάσιμες μέρες. Περνάμε τώρα στο σημείο 7. Αφορά μια συζήτηση πολύ σημαντική, πολύ θα είδατε κάποιες εικόνες από τη Συρία αυτό το Σαββατοκύριακο και χθε το βράδυ στο BBC σοκαρίστηκα που είδα δολοφονίες χωρικών. Δεν έδειχναν τις πιο κτηνώδεις σκηνές ε, για το τι συμβαίνει στη Συρία. Όπως ε, ξέρετε υπάρχουν πάνω από 3 εκατομμύρια άνθρωποι που έχουν εγκαταλείψει τώρα τη Συρία και υπάρχουν πάρα πολλοί και εσωτερικά εκτοπισμένοι. Μαζί μας έχουμε το Γενικό Διευθυντή από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Ανθρωπιστική Βοήθεια και Πολιτική Προστασία, Κλάου Σόρσεν, και εκπροσώπους από δύο ΜΚΟ που εμπλέκονται ενεργά στην ε, Συρία και προσπαθούν να βοηθήσουν του εσωτερικά εκτοπισμένου να μετακινηθούν στι γειτονικέ χώρε τον Κάστεν Χάνσεν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφύγων και τον Ζιλ Ανσούλ από τον Ερυθρό Σταυρό. Είχαμε μία συζήτηση πριν λίγες εβδομάδες με την Κρυσταλίνα Τζιουρκίεβα, την πρώην Επίτροπο για την ανθρωπιστική βοήθεια και μας ε, μίλησε για μια τρομερή κατάσταση. Από ό,τι φαίνεται δεν έχουν βελτιωθεί τα πράγματα. Θέλουμε να ακούσουμε τι συμβαίνει επί τόπου από τους συναδέλφους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη συνεισφέρουν ε, στην παγκοσμία απάντηση. Πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν ενεργοποιηθεί μέχρι τώρα ε, για μέτρα ανακούφισης στη Συρία. Όμως εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλή η ανθρωπιστική βοήθεια στη Συρία και υπάρχουν, υπάρχει πρόβλημα πώς να φτάσουν τα χρήματα σε αυτούς που τα χρειάζονται περισσότερο. Θα καλέσω λοιπόν τους τρεις ομιλητές να πάρουν το λόγο και κατόπιν ε, οι βουλευτές θα έχουν την ευκαιρία να θέσουν κάποιες ερωτήσεις και να σχολιάσουν για τα όσα θα ακούσουν. Θα ακούσουμε και από την Κομισιόν τι συμβαίνει, επιτόπου, αν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα Καταρχήν λοιπόν θα δώσω το λόγο στον κύριο Κλάους Σέρεσεν για να μας παρουσιάσει τι συμβαίνει από την οπτική της Κομισιόν. Uh, Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ Λίντα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ παρά το γεγονό ότι το θέμα δεν είναι και το πλέον ευχάριστο. Πέραν αυτού, είναι πονίδιστο το γεγονός ότι και πάλι πρέπει να επανέλθουμε σε μια κρίση η οποία προφανώς ε, δεν ε, προβλέπεται να ολοκληρωθεί σύντομα ε, ανέφερες και εσύ ότι η Κρυσταλίνα Τζορτζιέβα ε, πολύ συχνά ε, ε, παρομοίαζε τις ανθρωπιστικές κρίσεις με καναρίνια στα ε, ορυχεία. Και πρέπει να σας πω ότι πραγματικά ε, εάν υπήρχαν καναρίνια σε ορυχεία πλέον θα είχαν πεθάνει πάμπολα διότι φαίνεται ότι η διεθνής κοινότητα δεν καταφέρνει να ξεφύγει από τη λογική αυτού του παιχνιδιού ισχύω και στην πραγματικότητα δεν έχει καταφέρει στερεότητα των ανθρωπιστικά ζητήματα ε, δεν θεωρούν ότι ε, είναι πάνω από τα προσωπικά του συμφέροντα και δεν θα ήθελα εδώ να αναφέρω συγκεκριμένα ε, ονόματα, αλλά νομίζω ότι η κατάσταση είναι πραγματικά τραγική. 58% υψηλότερο είναι το ποσοστό των ανθρώπων που χρειάζονται κατεπηγόντως ανθρωπιστική βοήθεια από ό,τι πριν από ένα χρόνο. Από το 6,8 εκατομμύρια ανέβηκε στα 10,8 εκατομμύρια σήμερα και έχουμε πάνω από 200.000 ανθρώπους ε, που 200.000 ε, νεκρούς, 6 εκατομμύρια παιδιά που χρειάζονται κατεπηγόντως ανθρωπιστική βοήθεια εντός της Συρίας και Έχουμε μεταξύ 1,6 και 2 εκατομμυρίων παιδιά ε, που δεν έχουν πάει σχολείο εδώ και ένα χρόνο ή και δύο χρόνια σε κάποιες περιπτώσεις βρισκόμαστε αντιμέτωποι με 4,7 ε, εκατομμύρια άνθρωποι που βρίσκονται σε περιοχές ε, δύσκολης πρόσβασης, ε, είτε βρίσκονται εκτοπισμένοι, είτε βρίσκονται σε περιοχές οι οποίες είναι αμφισβητούμενες και αυτό φυσικά αποτελεί τόσο μεγάλη πρόκληση από πλευράς ασφαλείας που είναι πολύ δύσκολο να φτάσει η βοήθεια σε αυτούς τους ανθρώπους. Και ταυτόχρονα κλιμακώθηκε η βία στην βόρεια-ανατολική Συρία με το Ισλαμικό κράτος ε, το οποίο πλέον ε, έχει τα όπως έχετε δει στην τηλεόραση. Επομένως ε, οι Σύριοι είναι παγιδευμένοι και καθυλωμένοι στα χωριά τους και διακινδυνεύουν πάρα πολύ σοβαρά τη ζωή τους αν τολμήσουν να βγουν έξω από αυτά τα στενά όρια. Βρισκόμαστε λοιπόν ενώπιον μιας κατάστασης ε, για τη Συρία, Συρία που ήταν μια χώρα που είχε μια μέση ανάπτυξη και πλέον έχει καταρρεύσει πλήρως ε, το σύστημα υγείας. Έχουν καταστραφεί ε, είτε ολοσχερός είτε εν μέρη νοσοκομεία μέσω των διαφόρων επιθέσεων και δεν ξέρουμε τι θα γίνει εάν δεν μπορούμε να παράσχουμε ακόμα και βασικές υπηρεσίες υγείας και για τους ενήλικες αλλά πρωτίστω για τα παιδιά και φυσικά ε, αρχίζει να ξεκινά αυτή η έννοια της χαμένης γενιάς. Ε, δεν υπάρχει σχολείο, δεν υπάρχουν ε, παροχές υγείας. Πού θα καταλήξουν αυτά παροχέ συμβαίνει. Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες στις γείτονες χώρες που έχουν καταφέρει εδώ και πάρα πολύ καιρό να διατηρούν τα σύνορά σκανδαλώδε αυτο ανοιχτά, αλλά αρχίζουν να στι γείτονε χώρε ένα σημείο καμπής και παρα πολυ καιρο να διατηρουν τα συνορα του ανοιχτα αλλα αρχιζουν να φτανουν σε ενα σημειο καμπή και αυτα Αν δούμε τι γίνεται στο Λίβανο, για παράδειγμα ο αριθμός των προσφύγων που έχουν περάσει τα σύνορα είναι τόσο μεγάλος και πιέζει τόσο πολύ τον κοινωνικό ιστό των συγκεκριμένων κοινοτήτων που ε, αρχίζουν και αυτοί και καταραίουν. Και ε, πρέπει να πω ότι δεν ε, ε δείχνω καμία κατανοησία, αλλά καταλαβαίνω ότι για μια κυβέρνηση και μια κοινωνία σαν το Λιβάνο είναι πάρα πολύ δύσκολο ε, να τηρήσουν την αρχή της μη επιστροφής και να διατηρήσουν ανοιχτά τα σύνορά τους, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν αυτές οι σφαγές και αυτά τα τραγικά γεγονότα καθημερινά δίπλα τους το συζητάμε εδώ και δύο χρόνια πλέον το ζήτημα. Είχαμε προβλέψει ότι θα καταρρεύσει τελείως ε, το κράτος του Λιβάνου και αυτά που έμαθα από το Βερολίνο την προηγούμενη εβδομάδα στη διάσκεψη είναι ότι ε, ανέφερε ο πρόεδρος ότι φοβάται ότι δεν θα μπορέσουν να αντέξουν για πολύ και ε, παρά το γεγονό ότι είμαστε ευγνώμονε που καταφέρνουν να διατηρήσουν ανοιχτά τα σύνορα, από την άλλη ήταν πάρα πολύ δύσκολο να επιχειρηματολογήσουμε με αυτού του ανθρώπου για να προσπαθήσουμε να έχουμε αναφορέ στη μη επιστροφή, στη μη επαναπροώθηση στο κείμενο, γιατί βρίσκονται σε ένα σημείο καμπή. Το αυτό ισχύει ε, λιγότερο ίσω και για την ε, Ιορδανία, είναι πιο σταθερή χώρα, έχουν περισσότερου πόρου, αλλά και αυτοί βρίσκονται αντιμέτωποι με μια τεράστια πρόκληση είδατε αυτά που είδατε στη τηλεοράσεις σας. Ε, έχουμε ακόμα επιθέσεις. Ε, ε, πριν από δύο εβδομάδες είχαμε βομβαρδισμούς. Είχαμε επιθέσεις. Αυτή τη στιγμή στην ανατολική πλευρά της Συρίας έχουμε περίπου 4 με 5.000 ανθρώπους που βρίσκονται καθολωμένοι βόρεια των συνόρων γιατί ενώ θεωρητικά τα σύνορα είναι ανοιχτά, στην πραγματικότητα δεν είναι και έχουν βρεθεί εκεί καθυλωμένοι ε, σε πολύ επισφαλείς συνθήκες ε, διαβίωσης ε, πραγματικά δίνουν μάχη απλώς και μόνο για να μπορέσουν να επιβιώσουν και κανείς ε, δεν μπορεί να κάνει και πάρα πολλά για να ε, τους ε, δείξει είτε μια πιο ασφαλή οδό ή να σταθεροποιήσει λίγο την κατάστασή τους. Έχουμε δώσει πάρα πολλά χρήματα και θα συνεχίσουμε να δίνουμε χρήματα τι να πω, αλλά εγώ διαμαρτύρομαι για τον προπολογισμό μα, το γνωρίζετε. Υπάρχει μια συζήτηση εν εξελίξη αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο. Η Επιτροπή Προπολογισμών ε, προσπαθεί να εξασφαλίσει περισσότερα χρήματα για τι ανθρωπιστικέ μα βοήθειε και πραγματικά προσεύχομαι να μα τα δώσουν, διότι όπω ε, πολύ σωστά είπε και εσύ, Λίντα, χρειάστηκε να γίνουν περικοπέ ε, στι συνολικέ μα δεσμεύσει φέτο σε σχέση με πέρσι, απλώ και μόνον γιατί φτάσαμε σε ένα ανώτατο όριο σε πιστώσει πληρωμέν, κάτι το οποίο σημαίνει ότι είναι αδύνατον να υπογράψουμε νέε συμβάσει, διότι όσοι από εσά έχουν ασχοληθεί με ανθρωπιστικά ζητήματα γνωρίζουν ότι αυτή τη στιγμή υπογράφεται η σύμβαση, θα πρέπει φυσικά να δοθούν τα κονδύλια αρκετά σύντομα. Δεν είναι σαν την κατασκευή ενό αυτοκινητοδρόμου που μπορεί να περάσουν δύο χρόνια, υπάρχουν μελέτε φυκτό, σκοπιμότητα και γίνεται και ο δημόσιο διαγωνισμό. Οι δικέ μα δουλειέ είναι άμεσε, γι' αυτό και χρειαζόμαστε φρέσκο χρήμα. Και ξέρω ότι μπορώ να βασιστώ σε εσά, στην Επιτροπή Ανάπτυξη, για να μα βοηθήσει, αλλά απλώ να σα πω ότι αν δεν λάβουμε αυτά τα χρήματα θα βρεθούμε σε μια πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Ε, σας παρακαλώ λοιπόν ε, να βεβαιωθείτε ότι θα μιλήσετε στους συναδέλφους σας ε, στην Επιτροπή Προπολογισμών ή και στη χώρα σας, ε, στα Υπουργεία Οικονομικών, από όποια χώρα και αν κατάγεστε, για να τα έχουν κατά νου αυτά τα κονδύλια, γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει αν βρεθούμε ξαφνικά την επόμενη χρονιά με μισό το προπολογισμό σε σχέση με το προηγούμενο και περικοπές τόσο μεγάλες που δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Ε, πραγματικά λοιπόν θα πρέπει ε, να δράσουμε και να είμαστε βέβαιοι ότι διαθέτουμε και τα κατάλληλα κονδύλια. Τώρα, ε, αυτό που βλέπουμε ότι γίνεται αυτή τη στιγμή στο βόρειο τμήμα του Ιράκ είναι φρικτό, διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιέζονται προς το Κουρδιστάν, ε, αν είναι Σιήτες καλούνται να πάνε ακόμα και στη Βασόρα, να κατέβουν νότια και ζουν εκεί με τους συγγενείς τους και φίλους, αλλά οι κοινότητες αυτές δεν έχουν τις δυνατότητες να τα απεξέλθουν που θα περίμενε κανείς. Επομένως υπάρχουν πιέσεις και εντός της Συρίας, αλλά υπάρχουν και αυξημένες ανάγκες στα σύνορα στο Ιράκ και πρέπει να μπορούμε πούμε, να τα αντιμετωπίσουμε αυτό. Όσον αφορά το κομπάνε και του ανθρώπου που διέφυγαν από εκεί, θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμή εδώ στις προσπάθειε τη Τουρκία που προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτή την μαζική εισρωή προσφύγων από την άλλη πλευρά. Από πολιτική σκοπιά είναι πολύ ακαθόδε το ζήτημα για αυτού. από χρηματοοικονομική σκοπιά είναι πολύ μεγάλη επιβέρενση και εμεί θα θέλαμε να δείσουμε ε, έστω ελάχιστη αλληλεγγύη, γι' αυτό λοιπόν και μετέφερα και κάποια κονδύλια εκεί. Βεβαίω είναι ευγνώμονε που εμεί εμείς ακόμα καταφέρνουμε τουλάχιστον να διοχετεύσουμε ουσιαστική βοήθεια ε, στη Συρία είτε ε, διασυνοριακά αλλά ε, πρωτίστως μέσα στη χώρα από τα νότια και πάνω διότι αναγνωρίζουν ότι αν εμείς μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τους ανθρώπους εντός της Συρίας εάν μάλλον δεν μπορέσουμε εμείς να αντιμετωπίσουμε τους ανθρώπους εντός της Συρία η πρόκληση να πάνε προς τα σύνορα θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα. Εγώ πραγματικά δεν βλέπω να τελειώνει αυτή η κρίση. Ε, αν δεν μπορέσει κάποιος να ασχοληθεί περισσότερο με την ε, ε Γενέβη, ε, εγώ εμπιστεύτηκα και τον Μπραήμι και τον Κόφι Ανάν, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε, ε, και εμπιστεύομαι και την ίνη αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε λύση. και θα καταλήξουμε σε χάος αν δεν μπορέσουμε να βρούμε μια λύση. Αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι όλοι οι μεγάλοι εκεί σκέφτονται ποιο είναι το συμφέρον τους. Και αυτό θα μας τυχιώνει για δεκαετίες, εάν δεν καταφέρουμε να ε, ε, ε, έχουμε και πάλι τον έλεγχο των πραγμάτων. Και αυτό είναι πέραν της ανθρωπιστικής με αλλά εγώ είμαι αυτός που μαζεύει εδώ το λογαριασμό, με αυτούς τους καλούς ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν, αλλά χρειαζόμαστε και μια πολιτική λύση. Δεν μπορεί να συνεχιστούν έτσι τα πράγματα. Θα σταματήσω τώρα, Λίντα. Συγγνώμη αν ήμουν λίγο παθιασμένος, ε, αλλά είμαστε στις 3 Νοεμβρίου. Αν ε, βλέπετε τις ειδήσει, ε, προφανώς και αισθανόμαστε πόσο κατεπίγουσα είναι η πολιτική τράση και βλέπουμε ότι πραγματικά ε, κατασφαγιάζονται ολόκληρα χωριά λόγω των διαφορετικών θρησκευτικών του πεπιθήσεως. Και όπως είπατε, η εικόνα έχει διαμορφωθεί με πάρα πολύ δύσκολο τρόπο. Έχετε λοιπόν τον χάρτη που δείχνει τους αριθμούς των εκτοπισμένων ανθρώπων. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο στην Τουρκία, 1,4 εκατομμύρια στο Λίβανο. Μιλώντας λοιπόν για θέματα μετανάστευσης, καταλαβαίνετε το εύρος, την κλίμακα του προβλήματος. Για να μην αναφερθούμε καν στον αριθμό των εσωτερικά εκτοπισμένων μέσα στη Συρία. Και γι' αυτό λοιπόν χαίρομαι ιδιαίτερως που έχουμε εδώ μιλητές από μη κυβερνητικές οργανώσεις επιτόπου να δώσω πρώτα το λόγο λοιπόν στον κύριο Χάνσεν από το Νορβηγικό Συμβούλιο για τους Μετανάστες που δραστηριοποιούνται έντονα επί τόπου και μας έχει δώσει και κάποιες ε, σχετικά έγγραφα ενημερωτικά. Πείτε μας λοιπόν, μιλήστε μας για τις εμπειρίες από τη δική σας οργάνωση και τι πιστεύετε ότι χρειάζεστε, ποια βοήθεια χρειάζεστε, τι μπορούμε να κάνουμε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω εδώ στο φόρουμ αυτό. Θα ήθελα να κάνω μια σύντομη εισαγωγή για το Νορβηγικό Συμβούλιο Προσφύγων. Δραστηριοποιούμε στις 25 χώρες παγκοσμίω και παρέχουμε υποστήριξη σε πρόσφυγες και εσωτερικά εκτροπιστέντες σε περιοχές συγκρούσεων. Σε ό,τι αφορά την κρίση στη Συρία το NRC, το Συμβούλιο μας, παρέχει αρρωγή εντός της Συρίας αλλά και στις χώρες που υποδέχονται τους πρόσφυγες από τη Συρία. Λίβανο, Ιράκ, ε, Ιορδανία. Έχουμε πολύ προσωπικό επιτόπους, 1.400 άτομα υπάλληλοι άκοπα, ακούραστα δίνουν αυτή την ανθρωπιστική βοήθεια και ε, αυτό το έτος φτάσαμε τους 2,1 εκατομμύρια δικαιούχους. Κυρίως ε, εκπαίδευση, ε, τρόφιμα, ασφάλεια τροφίμων, παροχή αρρωγής το 2014 είχαμε περίπου the, the Syrian crisis, which is now into its... 110 εκατομμύρια ευρώ. Θα έπρεπε νομίζω καταρχάς να σχολιάσουμε τις χώρες που υποδέχονται τους πρόσφυγες και να τις ε, πενέσουμε. Αλλά αυτή η φιλοξενία τους ε, δεν σήμαινε ότι δεν υπήρχαν μεγάλες προκλήσεις και για την χώρα του πληθυσμού και για τη χώρα που υποδέχονται τους ε, πρόσφυγες και για τους πρόσφυγες. Μεγάλες οι προκλήσεις λοιπόν. Και φυσικά το αυξανόμενο κόστος για τα τρόφιμα για τα καταλήμματα. Αυτό δημιουργεί τριβές μεταξύ των κοινοτήτων και έτσι οι προκλήσεις αυτές που αντιμετωπίζονται καταρχάς η τάση είναι να περιορίζονται τα δικαιώματα των προσφύγων και κατά δεύτερον να περιορίζεται η εισρωή προσφύγων στη χώρα. Για τους λόγους που παρουσίασε και ο κ. Σόρενσεν, εκ παραλλήλου οι χώρες, οι όμορες ε, της Συρίας ε, επιτρέπουν περιορισμένο αριθμό επαναπατρισμών. Άρα, το κλείσιμο των συνόρων, ε, ο ακατάλληλος επαναπατρισμός και οι αυξανόμενες, αυξανόμενοι περιορισμοί για τους πρόσφυγες είναι τα τρία θέματα που με απασχολούν. Κοιτάτε τι γίνεται λοιπόν σε ό,τι αφορά το κλείσιμο των συνόρων. Υπάρχει το θέμα της σωματικής ε, ακεραιότητας και ασφάλειας ε, στα κέντρα αυτά η πρόσβαση σε τέτοιους περιφερειακούς δρόμους, η διαθεσιμότητα μεθόδων και μέσων ε, μεταφοράς. Ωστόσο, όλο και πιο σημαντικός φορέας κατατίσταται το θέμα των συνοριακών ελέγχων με την εξαίρεση της Τουρκίας σε ό,τι αφορά την εισρωή προσφύγων από το κομπάνι. Έχει περιοριστεί η προθυμία απορρόφησης προσφύγων και έχει μειωθεί δραματικά ο αριθμός των ε, προσφύγων που φεύγουν από τη Συρία. Αυτοί οι περιορισμοί σε συνδυασμό με την έλλειψη της ελευθερίας, ελεύθερης μετακίνησης ε, στη Συρία προκάλεψαν αναθεώρηση των σχετικών εκτιμήσεων του ΟΗΕ για το 2015. Περίπου 78.000 ε, πρόσφυγες κατά μέσο ώρες έχουν καταγραφεί για το 2014 από το UNCAGR. Οι μηνιαίοι αριθμοί για τον Οκτώβριο ήταν 18.000. Δραματική πτώση σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Κάποια παραδείγματα για τις χώρες που είναι γύρω από τη Συρία. Ο Λίβανος, τον Οκτώβριο του 2014 το Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι ο Λίβανος δεν επρόκειται να αποτεχθεί νέους πρόσφυγες στη χώρα. Πάνω από το 75% των πρόσφυγων στη Συρία ε, αποτράπηκαν από το να μπουν στη χώρα. Τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Η Ορδανία τώρα. Η Ιορδανία εξακολουθεί επισήμως να κρατά ανοιχτά τα σύνορά της, άτυπα και τα τυπικά της σύνορα στους πρόσφυγες από τη Συρία. Εισήχθησαν όμως περιορισμοί πριν από ένα χρόνο. Το Σεπτέμβριο του 2014 η κυβέρνηση της Ιορδανίας έκανε, έλαβε βήματα προκειμένου να είναι ουσιαστικά αδύνατη η προσχώρηση των προσφύγων στον βόρειο-ανατολικό στη βορειοανατολική Ιορδανία. Αυτό έχει σημαντικέ επιπτώσει για του Σύρου που θέλουν να φύγουν από την κατάσταση του εμφυλίου. Μόνο 250 άτομα κατέφτασαν μεταξύ τέλη Σεπτεμβρίου και αρχές Οκτωβρίου σε ένα κατάλημα στην Ιορδανία. Πολύ λιγότερο αριθμό από ό,τι αναμενόταν. Και έχουμε λοιπόν στην παρούσα φάση πάρα πολύ μεγάλο αριθμό άτομων που περιμένουν στα άτυπα σημεία εισόδου, περιμένοντας ανθρωπιστική βοήθεια και προστασία. Επισήμως δε η Τουρκία επιτρέπει να, να συνεχίσουν να έρχονται οι Σύριοι πρόσφυγες στην επικράτειά της, αλλά τα καταλήμματα για τους πρόσφυγες είναι όλο και πιο πλήρη και έτσι έχει αρχίσει να περιορίζεται η είσοδος μόνο σε ανθρωπιστικές περιπτώσεις, ανθρωπιστικής βοήθειας, σε όσους δηλαδή χρειάζονται ιατρική βοήθεια. Τα καταλήμματα λοιπόν φιλοξενούν 170.000 άτομα και εικάζεται ότι πάρα πολλά άτομα προσπαθούν να φτάσουν στα σύνορα της Τουρκίας. Τα σύνορα μεταξύ Ιράκ τώρα και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την κουρδική περιοχή της, ε, του Ιράκ και της Συρίας έμειναν σχεδόν ε, τελείως κλειστά τους τελευταίους 7 μήνες με εξαίρεση δύο εβδομάδες ε, το 2013 και το 2014 όπου οι πρόσφυγες ε, μπόρεσαν να μπουν στη χώρα από τη Συρία. Και τώρα κοιτάμε συγκεκριμένες ομάδες που αντιμετωπίζουν ε, έντονους περιορισμούς. Οι άντρες κάθε ηλικία υπόκειται σε εκτενείς ελέγχους στα σύνορα και είναι πιο πιθανή να τους αρνηθούν την είσοδο. Οι Παλαιστίνοι πρόσφυγοι, πρόσφυγες δεν μπορούν να εισέλθουν στις χώρες αυτές ουσιαστικά και η κυβέρνηση του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι οι Παλαιστίνοι πρόσφυγες από τη Ρουσία θα μπορούσαν να πάρουν κάποιες βίζες προέγκρισης από τις ε, μυστικές υπηρεσίες ή χρειαζόταν ε, βίζα κατοικίας. Ακόμα διαμονής, ακόμα πιο δύσκολο δηλαδή να τη λάβουν. Ήταν πάρα πολύ αυστηρή η όρη και έτσι ήταν σχεδόν αδύνατο. Η Ορδανία. Η Ορδανία επίσημα δεν επιτρέπει στους Παλαιστίνιους προσφύγους από τη Συρία να μπει στη χώρα από τον Γενάρη του 2013. Και από διάφορες μελέτες προκύπτει ότι οι Παλαιστίνοι έχουν διωχθεί στη Συρία όταν μπαίνουν από ανεπίσημα σημεία εισόδου. Σε ό,τι αφορά τον επαναπατρισμό τώρα, οι χώρες ε, γειτονικές ε, της Συρίας ε, αναγκάζουν σε πολλές περιπτώσεις τους πολίτες, του Σύρους να φεύγουν και να ξαναπάνε στην Συρία. Από τις 100.000 το UNHCR θέλει να επαναπατρίσει μεγάλο ποσοστό το 2014 αλλά δεν ξέρουν πού ακριβώς θα πάνε αυτά τα άτομα. Η Τουρκία έλαβε πιο πολλούς πρόσφυγες σε τρει μέρε το Σεπτέμβριο από ότι δέχθηκε τα τελευταία τρία χρόνια ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν κάνουν αρκετά για τους ε, Σύριους πρόσφυγες. Γερμανία, Αυστρία και Σουηδία είναι τα φωτεινά παραδείγματα, οι φωτεινέ εξαιρέσει. όπου ανακοινώθηκε ότι θα δοθεί μόνιμη διαμονή σε όσους ήρους το επιθυμούν. Το Ηνωμένο Βασίλειο ε, έκανε επαναπατρισμό 500 σύρων στην ε, τελευταία περίοδο. Θα πρέπει να λοιπόν να υπάρξει μια χρηματοδοτημένη ανταπόκριση ανθρωπιστικής εκτακτού ανάγκης. Και θα πρέπει να βρεθεί τρόπος εγκατάστασης των προσφύγων κάπου αλλού. Να επιτυχθεί πραγματική αλληλεγγύη με τις χώρες που είναι γειτονικές της Συρίας. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε. Κατά το ελάχιστο θα πρέπει να συνεχίσουμε την υφιστάμενη ανθρωπιστική βοήθεια και αναπτυξιακή βοήθεια στις χώρες που συνορεύουν με τη Συρία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό νομίζω να βρούμε έναν τρόπο να συνδυάσουμε τις αναπτυξιακούς πόρους και τους ανθρωπιστικούς πόρους για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις των χωρών υποδοχής σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα των κοινοτήτων τους. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη διαβούλευση των, της κοινωνίας των πολιτών να βρει μια συνολική, συνεκτική στρατηγική για να ανταποκριθεί στην κρίση στη Συρία, όπως ζητήθηκε από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην τελευταία σύνοδο του Υπουργείου εξωτερικών υποθέσεων και θα πρέπει αυτό να εμπλέξει όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα της Ένωσης. Θα πρέπει να καλέσουμε τους παγκόσμιους οργανισμούς και τις πλούσιες χώρες να κάνουν πιο πολλά. Οι επενδύσεις θα πρέπει να στοχεύσουν στη βελτίωση της υποδομής, στις ε, εγκαταστάσεις εκπαίδευσης και υγειονομικής περίθαλψης, προκειμένου να βελτιώσουμε την κατάσταση για τους πρόσφυγες να υπάρχουν προγράμματα για καταλήμματα. Να υπάρχει αυτάρκεια στις κοινωνίες υποδοχής. Να δοθούν κίνητρα προκειμένου να συνεχίσουν να υποδέχονται πρόσφυγες. Και τέλος, να υπάρχει υποστήριξη από την διεθνή κοινότητα, η οποία θα περιλαμβάνει και οικονομική αρρωγή. Για να μπορέσει να υπάρχουν δυνατότητε και για τον πληθυσμό στη χώρα υποδοχής, αλλά και για τους πρόσφυγες σε ό,τι αφορά την επανεγκατάσταση των, την επανένωση οικογενειών θα πρέπει να λεφθούν ειδικέ πρωτοβουλίε, ιδιαίτερω από πλευρά των αναπτυγμένων χωρών, των πλούσιων χωρών. Ιδιαίτερα όσες έχουν προσυπογράψει τη συνθήκη του 51 για του πρόσφυγες. Προκειμένου να υπάρξει επανεκατάσταση μεγάλου ποσοστού των σύρων προσφύγων θα πρέπει η υποστήριξη στου Σύρους πρόσφυγες να είναι σαφέ ότι δεν είναι ει βάρο της αρρωγής προσφύγων αλλού. Θα πρέπει επίση η επανεγκατάσταση να βασίζεται σε κριτήρια ευαλωτότητας και να, αυτό να είναι σε, σε να υπακούει στους κανόνες που έχουν οριστεί στη συνθήκη του 51. Σε ό,τι αφορά τώρα τον έλεγχο των συνόρων θα πρέπει να γίνεται χωρίς να καταπατούν τα δικαιώματα των προσφύγων. Είναι τεράστιο το κόστος ε, της υποδοχής των προσφύγων. Θα πρέπει λοιπόν να κατανεμηθεί δίκαια και όλοι όμως, ε, όλες οι κυβερνήσεις θα πρέπει να πληρούν και να σεβαστούν τις σχετικές αρχές. Η Πρόεδρος Διακόπτη, δεν ξέρω πόσο θέλετε να σκοπεύετε να μιλήσετε ακόμα, αλλά μπορούμε να διαβάζουμε και τα PowerPoint. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα γίνονται σεβαστά τα ψηφίσματα 2139 και 2165 και σε ό,τι αφορά πρέπει να διασφαλίσουμε λοιπόν ότι αυτά τα μέτρα θα συνδυάζονται όλα μαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρο, Να περάσουμε στον επόμενο ομιλητή. ο οποίος είναι ο κύριος Ζήλ Ανσούλ και είναι ανώτερος σύμβουλος για θέματα επιχειρησιακών υποθέσεων του Ερυθρού Σταυρού. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να κάνω μια μικρή διόρθωση για το πώ παρουσιάστηκε η διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού επικεφαλής τη αντιπροσωπεία μου δεν θα χαιρόταν, δεν ε, είναι ε, η κυβερνητική οργάνωση ο Ερυθρός ε, αλλά μια διεθνή οργάνωση, όπως γνωρίζετε, ένας διεθνή οργανισμός. Δεν θα επανέλθω στα αριθμητικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν από τον κύριο Σόρενσεν αυξάνονται συνεχώς τα νούμερα. Επομένως, θα περάσω σε αυτά που αφορούν τη Διεθνή Επιτροπή του Ερθρού Θα ήθελα να κατανοήσετε πώς είναι για τους συναδέλφους μου εκεί να εργάζονται σήμερα και να συμμετέχουν σε κάποια ανθρωπιστική επιχείρηση. Καταρχήν η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού από την έναρξη της κρίσης έχει επιλέξει να οικοδομήσει μια ανθρωπιστική δράση από το εσωτερικό της χώρας δηλαδή. Δεν ε, κατέφυγε σε διασυνοριακές επιχειρήσεις ε, που ε, δεν επιτρέπεται από την κυβέρνηση της Συρίας και αυτό σύμφωνα με το συνήθι τρόπο δράσης, του operandi, της Διεθνούς Επιτροπής, δηλαδή να κάνουμε διάλογο με όλα τα μέρη της σύραξης και να υπάρχει συμφωνία για τις επιχειρήσεις μας. Αυτό, όπως μπορείτε να φανταστείτε οι περισσότεροι, σήμαινε ότι έπρεπε να κάνουμε μήνες υπομονή και να είμαστε αποφασισμένοι για να προσπαθήσουμε να αποδείξουμε το πόσο σχετική είναι η δουλειά της Διεθνούς Επιτροπής του Ερθρού Σταυρού, δηλαδή ουδέτερη, αμερόληπτη και ανεξάρτητη δράση στη Συρία. Μπορώ να πω όμως ότι η Διεθνής Επιτροπή έχει φτάσει τώρα σε μια επιχειρησιακή ικανότητα να απαντήσει σε ορισμένες από τις πιο επίγουσες ανάγκες. Πράγματι, στην ε, Δαμασκό, πέρα από τα γραφεία και τις αποθήκες ε, και στο Τατού, στην Ακτή. Η Διεθνής Επιτροπή του Σταυρού έχει τώρα μόνιμη παρουσία στη Χόμς, καθώς και στο Χαλέπι. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε πως φαίνεται να μην υπάρχει ακόμη προθυμία να δοθεί στη Διεθνή Επιτροπή του Ρυθού Σταυρού μια γενική και επανειλημμένη πρόσβαση σε όλα τα θύματα που χρήζουν προστασίας και βοήθεια στη Συρία. Παρ' όλα αυτά, η Διεθνής Επιτροπή τους τελευταίους δύο μήνες έχει λάβει αυξημένες θετικές απαντήσεις ε, στα επανειλημμένα αιτήματά της ε, να προσφέρει βοήθεια στους πληθυσμούς που βρίσκονται σε κίνδυνο και έχουν ανάγκες ε, και στις δύο γραμμές του μετόπου. Από το καλοκαίρι η Διεθνής Επιτροπή έχει πολλαπλασιάσει σε στενή συνεργασία με την Ερυθρέα Μισέλινο κάποιες Διασυνορικές επιχειρήσει, με τοπικές μάλλον επιχειρήσεις ε, στο Χαλέπι και προσφέρει βοήθεια στα δυτικά του Χαλεπίου που ελέγχονται από κάποιες ομάδες της αντίστασης. Η ανατολική πλευρά του ε, Χαλεπίου ελέγχεται από το Ισλαμικό κράτος και το νότιο τμήμα ελέγχεται από την κυβέρνηση. Και αυτό συμπεριλαμβάνει και χειρουργική βοήθεια όπως καταλαβαίνετε δεν πρόκειται για κάτι εύκολο, δεν μας επιτρέπουν, πολύ εύκολο, να λάβουμε το πράσινο φως. Για 10 ημέρες στην ανατολική περιοχή του Χαλεπίου, η RCC, η Διεθνής Επιτροπή, προσέφερε τρόφιμα σε 95.000 ανθρώπους που ζουν στην περιοχή αυτή που πλήττεται από τη σύραξη. Ένα δεύτερο παράδειγμα είναι τις τελευταίες εβδομάδες η στη Διεθνή Επιτροπή δόθηκε πρόσβαση σε κάποιες πολιορκημένες περιοχές όπου έχουν παγιδευτεί άμαχοι για μήνες, μερικές φορές και για έτη. το χάρη στη Μαχαδεμία και στο Γιάμουκ λάβαμε πρόσβαση για πρώτη φορά εδώ και ένα χρόνο, καθώς και στη γειτονιά Λουέρ στη Χόμς, όπου μπορέσαμε να προσφέρουμε ιατρική βοήθεια για κάποιες χιλιάδες ανθρώπους. Επομένως, η Διεθνή Επιτροπή του Ρήθου Σταυρού μπόρεσε φέτος να αυξήσει την ανθρωπιστική της απάντηση και αυτή τη στιγμή έχει τη μεγαλύτερη επιχειρήση με 300 άτομα του προσωπικού επιτόπου, μοιράζει τρόφιμα κάθε μήνα περίπου σε 50 σε 500.000 μας ανθρώπους και διασφαλίζει την πρόσβαση σε πόσιμο νερό για το 80% του πληθυσμού που ξεκολουθεί να ζει στη Συρία. Αυτή η αρρωγή από μόνη της είναι αξιοσημείωτη θα έλεγα όμως, αν ε, λάβουμε υπόψη τα αριθμητικά στοιχεία που ακούσαμε στην αρχή, κατανοούμε ότι είναι πολύ ελλειπής η κατάσταση, δεν είναι καθόλου ικανοποιητική και σχεδιάζουμε αύξηση του προπολογισμού για του χρόνου άνω του 35%. Έτσι λοιπόν πέρα από αυτές τις λίγες θετικές εξελίξεις ό,τι αφορά την πρόσβασή μας η παρουσία της Διεθνούς Επιτροπής επιτόπου αντιμετωπίζει πάρα πολλές δυσκολίες ε, λόγω της κατάστασης. Καταλαβαίνετε ότι είναι ιδιαίτερα σταθής και λόγω του αριθμού των ενόπλων ομάδων έχουμε, δω, έχουμε δεκάδες τέτοιες ενόπλες ομάδες που ε, υπάρχουν εκεί και υπάρχει και εχθρότητα που εκφράζεται απέναντι στις ομάδες ανθρωπιστικής βοήθειας, κυρίως στην Ανατολή και στον Νότο και φυσικά ε, έχουμε και τρεις συναδέλφους που έχουν απαχθεί τον Οκτώβριο του 2013. Έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος και δυστυχώς ακόμη αγνοούνται. Ίσως ε, θα είδατε τη συνέντευξη ε, του Πρόεδρου Πετωμαΐν στη Λεμόντ την περασμένη εβδομάδα υπενθύμησε ότι ο Ερυθρός ε, Σταυρός προσπαθεί να διασφαλίσει πρόσβαση στους ευάλωτους πληθυσμούς σε όλες τις πλευρές της Συρίας και στις περιοχές που ελέγχονται από το Ισλαμικό κράτος. Και εδώ θα περιμένω κάποιες ερωτήσεις που μάλλον έχετε. Με αυτούς ε, η ελεπίδραση μπορεί να λάβει χώρα στην περιφέρεια των επικρατιών που ελέγχουν. Ε, συχνά υπάρχουν και κάποιοι μεσάζοντες όμως θέλουμε να φέρουμε βοήθεια, ιατρική βοήθεια, τρόφιμα, νερό σε αυτές τις επικράτειες για τους αμάχους. Στη Χάκα, παραδείγματος χάρη πρόσφατα, καθώς και στο Ανατολικό Χαλέπι, στο Ιράκ, στο Φαλούτζια και στη Μοσούλη. Στη Φαλούτζια και στη Μοσούλη. Θα ήθελα λοιπόν να επαναλαβώ και εγώ αυτά που λένε οι συνάδελφοι τα τελευταία τέσσερα χρόνια, να απευθύνω έκκληση σε όλα τα μέρη της σύραξης να σεβαστούν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, να μη στοχεύουν στους αμάχους και να επιτρέψουν να υπάρχει αμερόληπτη και ανεξάρτητη ανθρωπιστική βοήθεια. Σα ευχαριστώ για την επισκόπηση αυτή. μα παρουσιάσατε πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση. Ευχαριστώ και τον κύριο Σόρσεν. μα είπε πω η Κομισιόν προσπαθεί να βοηθήσει σε πάρα πολύ δύσκολε συνθήκε. Συνάδελφοι, έχω δύο άτομα που ζητούν το λόγο. Καταρχήν, ε, κύριο Σαλόμ, που είναι ο μόνιμος εισηγητής της Επιτροπής μας για την ανθρωπιστικά θέματα και κατόπιν κύριο Στήρ. Ναι, ευχαριστώ πολύ τους κυρίους ε, Σόρετς, Μιχανσούλ και Χάτσεν όχι μόνο για την ενημέρωση και τις πληροφορίες που μας έδωσαν, αλλά και για τα όσα κάνουν κάθε μέρα προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτή την ανθρωπιστική κρίση, η οποία πλέον διαρκεί πάνω από τρία χρόνια και στη διάρκεια αυτών των τριών ετών έχει αρχίσει να αλλάζει το πολιτικό στρατηγικό στρατηγικό και στρατιωτικό προφίλ της σύραξης. Έχουμε δει αυτές τις αλλαγές, αλλά παρόλα αυτά η ανθρωπιστική κρίση ε, ακολουθεί την ίδια πορεία και επιδεινώνεται συνεχώς. Από τις τέσσερις ανθρωπιστικές κρίσεις ε, ε, υψής του επίπεδου που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, οι δύο είναι στην περιοχή. Η Συρία και το Ιράκ. Οι άλλες δύο είναι το Νότιο Σουδάν και η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Η κρίση αυτή Δεν θα ήθελα να επαναλάβω τα στατιστικά στοιχεία, αλλά θα ήθελα να επισημάνω κάτι το οποίο κατά την άποψή μου αξίζει τον κόπο να αντιμετωπίσουμε από αυτό το πρίσμα. Μία χώρα σαν το Λίβανο συγκεντρώνει ένα αριθμό προσφύγων ισοδύναμο με το να, λάβει, να υποδεχτεί η Γερμανία 16 εκατομμύρια πρόσφυγες ε, στη χώρα της. Σαν να δεχόταν 8 εκατομμύρια πρόσφυγες η Ισπανία στη χώρα της. Μία χώρα ε, σαν την Ιορδανία που είναι μια χώρα που ούτως ή άλλως αυτές διαθέτει πολλαπλά προβλήματα, ο αριθμός των προσφύγων είναι σαν να είχε η Γερμανία 6 εκατομμύρια πρόσφυγες και η Ισπανία 3,5 εκατομμύρια πρόσφυγα. Δηλαδή θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πόσο μεγάλη είναι η θυσία που κάνουν αυτές οι χώρες και θα πρέπει να δείξουμε την ευγνωμοσύνη μας εμείς από αυτή την πλευρά του κόσμου όπου είμαστε πολύ περισσότεροι εγωιστές και πολύ πιο ε, προστατευτικοί ως προς την ευημερία και τη σταθερότητά μας. Πέραν αυτού όμως θα ήθελα να επισημάνω διότι ε, κάποια στιγμή στις παρεμβάσεις επισημάνθηκε η ανθρωπιστική πτυχή. Όντω, εμεί συζητάμε το θέμα από ανθρωπιστική πλευρά, αλλά μια συζήτηση ανθρωπιστική μεν που χρειάζεται και ένα πολιτικό προσανατολισμό. Διότι πολλά από τα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να επιλύσουμε προκειμένου να ε, βοηθήσουμε από ανθρωπιστική σκοπιά στου εκτοπισμένου, στου ανθρώπου που ζουν στη Συρία, χρειάζεται πολιτική δράση. Και χρειάζεται πολιτική δράση αφενό για την πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια. Διότι γνωρίζουμε ότι τόσο εντό τη Συρία, όπου η κυβέρνηση δυσχεραίνει την πρόσβαση σε αυτή την ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά ταυτόχρονα και αυτοί οι οποίοι ε, πολεμούν την ε, ε, κυβέρνηση της Συρίας και αυτοί τη δυσχεραίνουν. Ε, επομένως υπάρχει ένα πολλαπρό πρόβλημα πρόσβασης ανθρωπιστικής βοήθειας και ε, αντιλαμβανόμαστε όπως θα μπορέσουμε ίσως να καταλάβουμε και ότι οι όμορες χώρες που υποδέχονται αυτές τις ε, τόσο μεγάλες, τόσο μεγάλους αριθμούς προσφύγων θα αρχίσουν να δημιουργούν προβλήματα στα σύνορα, θα έχουν φραγμούς ώστε να μην ξεφύγει από τα χέρια τους η κατάσταση ε, στην οποία βρίσκονται. Θεωρώ λοιπόν ότι ένα από τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε εμεί σε αυτή την Επιτροπή και να φτάσει και προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μέσω τη Γενική Διεύθυνση τη ΕΚΟ, αλλά να φτάσει και στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ή δυνατόν να φτάσει και στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, θα πρέπει λοιπόν να γίνει πολιτική δουλειά ώστε να υπάρχουν ανθρωπιστικές παύσεις, ανθρωπιστική διάδρομη, μέτρα τα οποία θα επιτρέψουν σε όσοι ε, με προσωπικές, σε όσους με προσωπικές ε, θυσίες βοηθούς τους εκτοπισμένους που ζουν αυτή τη βία εντός της Συρίας να έχουν πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια. Επίσης χρειαζόμαστε πολιτική δράση προκειμένου να γίνεται σεβαστή η διεθνής ανθρωπιστική νομοθεσία. Αυτή τη στιγμή υπάρχει βία, όπως είπαν αρκετοί, η οποία ε, είναι κατά του άμαχου πληθυσμού. Ε, σε σχολεία, σε νοσοκομεία, σε αγορές, ε, δηλαδή σε χώρους και επιπλέον εδώ και είναι καταδικασμένοι σε πείνα πληθυσμοί οι οποίοι βρίσκονται κοντά στα σύνορα ε, και σε περιοχές οι οποίες είναι κατεχόμενες από τις αντιμαχόμενες πρευλέ στη σύραξη. Επομένως θα πρέπει να υπάρξει πολιτική ε, δράση ώστε να μην χρησιμοποιείται ο άμαχος πληθυσμός ως ε, όπλα κατά του πολέμου, να μην υπάρχει βία κατά των παιδιών, βία κατά των γυναικών και να μην προκαλείται η πείνα και η ένδυα. Εγώ είμαι βέβαιος ότι η Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ συμμερίζεται ή τουλάχιστον συμμεριζόμαστε εμεί μαζί τους αυτή την ανάγκη για πολιτική δράση και θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια για το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, πώς θεωρείτε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε εμείς από πλευράς μας, ε, από πλευράς Επιτροπικής Ανάπτυξης. Δύο ακόμα σημεία και μετά ε, ολοκληρώνω πολύ σύντομα. Είναι σκανδαλώδης η αντίδραση των χωρών τη ευρωπαϊκή ένωση ως προς το πρόβλημα για το θέμα της υποδοχής των προσφύγων. Η Oxfam προτείνει για το 2015 σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση να υποδεχθούμε 180.000 πρόσφυγες. Και θα πρέπει να σας πω ότι ο συνολικός αριθμός των προσφύγων αυτή τη στιγμή είναι περίπου 4 εκατομμύρια στις όμορες χώρες. Επομένως, εμείς θέτουμε ε, ως ε, στόχο τις 180.000. Και όπως ακούστηκε, υπάρχουν, όπως σας είπα μάλλον, υπάρχουν και κάποιες χώρες οι οποίες ε, τηρούν τα όρια, η Γερμανία, η Αυστρία, μπορεί και η Νορβηγία που δεν είναι μελών της Ένωσης ΜΕΝ, αλλά αποτελεί παράδειγμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν κάνουν βέβαια το ίδιο και οι περισσότερες χώρες. Είναι γελίο αυτό το ποσό ε, υπάρχει κάποια χώρα, δεν θα την αναφέρω, που έχει 50 πρόσφυγες υποδεχθεί. Ε, αυτό είναι ξεκάθαρα εγωισμός και τίποτα άλλο. Ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, διότι εγώ ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαμαρτύρεται για τον προϋπολογισμό, αλλά ο προϋπολογισμός του 2014 είναι μικρότερος από το 2013 και νομίζω την περασμένη Παρασκευή στην έκθεση στο Συμβούλιο Ασφαλείας ε, από πλευράς Ηνωμένων Εθνών επισημάνθηκε ότι οι δεσμεύσεις που αναλήφθησαν από τους διάφορους δωρητές αυτή τη στιγμή με το ζόρι φτάνουν στο 40% των αναγκών. Και με αυτό θέλω να τονίσω και θα ήθελα να ρωτήσω ε, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν δύο εβδομάδες στην συνεδρίαση στη Γερμανία ε, γιατί δεσμεύτηκε και τι θα πρέπει να κάνουμε ώστε ο καθένας στη χώρα του από εκεί και πέρα να πιέσουμε όχι μόνο για να δοθούν κονδύλια αλλά γιατί όπως είπε και ο κύριος ε, ε, Σόρενσε να έχουμε και ταχύτατα χρήματα γιατί χρειαζόμαστε χρήματα για ανταπόκριση στην κρίση και όχι ενδιάμεση γραφειοκρατία που ο μόνον ε, οδηγεί σε απώλεια των χρημάτων διότι καθυστερούν πάρα πολύ αλλά και σε πολλές περιπτώσεις ε, το να έρθουν τα πράγματα, τα χρήματα κατόπιν εορτής είναι το ίδιο με το να μην δοθούν καθόλου. Και όταν χάνουμε ανθρώπινες ζωής ε, ε, είναι το ίδιο με το να χάνουν οι άνθρωποι τη δυνατότητα επιβίωσής τους. Ο κύριος Στήρ και μετά η κυρία Χάουταλα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ και εσάς τρεις ομιλητές για τις παρουσιάσεις σας. Τρεις σύντομες παρατηρήσεις από δική μου πλευρά. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά το θέμα που αναφέρθηκε για την ικανότητα απορρόφησης και σε ό,τι αφορά το θέμα της ανθρωπιστικής κρίσης. Δεν μπορούμε να μιλάμε όμως για θέματα ανθρωπιστικής κρίσης χωρίς να μιλάμε για την πολιτική λύση. Υπάρχει λοιπόν αυτή η ανάγκη πολιτικής επίλυσης του θέματος. Και νομίζω ότι ανεξάρτητα από τις διαφορές των απόψεων των πολιτικών συνιστώσεων, για το ποια θα έπρεπε να είναι η σωστή πολιτική λύση που θα έπρεπε να έχει εφαρμοστεί, όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι η πολιτική μας που έχει αλλάξει διαρκώς μάλλον στη διάρκεια της κρίσης ουσιαστικά επιδίνωσε την κρίση. Δεύτερο θέμα, δεύτερο, δεύτερη σκέψη σε ό,τι αφορά τις όμορες χώρες. Πολλά στοιχεία μας δώσατε. από δικής μου πλευράς, με την εμπειρία της δικής μου χώρας που αντιμετώπισε την πρόκληση ε, εκατομμύρια προσφύγους με σύνολο 4,4 εκατομμύρια πληθυσμού στην επικράτειά μας. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ποιες είναι οι προκλήσεις. Να εκφράσουμε ευγνωμοσύνη λοιπόν στις όμορες χώρες που υποδέχονται τις πρόσφυγες. Η ερώτηση έρχεται μετά από την συζήτηση που είχαμε στην Ολομέλεια για το κομπάνι, όπου πολλοί ομιλητέ αναφέρθηκαν στο θέμα της σχέσης με την Τουρκία. Φυσικά αυτό αναφέρθηκε από πολιτική σκοπιά. σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση της Τουρκίας για την στρατιωτική στρατηγική, σε ό,τι αφορά την πράσπιση των πολιτών στο κομπάνι. Αλλά αυτό, όπως αναφέρθηκε, έχει και μια ανθρωπιστική πτυχή. Σήμερα λοιπόν βλέπουμε ότι η νέα επιτροπή και η νέα, ο νέος επίτροπος ε, πλέον δραστηριοποιούνται. Και ποια λοιπόν είναι τα βήματα σε ό,τι αφορά τη σχέση με την Τουρκία. Και νομίζω ότι ο διάλογος θα πρέπει να εμπεριέχει όλες αυτές τις ανησυχίες. Το τρίτο θέμα είναι φυσικά το θέμα της χρηματοδότησης, του προπολογισμού. καθήκον μας είναι λοιπόν ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν όλοι μιλούν και στο ιστορικό των πολιτικών ομάδων το συζητάμε το θέμα αυτό, το κάναμε και στη δική μας ομάδα, εκφράζεται η ανησυχία ότι αν το θέμα αυτό δεν επιληθεί, αν υπάρχουν πόροι από την προηγούμενη χρηματοοικονομική περίοδο, για πόσο χρονικό διάστημα θα μπορεί να συνεχίσει τις προσπάθειές της η Γενική Διεύθυνση ΕΚΟΝ, για παράδειγμα. Μία εκτίμηση ενός συναδέλφου από την Επιτροπή Προϋπολογισμών ήταν ότι θα μπορούσε να συνεχίσει για, τρία, για τρεις μήνες μόνο τη δράση της. Ίσως να είναι απεσιόδοξη αυτή η εκτίμηση, αλλά θα με ενδιαφέρει να ακούσω και τη δική σας γνώμη. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. και μετά, η κυρία Θεοχάρους. Ε, ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σύμφωνο ότι το πρόβλημα των πληρωμών είναι πραγματικά παράδεκτο, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ανθρωπιστική βοήθεια και ελπίζω τα θεσμικά όργανα μπορούν να βρουν μία λύση, γιατί είναι πραγματικά ντροπή το πόσο λίγους πρόσφυγες έχουν υποδεχθεί ε, τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα ε, καλό παράδειγμα είναι η Σουηδία. Η Σουηδία δήλωσε ότι όλοι οι πρόσφυγες από τη Συρία θα λάβουν ε, βίζα διαμονής. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό το παράδειγμα αυτό. Επισκύφθηκα την Ιορδανία κοντά στα σύνορα με τη Συρία πέρσι τον Ιούνιο και διαπίστωσα με μεγάλο ενδιαφέρον τότε ότι ο επικεφαλής του καταλήμματος είχε δώσει διάφορες συνεντεύξεις στον δημόσιο τύπο και θεωρείται αυτό του σαν ένα δήμαρχο ουσιαστικά μιας κομμόπολης. Γιατί η κατάσταση είναι σαφή, θα μείνουν τα άτομα αυτά για κάποιο διάστημα, ίσως και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, στους χώρους αυτούς και χρειάζονται λοιπόν κάποιες υποδομές σε ό,τι αφορά την οργάνωσή τους. Είναι πολύ μικρό όμως το τμήμα των σύρων προσφύγων που τελικά φιλοξενείται στα καταλήμματα αυτά. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει κάποια βασικά, κάποιες βασικές προϋποθέσεις να παρέχουμε στους ανθρώπους αυτούς προκειμένου να μην αναγκαστούν να μένουν σε πρωτόγονες συνθήκες. Ξέρω ότι το Νορβηγικό Συμβούλιο κάνει πολλά σε ό,τι αφορά τα καταλήμματα προσφύγων. Πώς μπορούμε λοιπόν να βελτιώσουμε την κατάσταση για να βοηθήσουμε πιο πολλούς ανθρώπους και πιο καλά, πιο αποτελεσματικά. Ευχαριστώ κυρία Θεοχάρους. Και μετά Νόρμπετ Νόιζερ. Και μετά θα κλείσω το κατάλογο ομιλητών. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να επισημάνω ότι κάθε φορά που συζητάμε ένα πρόβλημα, λες και εκείνη την ώρα έχει δημιουργηθεί το πρόβλημα. Δες, λες και δεν υπάρχει μια προϊστορία πάνω στην οποία έχουμε συζητήσει πολλές φορές στο παρελθόν και έχουμε προσπαθήσει να αναλύσουμε την πολιτική σημασία του κάθε όρου. Δεν μπορώ να μιλήσω με οικονομικούς όρους, όμως με πολιτικούς ορούς θα σας πω τα εξής. Ε, έλαβα μέρος σε μια ανθρωπιστική αποστολή στη Χόμς πριν από δύο χρόνια ως γιατρός τον Νοέμβριο του 2012 και είχα αποστείλει επιστρέφοντας μια επιστολή προς όλους τους συναδέλφους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιγράφοντας αυτά τα οποία είχα βιώσει την αγριότητα εκείνη του πολέμου και το γεγονός ότι αυτοί που διεκδικούσαν να ανατρέψουν τον Άσαντ δεν ήσαν καλύτεροι από τον Άσαντ. Μπορεί να ήταν και χειρότεροι. Είχα επισημάνει αυτό που είπε ο κύριος Χανσούλ και συμφωνώ απόλυτα μαζί του ότι το πιο σωστό ήταν να δημιουργήσουμε κάποιους ανθρωπιστικούς διαδρόμους μέσα στη Συρία, κάποιες ζώνες προστασίας των ανθρώπων εκεί πέρα γιατί αυτή η φυγή πού θα οδηγήσει, πού θα πάνε όλοι αυτοί. Δηλαδή αν ανοίξουμε τα σύνορα είναι σίγουρο ότι όλος ο, ο πληθυσμός της Συρίας θα φύγει από εκεί. Δεν πρόκειται να μείνει εκτός από αυτούς που σκοτώνει ο ένας τον, ε, ο ένας τον άλλο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλοί ευρωπαϊκοί πληθυσμοί, ειδικά οι πληθυσμοί του Νότου, δεινοπαθούν ήδη οικονομικά. Περνούν μια άγρια οικονομική κρίση που δεν επιτρέπει κάποιο να σκέφτεται ότι θα βγάλει από το ιστέρημα του να βοηθήσει εφόσον οι ανάγκε είναι τόσο τρομακτικέ. Για παράδειγμα, στη δική μου τη χώρα έχουμε ιατρία για του φτωχού, τα έχουμε δημιουργήσει και τα έχουμε διασπείρει όλη τη χώρα. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να νιώσει όσο μεγαλοψυχία και να έχει ένας ότι θα βγάλει και να βοηθήσει για τους Σύρους τους πρόσφυγες. Επίσης οι Σύροι πρόσφυγες όταν επιχειρούν να διαφύγουν για παράδειγμα με πλεούμενα όπως αυτό που βυθίστηκε πρόσφατα ανοιχτά της Κύπρου και διασώθηκαν περίπου 300-400 τόσοι άνθρωποι στόχος τους δεν είναι ούτε η Κύπρος, ούτε η Ελλάδα, ούτε η Μάλτα. Στόχος τους είναι να φτάσουν στην Ιταλία και από εκεί να διοχετευτούν στις πλούσιες χώρες της Ευρώπης. Άρα και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας όταν κάνουμε αυτή την κριτική ότι θέλουν η Σουηδία ε, και η Γερμανία υποδέχονται περισσότερους πρόσφυγες. Μα θέλουν οι πρόσφυγες να πάνε σε αυτές τις χώρες. Δεν επιδιώκουν να φτάσουν σε φτωχές χώρες όπως είναι η Κύπρος όπου και της Κύπρου ο πληθυσμός της κατά 40% είναι προσφυγοποιημένος εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ζει σε πολύ πρωτόγονες συνθήκες. Όσον αφορά την ευθύνη και τα συμφέροντα αναφέρθηκαν από τον κύριο Σόρενσεν, τα συμφέροντα των μεγάλων χωρών. Ε, στις μεγάλες χώρες εγώ θα βάλω και την Τουρκία η οποία για χρόνια εξολόθρευε τον κουρδικό πληθυσμό και έσβηνε κουρδικά χωριά από τον χάρτη και τους έστελνε στο Καμισλή και στη Βόρεια Συρία και στο Ιράκ και συνεπώς είναι λογικό αυτή τη στιγμή κάποιοι άνθρωποι να θέλουν να είναι να θέλουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Άρα θα πρέπει να δούμε και αυτή τη ε, ε, διάσταση καθώς και το γεγονός ότι η Τουρκία ευθύνεται σαφέστατα για την ε, έκταση που πήρε η σύγκρουση μέσα στη Συρία και για τις σχέσεις της που έχει με, με το Ισλαμικό κράτος να θυμίσω ότι στην αρχή της προηγούμενης περίοδου είχα εισηγηθεί στην κυρία Γεωργίευα την ανάγκη δημιουργίας ενός humanitarian task force το οποίο να μπορεί να κινείται εύκολα, άνετα, αποτελεσματικά και δυναμικά προς τους χώρους που χρειάζονται ανθρωπιστική παρέμβαση. Δυστυχώς η πρότασή μου παρόλο που ήταν τεκμηριωμένη δεν εισακούστηκε και δημιουργήθηκε ένα σώμα εθελοντών το οποίο δεν έχω δει να λειτουργεί. Δεν ξέρω, συγχωρέστε μου την άγνοια, αλλά νομίζω ότι δεν έχει λειτουργήσει ακόμη αυτό το σώμα των εθελοντών. Έχω μια ερώτηση μόνο αν το Ισραήλ έχει υποδιεχθεί οποιουσδήποτε πρόσφυγες και αν όχι πώς μπορεί να ερμηνευτεί αυτό γιατί είναι και αυτό μια όμορη χώρα και ε, θα ανέμενε κάποιος ότι κάποιοι θα επιχειρούσαν να πάνε και προς το Ισραήλ. Σας ευχαριστώ πολύ. And ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχάς, εν συντομία, να παρουσιάσω πώς εμείς ως Ευρωπαϊκή Κοινότητα στην περίπτωση αυτή συμπεριφερθήκαμε τώρα. Δύο λέξεις νομίζω μπορούμε να, να χρησιμοποιήσω. Ντροπή και φτωχά. Και νομίζω ότι ο Ενρίκε, ο συζητητής για την ανθρωπιστική βοήθεια, ε, επεσήμανε τα ελλείμματα. Γνωρίζουμε και την κατάσταση εδώ στην Επιτροπή εδώ και καιρό. Σε όλες τις ανθρωπιστικές καταστροφές, η Επίτροπος Τζοτζίεβα μας λέει ότι δεν είχαμε πολλά χρήματα για να αντιμετωπίσουμε την ε, ανθρωπιστική κρίση και τα κράτη-μέλη δεν έμαθαν τίποτα. Ακόμα πιο λίγα χρήματα έχουμε φέτος στη διάθεσή μας από την Πέρση και αυτό θα συνεχίσει στο μέλλον. Νομίζω λοιπόν θα πρέπει να συνεχίσουμε την πίεση στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να δίνει τα χρήματα για την ανθρωπιστική βοήθεια η Ευρωπαϊκή Ένωση που χρειάζονται. Κατά δεύτερον, οι πολιτικές ε, λύσεις, οι προτάσεις λύσεων αναφέρθηκαν. Νομίζω ότι ο ΙΕ θα πρέπει να σπρώξει πολύ πιο πολύ και η Ρωσία και η ΙΠΑ θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν όσο δύσκολε και είναι οι σχέσεις ε, ε, των δύο χωρών λόγω της Ουκρανίας. Και θα καλέσω την κυρία Μορκαρίνη να δραματίσει σημαντικό ρόλο. Επίσης, οι δύο άλλοι μεγάλοι ε, γείτονε, το Ιράν και η Τουρκία, θα πρέπει και αυτούς να τους παρακινήσουμε γιατί μπορούν να βοηθήσουν να σταθεροποιηθεί κατά κάποιο τρόπο η περιοχή. Και χαίρομαι που το συνέδριο του Βερολίνου την προηγούμενη εβδομάδα κατέστησε σαφές ότι η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να δράσει πιο έντονα σε ό,τι αφορά τις τρεις χώρες υποδοχής, η Λίβανος, η Ορδανία και η Τουρκία, προκειμένου λοιπόν να δοθεί βοήθεια στις τρεις χώρες αυτές, προκειμένου και κυρίως ό,τι αφορά τον Λίβανο και την ε, Ιορδανία, να τους ε, χορηγήσουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε την σταθερότητα των χωρών αυτών. Τελευταία ερώτηση και ευχαριστώ τους συζητητές για την παρουσίασή τους, αλλά είπατε και μιλήσατε για την προσέγγιση της ε, Συρίας σε όλες τις διάφορες πολιτικές ομάδες και είπατε ότι υπάρχει πρόσβαση και ότι προσπαθούμε μέσω διαπραγματεύσεων να διασφαλίσουμε και την πρόσβαση σε κοινότητε προσφύγων που ω τώρα δεν λάμβαναν ανθρωπιστική βοήθεια. Να ρωτήσω, οι πολιτικές ομάδες εντό τη Συρίας διαφοροποιούνται ιδιαίτερω και τι γίνεται με την αντιμετώπιση του ίσης. Νομίζω ότι θα είναι χρήσιμο να γνωρίσουμε πώς οι διάφορες πολιτικές ομάδες στη Συρία αντιμετωπίζουν την ανθρωπιστική βοήθεια. Okay, thank you. I'm Ευχαριστώ. Θα ξαναδώσω το λόγο στους προσκεκλημένους μας. Απλώς ε, έχω μια ερώτηση και εγώ. Ακούσαμε ότι η Κομισιόν ε, ένα trust fund κατά τη πραγματικό ταμείο για τη Συρία. Σωστό είναι αυτό. Ε, και γιατί, ποια θα είναι η διαφοροποίηση και θα, ποιος θα είναι ο έλεγχος του Κοινοβουλίου σε αυτό το Trust Fund. Επειδή αργήσαμε να αρχίσουμε, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να είστε σύντομοι, τρία-τέσσερα λεπτά και κατόπιν θα ακολουθήσουν και συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ Λίντα. Ευχαριστώ και για τις ερωτήσεις για το Trust Fund. Και εγώ το έχω ακούσει, το συζήτησα με τους συναδέλφους από την ΤΕΦΚΟ και θα ήθελα να συζητήσουν ε, κάποια θέματα μαζί σας. Νομίζω λοιπόν ότι θα συμβουλευτούν πλήρως, συνεχίζονται οι συζητήσεις ε, μεταξύ των οργάνων ε, και νομίζω ότι η ΔΕΦΚΟ θέλει να υπάρχει μια ταχεία κατανομή των χρημάτων, δηλαδή να έχουν ένα μηχανισμό που θα τους επιτρέψει να λάβουν αποφάσεις πιο γρήγορα και επίσης ε, θα μπορούσε να γίνει και ένα είδος δοχή όπου άλλοι θα μπορούσαν να έλθουν, δηλαδή κάποιοι μικροί δωρητές και κάτι τέτοιο θα μπορούσε να βοηθήσει το συνολικό επίπεδο χρηματοδότησης. Όμως καλύτερα να απαντήσουν οι συνάδελφοι από την ΤΕΦΚΟ για αυτό το θέμα, θα επανέλθουν σε αυτό το θέμα, να είστε βέβαιοι. Τώρα, σε γενικές γραμμές, ε, ε, η μιστούρα έχει ε, ε, ταξιδέψει στην περιοχή, επέστρεψε και μας στο Βερολίνο ότι η έκφραση που άκουγε συνέχεια ήταν «χαλάσει καλάς» σημαίνει ότι φτάνει πια, έχουμε βαρεθεί. Από παντού άκουγε την έκφραση αυτή, από ανθρώπους που είναι κοντά στην κυβέρνηση της Συρίας, από ανθρώπους της αντιπολίτευσης, από γυναίκες, ομάδες γυναικών, από ανθρώπους που θέλουν δημοκρατία, από πιο φοντομεταλλιστικές ομάδες. Όλοι ε, θεωρούν ότι φτάνει πια και νομίζω ότι η ικανότητα να το αντιμετωπίσουν ε, αυτή την κατάσταση έχει κορεστεί. Αυτό τώρα να μας δίνει κάποια ελπίδα δεν ξέρω. Αυτό τώρα που προσπαθούμε να δούμε ε, είναι το εξή. Βλέπουμε ότι ε, η πολιτική σε μεγάλο επίπεδο δεν προχωρά. Έτσι λοιπόν ίσως θα πρέπει να δημιουργήσουμε κάποια μικρότερα παράθυρα εγώ πιστεύω ότι χρειαζόμαστε πολιτικές λύσεις και ο ρόλος μας είναι να εργαστούμε για αυτές από κοινού και βλέπω ότι και η κυρία Μογκερίνη έχει αναλάβει δεσμεύσεις στον τομέα αυτό θέλουμε να τα συζητήσουμε τα θέματα αυτά και αν θέλουμε να σώσουμε ζωές, νομίζω ότι κάποιοι ε, θα πρέπει να κάνουν και κάποιες υποχωρήσεις. Ε, νομίζω ότι ίσως χρειαζόμαστε κάποιο νέο σκεπτικό για το πώς να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Γιατί δεν θα ήθελα να επανέλθω σε ένα χρόνο και να έχουν σκοτωθεί 100.000 άτομα ακόμα. και να έχουν αποκεφαλιστεί και άλλα άτομα από τη τα κτλ. Είμαστε πραγματιστές λοιπόν, ε, ανθρωπιστικοί διάδρομοι, ζώνε προστασίας. Ναι, εγώ είμαι θετικό, αλλά δυστυχώ γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι να γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ποιο θα διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχει μια νέα σεμπρένιτσα Δηλαδή, ναι, μπορούμε να κάνουμε κάποιε δράσει, αλλά και ξαφνικά κάτι γίνεται. Είναι πολύπλοκο, ακούγεται κάτι καλό, αλλά στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ δύσκολο και πρέπει να είμαστε ειλικρινέ, Δεν βάζουμε του ανθρώπου σε κίνδυνο, λέγοντα ότι θέλουμε να κάνουμε το ένα και το άλλο και ποιο ξέρει τι. Και πάλι για την πολιτική. Η πρώτη συνάντηση ΡΕΛΕΞ θα λάβει χώρα την Τετάρτη. Νομίζω ότι θα συζητηθεί το θέμα της Ουκρανίας, ο ιός του έμπολα και πιθανότατα η Συρία και νομίζω ότι εστιάζουν σε όλα αυτά και θέλουν να υπάρχει πρόοδος. Σε ό,τι αφορά το θέμα της επαναγκατάστασης και της βούλησης να δεχτούμε προσφύγους, το Δυσάρεστα είναι ότι ο κύριος Γκουτιέρες, ο οποίος ε, υπερασπίζει τους πρόσφυγες ξέρω ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μας ζητά εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δεχτούμε 130.000 πρόσφυγες. Τώρα έχουμε κάποιες δεσμεύσεις για 33.000. Σαφέστατα, υπάρχει μεγάλη απόσταση. Ε, ελπίζω ότι σύνοδος τη 9 η Δεκεμβρίου θα σημειώσει κάποια πρόοδο για τα νούμερα αυτά, όμως ε, αυτό πρέπει να είναι ένα μέτρο μεταξύ άλλων, γιατί δεν μπορούμε να δεκτούμε και τα 3,7 εκατομμύρια, ξεχάστε το. Μπορούμε να κάνουμε μία συνεισφορά και θα έπρεπε νομίζω, νομίζω ότι θα έπρεπε να σεβαστούμε αυτό το καθήκον, να αναλάβουμε αυτό το καθήκον. Ε, τώρα σε ό,τι αφορά τα χρήματα, σας ευχαριστώ για την υποστήριξη, πραγματικά ένθερμα. Ε, σας ευχαριστώ για τη δουλειά που κάνετε, να συνομιλήσετε με τους υπουργούς οικονομικών σας. Ε, είναι ιδιαίτερα πολύτιμο έργο αυτό, γιατί όπως είπατε κι εσείς, δεν ξέρω αν μπορώ να συνεχίσω τρει μήνε ή αν θα έπρεπε να μειώσω τις συμβάσεις το ίμιση στις αρχές του έτους, γιατί αυτά μπορώ να χρηματοδοτήσω εκ των προτέρων. Και ξέρετε, γιατί μετά θα ξέρουμε τι θα γίνει με τις αποφάσεις που πρέπει να λάβουμε. Εγώ πιστεύω με τη Δημοσιονομική Αρχή ότι θα λάβουμε τα χρήματα, ας μην βανικοβαλόμαστε, πρέπει να γίνει. Διαφορετικά δεν ξέρω πώς μπορώ να επιλύσω την κατάσταση. Είμαστε ενεργοί, η Κρυσταλίνα Τζορτζίβα, την οποία πάλι θέλω να ποτίσω φοροτιμής, είναι ικανοποιημένη που ε, κάναμε μία συνδιάσκεψη όπου είχαμε τη δεσμεύση ενός δισεκατομμυρίου. Ξέρω ότι θα χρειαστεί χρόνος, όμως υπήρχε ε, υπήρχαν χρήματα που δόθηκαν και από τις χώρες του κόλπου και από αλλού. Έτσι λοιπόν είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Δεν είμαστε μόνο εμείς λοιπόν, αλλά και άλλοι δωρητές που θα πρέπει να συνεισφέρουν. Τώρα, αν θέλετε να πω κάτι για την ανάπτυξη, τα ανθρωπιστικά θέματα και το σύνδεσμο μεταξύ αυτών. Σίγουρα πρέπει να συνεργαστούμε. Είμαι πεπισμένο και είμαι πεπισμένο πως όταν έχουμε μια τέτοια κρίση στο Λίβανο και στην Ιορδανία, όχι στη Συρία, στη Συρία είναι διαφορετικά τα πράγματα, αλλά για τις άλλες δύο χώρες ε, θα πρέπει ε, να συνδεθούμε με τα εθνικά αναπτυξιακά σχέδια, γιατί δεν να έχουμε αποτελέσματα και να προσφέρουμε εκπαίδευση στους πρόσφυγες ε, εκτός του σχολείου είναι κάτι πολύ πιο ακριβό από το να λειτουργούν τα σχολεία και επίσης είναι καλύτερα να λειτουργούν τα συστήματα υγείας για να προσφέρουν τις υγειονομικές υπηρεσίες. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να έχουμε αναπτυξιακά χρήματα και τα, τα χρήματα για ανθρωπιστική βοήθεια θα πρέπει να έρχονται σε συνέργεια αυτών και ίσως ε, θα ε, μπορέσουμε έτσι να επιτελέσουμε το καθήκον μας. Και αυτό είπα και στο Βερολίνο, ότι χρειαζόμαστε πολύ καλύτερο και ολοκληρωμένο σχεδιασμό μεταξύ των οργανισμών και των εθνικών αρχών και της Παγκόσμιας Τράπεζας κτλ. κτλ. Θα σταματήσω εδώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Κλάους. Δύο λεπτά το πολύ για να απαντήσετε, κύριε Ναι, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας πω δύο λόγια για την κατάσταση όσον αφορά την πρόσβαση. Για να δούμε την πρόσβαση, θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες βελτιώσεις από πλευράς ε, Δαμασκού για τα ε, μετά το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών που επιτρέπει τις διαμεθοριακές δραστηριότητες. Μπορεί να έχει καλύτερη πρόσβαση ε, είπατε αμορμοστεί από πλευράς ε, Δαμασκού, αλλά όσον αφορά τις ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις, ε, η κατάσταση είναι τελείως αντρίστροφη. Έχουμε εκθέσεις από συναδέλφους στη Δαμασκού που αντιμετωπίζουν τελείως διαφορετικά προβλήματα όσον αφορά την πρόσβαση. Και σε όλη την περιοχή εντός της Συρίας το γεγονός ότι πλέον υπάρχουν πολύ μεγάλες περιοχές που ελέγχονται από τον Ισλαμικό στρατό και στη Συρία και στο Ιράκ, περιοχές στις οποίες υπολογίζουμε ότι ζουν περίπου 6 εκατομμύρια άνθρωποι, το μήνυμα το οποίο ε, λαμβάνουμε είναι ότι δεν είμαστε ευπρόσδεκτοι, πρέπει να κρατηθούμε μακριά. Και αυτό είναι το ένα και το άλλο είναι ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Επομένως θα πρέπει να δούμε τώρα ποια είναι η λύση προκειμένου να παράσχουμε βοήθεια σε αυτά τα 6 εκατομμύρια ανθρώπων που ε, κατά πάσα πιθανότητα βρίσκονται σε ακραίες ε, συνθήκες. Ευχαριστώ κύριος Χοντσούλ. Ναι, τρεις πολύ σύντομες παρατηρήσεις ε, όσον αφορά την πρόσβαση. Ο, ο κύριος Νόγερ αναφέρθηκε σε αυτό. Κύριε Νόγερ, νομίζω ότι σας είπα ότι μέσω ε, της δικής μας της κοινότητας και μέσω κάποιων άλλων ενδιαμέσων καταφέραμε να έχουμε κάποια πρόσβαση. Είναι περιορισμένη, σίγουρα δεν είναι ικανοποιητική, αλλά ε, έχουμε μια αρχή και ελπίζουμε ότι θα έχουμε περισσότερα. Η μόνη εξαίρεση είναι η περιοχή του Αλασά και μάλλον ε, στα βόρειο-ανατολικά, όπου δεν ε, έχουμε δυνατότητα πρόσβασης μέσω της νότιας οδού γιατί τα πράγματα είναι πολύ επικίνδυνα και επίσης αυτή τη στιγμή ε, προσπαθούμε να ανοίξουμε μια άλλη οδό από τα βόρεια μέσω των συνόρων με την Τουρκία αλλά χρειάζονται κάποιες διαπραγματεύσεις οι οποίες είναι εξελίξει βέβαια και ακόμα δεν έχουν ε, αποφέρει καρπούς όσον αφορά τους διαδρόμους και τη περιοχή buffer, ε, να σας πω ότι θα υπάρξει συμμετοχή αν όλες οι πλευρές οι οποίες μπορεί να έχουν είτε μερικό είτε συνολικό έλεγχο στην περιοχή συμφωνήσουν ε, με κάποιες ελάχιστες εγγυήσεις και κάποιους τρόπους ε, διεξαγωγής των πραγμάτων, αλλιώς αποκλείεται να μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση γιατί θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Αυτή τη στιγμή ε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και μια τελευταία παρατήρηση τώρα για μια δυνατότητα ανακοχή που ίσως θα είναι ένας τρόπος να αρχίσουμε σιγά σιγά να δημιουργούμε κάποιες περιοχές στις οποίες θα επικρατεί η ειρήνη. Εμείς βέβαια δεν συμμετέχουμε σε ειρηνικτικές διαπραγματεύσεις. Ε, αλλά προσπαθούμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας ως ουδέτερος ενδιάμεσος ε, για την παροχή τροφίμων, ε, φαρμάκων, ε, την απομάκρυση κάποιων ανθρώπων ή να διευκολύνουμε ίσως κάποιες ανταλλαγές κρατουμένων. Υπάρχουν κάποιες συζητήσεις λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Okay, thank you very much. We should be grateful to both of you for coming here. Σας ευχαριστώ λοιπόν που ήρθατε όλοι εδώ σήμερα για την ευχαριστώ και τις οργανώσεις σας. Εύχομαι κάθε επιτυχία και εύχομαι να υπάρχει ευρύτατη υποστήριξη για το έργο που κάνετε επί τόπου. Υπό πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σόρενσεν, ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ γεμάτη η ατζέντα σας. Θα ακούσουμε και πιο πολλά θέματα. Έχουμε και την πρώτη, επιτροπή, την πρώτη ημέρα του νέου επιτρόπου. Θα σας δούμε τις επόμενες εβδομάδες για να μας ενημερώσετε τι γίνεται σε αυτό το πάρα πολύ δύσκολο θέμα επί το οποίο εργάζεστε σήμερα και νομίζω ότι η συζήτηση νομίζω ότι θα πρέπει να κινηθεί προς την πολιτική κατεύθυνση από πλευράς της Ολομέλειας σε ό,τι αφορά τις πολιτικές ομάδες χωρίς πολιτική λύση δεν θα υπάρξει πραγματική λύση στη Συρία. Αν λοιπόν οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε εδώ για να υποστηρίξουμε τις οργανώσεις που εργάζονται επί τόπου, σας παρακαλώ ενημερώστε μας κατά πόσον η Επιτροπή μας μπορεί να κάνει κάτι για να περάσει πιο πολύ βοήθεια σε αυτούς που τη χρειάζονται. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφοι, έχουμε μείνει πίσω. Ε, καθυστερήσαμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και θα περάσω κατευθείαν στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό τι σημαίνει ότι θα καθυστερήσουμε την ψηφοφορία πιο αργά από ό,τι προβλέπετε λοιπόν. Αν έχετε λοιπόν άτομα τα που έρχονται ε, για την ψηφοφορία, που θέλουν να έρθουν μόνο για την ψηφοφορία, δεν θα ψηφίσουμε πριν από τις 5 και 4. Η επόμενη συζήτηση τώρα έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Παγκόσμιο Πλαίσιο Ανάπτυξης για την περίοδο μετά το 2015. Σήμερα λοιπόν θα συζητήσουμε για την έκθεσή μας η οποία θέλει να συμβάλλει τη δική μας άποψη πριν από τα συμπεράσματα του Συμβουλίου το Δεκέμβριο. Ο κύριος Στήρη λοιπόν είναι ο υπεύθυνο, ο αρμόδιος συζητητής. 406 ε, τροπολογίες έχουμε. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε συμβαστικές λύσεις για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε. Να πω όμως το εξή στους συναδέλφους. Δεν χρειάζεται να τα πούμε όλα εδώ στην έκθεση αυτή. Το θέμα είναι να δώσουμε κάποια σαφή μηνύματα προς το Συμβουλίο. Αν είναι υπερβολικά πολύ άριθμα τα μηνύματα αυτά, πολύ απλά θα χαθούν στην όλη συζήτηση. Ας επικεντρωθούμε σε μηνύματα κλειδιά προς το Συμβούλιο. Πώς θέλουμε να αξιοποιηθεί η διαπραγματευτική μας θέση για το 2015. Νομίζω λοιπόν να περιοριστούμε σε αυτά θα βοηθήσει πολύ. Να δώσω το λόγο στον κύριο Στήρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ για να ολοκληρωθεί εγκαίρως η συζήτηση αυτή, πριν την ψηφοφορία. Εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια θεματικά θέματα παρόλα αυτά, σε ό,τι αφορά την έκθεση αυτή. Όπως τα ξέρετε όλοι, αυτό θα είναι το μήνυμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου και μάλιστα θα καθορίσει έτσι τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οποία ασφαλώς θα ενισχυθεί στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε λοιπόν ισχυρή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από τις διακυβερνητικές διαπραγματεύσεις σε ό,τι αφορά το νέο πλαίσιο που θα εγκριθεί του χρόνου. Αυτό για να τονίσω τη σημασία του να ψηφιστεί η έκθεση αυτή πριν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Στο, στην Ολομέλεια του Νοεμβρίου. Προκειμένου να υπάρχει και κάποιο αποτέλεσμα στην κοινή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι η διαδικασία ως τώρα ήταν πολύ συνεκτική και περιέλαβε, περιέλαβε πάρα πολλέ απόψεις. Έγινε διάλογος μεταξύ των πολιτικών ομάδων, μεταξύ σκιωδών, αλλά και σε ό,τι αφορά τις διαβουλεύσεις και τον ανοιχτό διάλογο που διεξήχθησε με μη κυβερνητικές οργανώσεις, με διάφορες ε, άλλες οργανώσεις και βλέπετε ότι οι απόψεις τους ε, αποτυπώνονται στις πολλές τροπολογίες που κατατέχθηκαν. 466 λοιπόν στον αριθμό τροπολογίες, πάρα πολλέ. Αυτό θεωρώ ότι επιβεβαιώνει απλά τη σημασία, τη σπουδαιότητα του θέματος, αλλά και το πόσο συνολική και ευρεία ήταν η προσέγγιση μας. Αποτυπώνονται όλες οι διαφορετικές ε, απόψεις. Τώρα, πλέον φυσικά έχει φτάσει η στιγμή που θα πρέπει να κάνουμε συμβιβασμούς, θα γίνει και η συνάντηση των σκιωδών την Τετάρτη. Καλό λοιπόν τους συναδέλφους μου να δείξουν πνεύμα σε μοιβασμό, γιατί θα χρειαστεί, αν θέλουμε να ψηφίσουμε εδώ στην Επιτροπή εγκαίρως. Όχι μόνο λόγω των χρονικών περιορισμών, ωστόσο, αλλά πρέπει να υπάρχει διάθεση συμβιβασμού για να στείλουμε και ένα σαφέ μήνυμα. Αν ακολουθήσουμε την προσέγγιση του χριστιανιάτικου δέντρου, τα βάζουμε όλα μέσα, θα αποδυναμωθεί το μήνυμά μας. Α προσπαθήσουμε λοιπόν να συμπεριλάβουμε όλα αυτά που έχουν προταθεί, αλλά να θέσουμε προτεραιότητες πλέον, προκειμένου να είναι σαφές το μήνυμά μας. Ένα από τα βασικά λοιπόν θέματα, για να μπούμε σε θέματα ουσίας, είναι η σημασία της προσέγγισης βάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο νέο πλαίσιο ανάπτυξης μετά το 2015. Και αυτό γιατί. Όχι επειδή πρόκειται για τη μοναδική προτεραιότητα. Προφανώς μας απασχολεί κατ' πρωτίστως η κατάργηση της φτώχειας. Αλλά μετά από μια κανονική, σωστή πολιτική ανάλυση, βλέπουμε ότι το αποτέλεσμα των εργασιών της ανοιχτή ομάδας εργασίας είναι ότι πρόκειται για έναν από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που δέχεται τα βέλη της κριτικής πιο πολύ από τους υπόλοιπους στόχους. Θέλουμε λοιπόν να παραμείνει αυτό, να είναι φωνή εντυρήμων δική μας φωνή και να παραμείνει αυτό ως προτεραιότητα. Θα πρέπει λοιπόν να είναι επιτακτική η προτεραιότητα αυτή και γι' αυτό λοιπόν έχει τόσο πρωτεύουσα θέση στο κείμενο. Και γι' αυτό λοιπόν το θέτουμε αυτό ως προτεραιότητα αμέσως μετά από την καταπολέμηση της ένδυας και μετά τους τρεις πυλώνες βιώσιμης ανάπτυξης. Θέτουμε λοιπόν ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα αυτό, το θέμα της ασφάλειας και της ειρήνης. Και αυτό αναφέρεται στους στόχους του 2016 στο έγγραφο του OWG. Και αυτό φυσικά απασχολεί ιδιαίτερα τα άτομα που βρίσκονται σε τέτοια ευάλωτα κράτη, γιατί εκεί δεν υπάρχει πιθανότητα και δυνατότητα ανάπτυξης χωρίς ασφάλεια και ειρήνης. Γι' αυτό λοιπόν προωθούμε το θέμα αυτό, για να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα. Σε κάποιες περιπτώσεις όσο λιγότερα λέμε τόσο πιο πολλά εννοούμε. Γιατί εάν δεν πλατιάσουμε νομίζω ότι θα είναι πιο σαφές το μήνυμα που θα στείλουμε και θα γίνει πιο καλά κατανοητό και από το Συμβούλιο αλλά και από την γενικότερη, την ευρύτερη, την εθνική κοινότητα που ασφαλώς θα αναλύσει το, το έγγραφο αυτό που θα αποτελέσει την τοποθέτηση του Κοινοβουλίου. Τώρα, λοιπόν, περνάμε από τα MDG στα SDG. Υπάρχει μια αξιολόγηση και είναι σαφές ότι το νέο πλαίσιο θα πρέπει να καταπολεμήσει τη ρίζα της στόχιας και ότι θέλουμε να ολοκληρώσουμε όσα δεν έχουν ολοκληρωθεί σε ό,τι αφορά τους στόχους της χιλιετίας. Επιλέγουμε λοιπόν τέτοια θέματα. Και αποστέλουμε το μήνυμα του που έγκυται οι προσωριότητες μας σε ό,τι αφορά τα πολιτικά συνθήματα. Όπως ξέρετε λοιπόν, ε, περιμένουμε και από τον ε, νέο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να παράγει να μας ε, δημοσιεύσει το σχετικό του έγγραφο. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να μεταφέρουμε το μήνυμα αυτό. Μιλάμε ασφαλώς όχι μόνο στον τομέα των προτεραιοτήτων για την ε, εξάλληψη της στόχης και για τη βιώσιμη ανάπτυξη ως ε, οριζόντιο στόχο. Μιλάμε και για το θέμα της ανισότητας ως ένα από τα βασικά ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στο νέο πλαίσιο. Και επίσης τονίζουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει η προσέγγιση βάσει των δικαιωμάτων. Δεν πρόκειται να επισέλθω στους διάφορους ε, τίτλους. Θα το συζητήσουμε και στην συνεδρίαση των σκιωδών την Τετάρτη. Θα συζητήσουμε τους διάφορους προτινόμενους εμβιβασμούς. Ελπίζω να μπορέσω να σας αποστείλω πιο πολλά στοιχεία μέχρι αύριο. Αλλά θεωρώ ότι επίσης σημαντικό είναι να πούμε το εξής. Στην έκθεση μιλάμε για το κεντρικό ρόλο των γυναικών στο νέο πλαίσιο ανάπτυξης. Και εδώ θέλουμε να πούμε ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται για θέμα του, της εξάλληψης των ανισοτήτων απλά. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο υπερβαίνει τα όρια της ανισότητας. Μιλάμε για τον κεντρικό ρόλο των γυναικών στην ανάπτυξη και στην ατζέντα της ανάπτυξης, γιατί αυτό άπτεται πολλών διαφορετικών τομέων της ανάπτυξης. Ένα άλλο θέμα το οποίο υπογραμμίζεται είναι το θέμα του OPCD γιατί δίχως αυτό δεν θα είναι δεν θα είναι δυνατόν να υπάρχουν πραγματικοί στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα γνωρίζετε ότι η έκθεση αυτή στην πρώτη της ε, στο πρώτο της σχέδιο έχει πολύ περιορισμένο αριθμό λέξεων και γι' αυτό δυστυχώς αναγκαζόμαστε να κάνουμε τόσες πολλές τροπολογίες. Αυτό εξηγεί εν μέρη γιατί υπάρχουν τόσες πολλές τροπολογίες. Ένα θέμα επίσης είναι του να γνωρίζουμε πόσο καθολικό είναι το νέο πλαίσιο, προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμπεριλάβει στο ιστορικό της τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Στο τέλος φυσικά υπάρχει ένα δίλημα. Να το πω ξεκάθαρα. Στο παρελθόν, στην Επιτροπή εδώ, συζητήσαμε το θέμα του υπαριθμό 16 στόχου. Και είπα εξ αρχής ότι στη διεθνή συζήτηση έχει συγκεντρώσει τα βέλη της κριτικής αυτός ο στόχος. Υπάρχει λοιπόν ο φόβος ότι αν μιλήσουμε για την ιδέα, την ιδέα της μείωσης ε, των ε, στόχων, προφανώς ο στόχος υπαριθμών 16 θα είναι ο πρώτος, από του πρώτους εν πάση περιπτώσει που θα διαγραφεί από τη λίστα. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν το επιθυμούμε. Από την άλλη, Έχουμε πολλούς συναδέλφους που θα ήθελαν να υπάρχει σημαντική μείωση, σημαντική απλούστευση των στόχων, ακολουθώντας τη λογική του ότι αν υπάρχουν 17 προτεραιότητες, τίποτα τελικά δεν αποτελεί σαφή προτεραιότητα. Πολύ απλά λοιπόν ότι θα πρέπει να περιορίσουμε τον αριθμό των προτεραιοτήτων. Υπάρχει λοιπόν μια ε, αντίφαση στο σημείο αυτό των δύο αυτών στόχων, αντικρουόμενοι ο συμβιβασμό που θα ήθελα να προτείνω. Και θα κλείσω με αυτό. Η πρόταση της ανοιχτής ομάδας εργασίας θα μπορούσε να απλουστευτεί. Όχι όμως εις βάρος της προσέγγισης βάσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να αποτελεί ένα μήνυμα που θα αποστείλουμε ως Κοινοβούλιο. Δεν είμαστε κατά της αρχής να, του να μειωθεί ο αριθμός των στόχων σε ό,τι αφορά τις διακυβερνητικές ε, διαπραγματεύσεις. Όχι όμως εις βάρος της προσέγγισης βάσει ανθρωπινών δικαιωμάτων. Και νομίζω ότι έτσι μπορούμε να επιλύσουμε αυτό το δίλημα, αυτή την αντίφαση που αντιμετωπίζουμε. Κλείνοντας. Όπως σας είπα, Βρισκόμαστε στην ε, φάση όπου ο χρόνος ε, μετράει πλέον. Αν καθυστερήσουμε τις διαπραγματεύσεις μας, διακινδυνεύουμε τελικά να μην υπάρξει ψήφισμα, να μην υπάρχει σαφές μήνυμα. Ο χρόνος περνάει και δεν είναι υπέρ μας. Έχουμε την συνεδρίαση των σκιωδών την Ελπίζω να είναι παραγωγική αυτή η συνάντηση και να συμπεριληφθούν οι διαφορετικές απόψεις αλλά στο τέλος ελπίζω οι συμβιβασμοί που θα επιτευχθούν να αποστείλουν ένα σαφές μήνυμα για το ποιες είναι οι προτεραιότητες και ποια είναι η θέση του Κοινοβουλίου μας. thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Καταρχήν θα δώσω το λόγο στους σκιώδεις εισηγητές και κατόπιν ε, θα περάσουμε στην ανοιχτή συζήτηση για τους σοσιαλιστές. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη δουλειά του. Αποτελεί μια καλή βάση εφετερία. Η ομάδα μα προσπάθησε να καταστήσει ακόμη πιο φιλόδοξο το κείμενο και να προσδιορίσει κάποιε προτεραιότητε όπου πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε να επηρεάσουμε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου. Είχαμε λίγο χρόνο, αλλά εργαστήκαμε καλά και παρουσιάσαμε πάνω από 100 τροπολογίε. Νομίζω ότι στη συζήτηση εμεί θα πρέπει να πάρουμε τα συμπεράσματα τη Ανοιχτή Ομάδα Εργασία σε βάση αφετηρία όχι να προσπαθήσουμε να τι γράψουμε εκ νέου, αλλά να προσπαθήσουμε να δώσουμε έμφαση σε κάποιες προτεραιότητες και να ζητήσουμε πιο ε, καινοτόμοι στόχοι να μην ε, ε, παραγωνιστούν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Εδώ συμφωνώ απόλυτα επί της ιδέας ότι μία πιθανή μείωση των ε, αριθμών ε, των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης μάλλον θα σε κίνδυνο ε, τους στόχους που μας ε, είναι οι πιο σημαντικοί και αναφέρομαι στην ισότητα ε, των δύο φύλων και στην ισότητα γενικά. Έτσι λοιπόν έχουμε προτείνει να αναδιαρθρώσουμε το κείμενο έτσι ώστε να τονίσουμε πόσο σημαντική είναι η παγκόσμια εταιρική σχέση και να μπορέσουμε να έχουμε μια ισχυρή θέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Έχουμε προτείνει και ένα τελευταίο κεφάλαιο που να ενώνει τα μέσα τη εφαρμογή σε ένα σημείο που θα είναι κεντρικό στι διαπραγματεύσει, δηλαδή πώ καταπολεμούμε τη φοροδιαφυγή, τη διαφθορά και πώ εμπλέκεται η κοινωνία των πολιτών, οι τοπικέ αρχέ και τα εθνικά κοινοβούλια. Επιμείναμε στην καταπολέμηση των ανισοτήτων. Κανένα στόχο δεν θα θεωρείται ότι έχει επιτευχθεί αν δεν καλύπτει καλύπτει όλες τις κοινωνικές ομάδες. Από ό,τι βλέπω και άλλες ομάδες έχουν τονίσει αυτό το θέμα. Θα πρέπει η ανισότητα να καταπολεμηθεί σε όλη, κάθε της μορφή και όχι μόνο ως προς το εισόδημα. Μείναμε στο ρόλο των γυναικών, των παιδιών και των μειονοτήτων και στη διασύνδεση μεταξύ ανάπτυξης και κλιματικής αλλαγής. Επίσης, ε, μείναμε στην προσέγγιση που βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως είπε και ο συγητής. Επίσης, τον κεντρικό ρόλο της υγείας και της παιδείας ε, ως κυρία δικαιώματα, όπως και στα δικαιώματα αναπαραγωγής. Ε, θέλουμε να υπάρχει πλήρη σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της αρχής της λογοδοσίας. Σε αυτή τη βάση είμαστε έτοιμοι να βρούμε συμβιβασμούς πεπισμένοι ότι αυτά τα θέματα και αυτές οι προκλήσεις ενδιαφέρουν όλες τις ομάδες. Ε, θέλουμε να καταλήξουμε σε μια ισχυρή θέση αυτού του Κοινοβουλίου και να υπάρχει και η μεγαλύτερη δυνατή πλειοψηφία στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φεράινεν για τους φιλελευθέρους. Λίντα. Πρόεδρε. Και η ομάδα των φιλελευθερών έχει καταθέσει κάποιες τροπολογίες. Ε, έχω καταθέσει κάποιες τροπολογίες και εγώ ίδιος. Θα μιλήσω μόνο για μία τροπολογία, η οποία αφορά το, θέμα της επαναδιοργάνωσης των ε, στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Η Κομισιόν στην ανακοίνωσή της δήλωσε ότι υπάρχει μια αναγκή των στόχων. Στο σχέδιο έκθεσης έχουμε την παράγραφο 32. Χαιρετίζει την πρόεδρο που έχει σημειώσει η νυχτή ομάδα εργασίας, αλλά θεωρεί ότι ο ρυθμός των στόχων που καθορίζονται στα συμπερασματά πρέπει να πλουστευτεί και να μειωθεί σημαντικά. Ποτέ δεν πρότεινα μείωση. Εγώ Απλώς μίλησα για επαναδιοργάνωση των στόχων αυτών. Εγώ νομίζω ότι θα μπορούσαν να είναι πάνω από 17. Όμως ε, ήδη, <laughs> γιατί 17 είναι χριστουγεννιάτικο δέντρο, είναι πάρα πολύ και από ό,τι φαίνεται θα έχουμε όλο ένα και περισσότερα στολίδια, αλλά δεν έχουμε δέντρο. Δεν έχουμε κλαδιά ούτε κορμό. Και γι' αυτό εγώ πρότεινα μια αναδιοργάνωση των στόχων υπό τους τίτλους «Μείωση της στόχιας», «Πρόθεση της βιώσιμης ανάπτυξης, οικολογικής, ε, περιβαλλοντικής ε, κτλ. και παγκόσμια εταιρική σχέση. Δεν, μίλησα για, δεν μίλησα για μείωση λοιπόν, μόνο για αναδιοργάνωση. Έχω λοιπόν καταθέσει μια σχετική τροπολογία. Ε, βέβαια είναι κάπως αόριστη διατύπωση έτσι ώστε να μπορεί να ερμηνευτεί με διάφορους τρόπους. Νομίζω ότι δεν είναι πολύ αργά για να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι και ελπίζω ότι το Συμβούλιο και η Κομισιόν θα μπουν σε διαπραγμάτευση. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω και τι είπε ο εκπρόσωπος της Αφρικανικής Ένωσης στη συνεδρίασή μας. Η Αφρικανική Ένωση έχει καταθέσει έξι προτεραιότητες, έχει προτείνει έξι στόχους. Θα μπορούσαμε ίσως να μάθουμε κάτι και από αυτούς. Ελπίζω λοιπόν ότι δεν θα υπάρχει παρανόηση, όχι μείωση, αλλά αναδιοργάνωση, ακόμη και προσθήκη σημαντικών στόχων στον κατάλογο των 17. Δεν μπορώ να παρευρεθώ στην ομάδα των σκέντων συγητών, αλλά ελπίζω ότι οι άλλες ομάδες θα υποστηρίξουν την τροπολογία μου περί αναδιοργάνωσης των στόχων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Σάντσες εξ ονόματος της Ενωτικής Αριστεράς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Βεβαίως και βιώνουμε στιγμές οι οποίες είναι ζωτική σημασίας ε, για το πλαίσιο για το 2015 και θεωρούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχουν μια ενωμένη θέση για να δείξουμε ότι είμαστε ένας ε, αξιόπιστος τέρος σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Εμείς θεωρούμε ότι υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία θα πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα. Πιο συγκεκριμένα είναι τρία. Η φτώχεια, η οποία θα πρέπει να πάψει να θεωρείται σε ένας παράγοντας ο οποίος ε, αφορά απλώ και μόνο το εισόδημα, διότι είναι πολλές οι διαστάσεις του και θα πρέπει να σταματήσουμε να το βλέπουμε μόνο με πρίσμα το εισόδημα. Επίσης ε, θα πρέπει να δούμε και τις ανάγκες των ανθρώπων όταν θα καθορίσουμε τους δείκτες, αλλά και τα μέτρα για να ε, εφαρμόσουμε το πλαίσιο. εάν δεν βασιζόμαστε στους ανθρώπους δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και πέρα από αυτό, οι στόχοι θα πρέπει να είναι η ισότητα και η έλλειψη διακρίσεων, διότι αυτά είναι πολύ σημαντικά προκειμένου να μπορέσουμε να μειώσουμε τις κοινωνικές εντάσεις, να ενισχύσουμε την ειρήνη και τη σταθερότητα. Γι' αυτό ακριβώς και θεωρούμε ότι θα πρέπει να επιτεθούμε στις ρίζες της ανισότητας, οι οποίες δεν είναι μόνο οικονομικές, αλλά και πολιτικές και κοινωνικές. Και επομένω οι τροπολογίε μας είναι προς αυτή την κατεύθυνση και ελπίζουμε ότι το Συμβούλιο θα τις λάβει υπόψη και θα υπάρξει μεγάλη υποστήριξη από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις τροπολογίες αυτές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Μαρία Χόιμπουκ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχουμε πάνω από 400 ε, τροπολογίες, αλλά από τη συζήτηση φαίνεται ότι υπάρχουν πολλές ε, επικαλύψεις και έτσι θα μειωθούν αυτόματα οι τροπολογίες. Κοιτώντα λοιπόν την έκθεση και θέλοντα, όπω είπατε, να αποστείλουμε ένα σαφέ μήνυμα, θα πρέπει να τη διαμορφώσουμε λοιπόν όσο πιο επακριβώς γίνεται την έκθεση αυτή. Ένα παράδειγμα, λέτε ότι οι γυναίκες είναι πολύ σημαντικέ. Θα πρέπει λοιπόν στο πλαίσιο αυτό να αναφέρουμε τα δικαιώματα συγκεκριμένα των γυναικών. Κάτι άλλο τώρα. Οι τρεις σημαντικοί πυλώνες. Περιβάλλον, κοινωνία και οικονομία. Θα πρέπει όλα αυτά να αναφερθούν προκειμένου με βιώσιμο τρόπο να συνεχίσουν να αναπτύσσονται. Και ως βάση θα ήθελα να αναφέρω την ομάδα εργασίας του ΟΗΕ και τη σχετική έκθεση να αναφερθούν συγκεκριμένα κάποιοι, κάποιες ομάδες στόχοι όπως οι γυναίκες, όπως οι γεωργοί, οι μικροί γεωργοί. Αν είναι λοιπόν τόσο σημαντική αυτή η προσέγγιση βάσει του ανθρώπου, θα πρέπει πάντα να συμπεριλαμβάνεται στους στόχους και να περιγράφεται ως τέτοια. Και θέμα των ανισοτήτων που αναφέρθηκαν αποτελεί σημαντικό ζήτημα και αυτό θα πρέπει λοιπόν να αναφέρεται στους, κάθε, στους όλους τους μεμονωμένους στόχους. Ένας άλλος στόχος που και αυτός δεν θα πρέπει να χαθεί είναι η αλλαγή του κλίματος. Η αλλαγή του κλίματος θα είναι πάρα πολύ σημαντική, σημαντικός παράγοντας για το τι συμβαίνει στις χώρες αυτές και γι' αυτό λοιπόν και ο στόχος λοιπόν αυτός θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνεται. Μίλησα και για τα δικαιώματα των γυναικών. Κάτι άλλο που με απασχολεί είναι η γεωργία. Όχι μόνο παραγωγική αλλά και βιώσιμη γεωργία και ιδιαίτερα ο ρόλος των μικρών γεωργών, τους οποίους και θα πρέπει να υποστηρίξουμε και να τους προστατεύσουμε σε ό,τι αφορά τα δικαιώματά τους, πρόσβαση στο νερό, πρόσβαση στους πόρους, τέτοια δικαιώματα. Όλα αυτά θα πρέπει να αναφέρονται στην έκθεση. Μιλώντας για ανάπτυξη δε, η ανάπτυξη αυτή θα πρέπει να αναφέρεται και στα πλαίσια των περιορισμών που επιβάλλει ο πλανήτης μας. Γιατί δεν είναι αένα η, η ανάπτυξη. Τα ευάλωτα κράτη, σημαντικό ζήτημα. Ένα άλλο θέμα που σας απασχολεί ιδιαίτερο είναι το θέμα της χρηματοδότησης. Γιατί δεν θα πρέπει να αναφέρεται μόνο ότι δεν θα πρέπει να μειωθεί η χρηματοδότηση. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το 0,7% του ΑΕΠ όλων των κρατών θα πρέπει να χορηγείται προς την κατεύθυνση αυτή και αυτό να αποτελεί την βάση παράνομες ροές χρημάτων. Θα πρέπει να το προσέξουμε το θέμα αυτό ιδιαίτερως και κατά πόσον το ΑΕΠ θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για τους στόχους ανάπτυξης, να το εξετάσουμε και αυτό ως μία δυνατότητα ή θα πρέπει να βρούμε μία εναλλακτική. Άλλους μηχανισμούς εποπτείας σε ό,τι αφορά την επιτήρηση των ροών χρημάτων. Άλλο σημαντικό θέμα για μας η θέση ενός μόνιμου εισηγητή δεν είναι σημαντικό μόνο να στείλουμε τώρα ένα σημαντικό και να είναι χειρό μήνυμα για το τι θέλουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και επιτήρηση από πλευρά του Κοινοβουλίου σε όλη την διαδικασία. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας μόνιμος εισηγητής πολιτική συνοχή, όχι μόνο στο ιστορικό της πολιτικής ε, ανάπτυξης, αλλά και σε όλους τους τομείς πολιτικής είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Στην εμπορική πολιτική, στη γεωργική πολιτική, πάντα πρέπει να τι ελέγχουμε τις πολιτικές αυτές για να μην προκαλείται τελικά ζημιά. Και αυτό θα πρέπει να αναφερθεί εδώ πέρα. Και η καλή διακυβέρνηση. Μεγάλη πρόκληση. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ξεχωριστό κεφάλαιο για το θέμα αυτό. Πιστεύω όμως, όπως σας είπα, ότι αλληλεπικαλύπτονται πολλές από τις ε, τροπολογίες και ότι θα είναι πολύ καλό τελικά το κείμενο της έκθεσης που θα Thank you. Ευχαριστώ. Η κυρία Χιμένεθ Μπεσερίλ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ήθελα να σας πω ότι ως εισηγήτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Γυναικών Χαίρομαι που ο εισηγητής, ο κύριος Στιέρ, ε, επεσήμανε τον κεντρικό ρόλο των γυναικών στο θεματολόγιο του πλαισίου για την ανάπτυξη. Και θεωρούμε ότι η πρόταση που κάναμε από πλευράς Επιτροπής Γυναικών θα εμπλουτίσει την έκθεση. Θεωρώ ότι το θέμα των γυναικών είναι εγκάρσια και άπτονται όλων των θεμάτων που έθιξε στην έκθεση του εισηγητής. Για να σας πω κάποια επιγραμματικά, παιδεία, η συμμετοχή των γυναικών στην τοπική οικονομία, στην λήψη αποφάσεων, στη μετανάστευση, ε, στην ε, διατροφή και φυσικά η βία και η ασφάλεια. Κατά την άποψή μας, ε, εγώ τόνισα πάρα πολύ το θέμα της βίας κατά των γυναικών ε, σε περιπτώσεις πολέμου, όπως βλέπουμε σε πολλές από αυτές τις αναπτυσσόμενες χώρες και θεωρώ ότι αυτό είναι ζωτική σημασία προκειμένου να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών που πολλές φορές αποτελούν όπλο ε, ε, η βία χρησιμοποιείται ως όπλο του πολέμου και η, καταχρ... Ε, και καταπίεση επίσης. Και θα ήθελα να συγχαρώ και τον εισηγητή για την έκθεσή του, διότι είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη, αλλά και πλήρης η έκθεσή του. Ε, οι βασικοί στόχοι της ανάπτυξης που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περιλαμβάνονται στην έκθεση αυτά και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να μιλάμε με μία ισχυρή φωνή για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσει. Επίσης χαίρομαι, ε, διότι αναφέρεστε και συγκεκριμένα στα ανθρώπινα δικαιώματα, διότι θεωρώ ότι αποτελούν πηγή έμπνευση όλη τη έκθεση. Αλλά θεωρώ ότι αυτή η έμπνευση θα πρέπει να μεταφραστεί και σε πολιτική βούλευση, βούληση προκειμένου να ενισχύσουμε τι δεσμεύσει μα ω Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Madam Hautala. Yeah, thank you. Ευχαριστώ. Η κυρία Μαρία Φρασείδη τη θέση της ομάδας μας και θα ήθελα να πω ότι ο εισηγητής ήταν πολύ ανοιχτός, ε, πολύ ανοιχτός στο να βρούμε μια συνενετική έκθεση, ένα συνενετικό κείμενο. Είμαστε πολύ κοντά νομίζω σε αυτό και πρέπει να σεβαστούμε και το χρονοδιάγραμμα. Νομίζω ότι η πραγματική στρατηγική ερώτηση εδώ είναι μία που θίξατε και πολλοί από εσά, δηλαδή τι να πούμε για τον αριθμό των στόχων. όταν η διακυβερνητική διαδικασία θα ξεκινήσει του χρόνου, νομίζω ότι θα υπάρχουν πολλές απόπειρε να μειωθεί ο αριθμό των στόχων εξ ονόματο μιας απλούστευσης. Αλλά στην πραγματικότητα υπάρχουν ε, πολύ ισχυρά πολιτικά κίνητρα για να μειωθούν κάποιοι στόχοι σε σχέση με τα δικαιώματα των γυναικών, παραδείγματο χάρη. Και χαίρομαι που ο εισηγητή ε, είναι υπέρ του να δοθεί έμφαση στην προσέγγιση που βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Νομίζω λοιπόν ότι η διατύπωση πρέπει να είναι πολύ καλή, γιατί πολλοί θα χρησιμοποιήσουν ε, τα επιχειρήματά μας αν θέλουν να πούν ότι είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο. Και Αναφέρθηκε και ο συνάδελφο ε, στο θέμα τη αναδιάρθρωση των στόχων. Είναι καλή ιδέα, αλλά νομίζω ότι ίσω αυτό θα πρέπει να το δούμε αργότερα. Φυσικά αυτό θα το αποφασίσουν οι σκιώδει. Πιστεύω λοιπόν όντω ότι όταν θα λάβουμε και την συνθετική έκθεση του Γενικού Γραμματέα, νομίζω ότι θα είναι, ελπίζω να είναι τόσο φιλόδοξη όσο και έκθεση της Ενωτής Εργασίας. Αλλά φυσικά δεν υπάρχει εγγύηση. Μάλλον θα πρέπει να δώσουμε αυτόν τον αγώνα όταν θα μπούμε στη διακυβερνητική διαδικασία. Α μην κάνουμε πιο δύσκολο αυτόν τον αγώνα. Ο κύριο Γκερερό Σαλόμεφ. Ναι, πολύ σύντομα, γιατί εγώ είμαι πολύ επιθαρχημένο. Ε, σέβομαι τη θέση τη ομάδα μου, που είναι εξέφραση τη ηγετρία. Όμω έχω θέσει πέντε τροπολογίες που βασικά συμπίπτουν με την εξή εστίαση, δηλαδή να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυ την κατάσταση των αποτυχημένων κρατών και να υποστηρίζουμε το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη διακυβέρνηση. Αλλά υπάρχει κάτι που θέλω να υπογραμμίσω και να ζητήσω κατανόηση και υποστήριξη από όλε τι ομάδε και είναι εξή ε, τροπολογία, ότι υπάρχει μια εγκάρσια αντίληψη που να προστατεύει ε, τους ανθρώπους που έχουν κάποια αναπηρία. Και αυτό έχει να κάνει μια προσέγγιση που αφορά και το περιβάλλον και την καταπολέμηση της όχιας κτλ. Δεν βλέπω να ζητά άλλο το λόγο, όμως κάποιος από την Κομισιόν θέλει να πει κάτι συντομία, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να πω ότι καλωσορίζουμε την έκθεση αυτή. Θεωρούμε ότι έρχεται σε καλά τάλληλη γλωσσική χρονική στιγμή, γιατί θα έχουμε και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου το Δεκέμβριο και επίσης και την ε, συνθετική έκθεση του Γενικού Γραμματέα. Υπάρχει μεγάλη σύγκληση μεταξύ των ιδεών της έκθεσης και αυτών που πρόθεσε η Κομισιόν στις δύο ανακοινώσει της ε, τον Ιούνιο. Ως παράδειγμα θα αναφέρω την εστίαση στη φτώχεια, την έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα και για θέματα φύλου. Επίσης, τη σημασία που προσδίδουμε όλοι στο ρόλο της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα, σε αυτό το πλαίσιο, τη σημασία των ανισοτήτων, το γεγονός ε, ότι ο στόχος υπαριθμών 16 για θέματα ασφάλειας ε, και διακυβέρνησης είναι κάτι πολύ σημαντικό, θέλουμε να τον προωθήσουμε και να αποφύγουμε να αποδυναμωθεί στην υπόλοιπη διαδικασία. Η σημασία της επιστημιστικής ασφάλειας και επίσης το θέμα της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής. Πιστεύουμε ότι αυτό θα είναι κεντρικό για την εφαρμογή αυτού του νέου Υπάρχουν κάποια δύσκολα ζητήματα μπροστά μας. Ε, ανέφερε ένα ο ίδιος ο εισηγητής, ανέφερε το θέμα της ε, καθολικότητας, ε, του καθολικού χαρακτήρα και πώς αυτό θα μεταφραστεί εσωτερικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης αυτό συνδέεται και με μέσα εφαρμογής γενικότερα. Όλοι κατανοούμε ότι χρειαζόμαστε μια νέα σχέση, αλλά υπάρχουν και αναδυόμενες χώρες που θα πρέπει να κατανοήσουν ότι έχουν ένα σημαντικό και αυξανόμενο ρόλο στην εφαρμογή αυτής της στρατηγικής και εντός αλλά και εκτός των χωρών τους. Και επίσης και οι εγχώριες πολιτικές θα πρέπει να τονιστούν. Για το μέλλον να σας πω ότι κάποιοι από τους βουλευτές και ο ηγητής αναφέρθηκαν ε, στον αριθμό των στόχων, δηλαδή το γεγονός ότι έχουμε 17 στόχους. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι σε έναν ιδανικό κόσμο 17 προτεραιότητες είναι πάρα πολλές. Μόλις όμως ε, μετέβη στη Νέα Υόρκη και συνομίλησα με στενούς ε, συνεργάτες του Γενικού Γραμματέα, και μίλησα και με βασικούς παίκτες, Βραζιλία, Ινδία, ΙΠΑ και νομίζω ότι υπάρχει μια ολένα και αυξανόμενη συντήρηση ότι ο Γενικός Γραμματέας δεν θα αμφισβητήσει τον κατάλογο των 17 στόχων και πιθανότητα θα περιοριστεί στο να κάνει κάποια ομαδοποίηση για λόγους παρουσίασης για να υπάρχει ένα πλαίσιο που θα είναι πιο εύκολο να το γνωστοποιήσουμε. Αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει και πολύ μεγάλη όρεξη να ξανανοίξει η συζήτηση επί τη ουσία στη Νέα Υόρκη. Και συμφωνώ και με του προλύσαντε ότι αν γίνει κάτι τέτοιο, πιθανότατα κάποιοι από του στόχου που είναι πολύ σημαντικοί για μα θα τεθούν σε κίνδυνο. Να κλείσω επαναλαμβάνοντας το εξή, υπόθηκε και από κάποιου βουλευτέ, ότι χρειαζόμαστε μια ισχυρή θέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τι διακυβερνητικέ διαπραγματεύσει που θα ξεκινήσουν τον Ιανουάριο και ελπίζουμε ότι όλοι μαζί, η Κομισιόν, Συμβούλιο, Κοινοβούλιο, θα μπορέσουμε να παρουσιάσουμε μια φιλόδοξη θέση που θα την υπερασπίσουμε και τους επόμενους μήνες. Να πω και κάτι για την κλιματική αλλαγή. Αναφέρεται βασικά στην έκθεση τη Ομάδα Εργασία, αναφέρθηκε και από του προλαλήσαντε. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτό το σημαντικό θέμα θα καλύπτεται παρκώ στο νέο πλαίσιο και ότι υπάρχει στην στρατηγική πρέπει να είναι συνεκτικό και θα πρέπει να υποστηρίζει και τις διαπραγματεύσεις περί κλιματικής αλλαγής ε, που θα φτάσουν ε, σε μια κορύφωση το επόμενο καλοκαίρι. Ευχαριστώ πολύ. Θα ψηφίσουμε για την κλιματική αλλαγή στη συνέχεια και ελπίζω να υπάρχει συνοχή μεταξύ των διαφόρων θέσεων. Κύριε Στήρ, θέλετε να απαντήσετε σε κάποιες από τις παρατηρήσεις που έγιναν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συνεισέφεραν σε αυτή τη συζήτηση και και όσους ε, ε, έκαναν και τροπολογίες για να σταθώ εν συντομία σε λίγα από τα θέματα τα οποία αναφέρθηκαν εδώ. Αναφερθήκατε στην ε, παγκόσμια εταιρική σχέση, το γεγονός ότι θα πρέπει να ενισχυθεί αυτό και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που σίγουρα θα λάβουμε υπόψη και θα ε, κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση στους συμβιβασμού. Βεβαίως υπάρχει και το θέμα της ανισότητας. Ε. Ανισότητας όλων των μορφών, όπως είπατε και εσείς, πρόκειται για ένα ακόμα ζήτημα το οποίο θα αντανακλάται στις συμβαστικές προτάσεις. Ε, θα το συζητήσουμε βέβαια με λεπτομέρεια στη ε, σύσκεψη των ε, συντονιστών, αλλά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει και δεσμευόμαστε να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. προς τον ιδιωτικό τομέα, νομίζω ότι η στάση μας είναι αντί να παραβλέπουμε το γεγονός ότι ο ιδιωτικός τομέας σίγουρα συνεισφέρει ιδιαίτερα και μάλιστα είχε και μεγάλη παρουσία και έχει διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη στόχων. Ε, καλό είναι να υπάρχει ο ιδιωτικός τομέας και να τονίσουμε ότι ο ρόλος που διαδραματίζει ο ιδιωτικός τομέας θα πρέπει να βοηθά στους στόχους της ανάπτυξης που έχουμε. Αντί λοιπόν να παραβλέπουμε το ζήτημα, θεωρώ ότι καλύτερα θα ήταν να αντανακλάται αυτό κάπως το κείμενο. Και βεβαίως ένας ιδιωτικός κλάδος που δεσμεύεται για τους στόχους αυτούς είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να αναζητούμε. Ο Πάβο, ο αντιπρόεδρος, σαφέστατα έκανε διάκριση. Δεν είναι θέμα μείωσης, αλλά αναδιοργάνωσης. Και όντως βρήκαμε και μαζί κάναμε και μία τροπολογία η οποία τρόπον τεινά μας δείχνει την άγουσα που θα έπρεπε να ακολουθήσουμε χωρίς να είμαστε πολύ ε, περιορισμένη στην εντολή ε, του Κοινοβουλίου για τη διαπραγματευτική διαδικασία. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο σίγουρα μπορούμε να επιτύχουμε. Αλλά και πάλι αυτή τη στιγμή ε, δεν θα ήθελα ε, να υπάρξει καμία παρανόηση, να μην θεωρηθεί ότι εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι λέμε ότι αυτοί είναι η κατάλληλη οδό, θα πρέπει να τα ομαδοποιήσουμε όλα και δεν υπάρχει άλλη διέξοδο. αλλά μπορούμε να κάνουμε μια πρόταση ακριβώ με τον τρόπο με τον οποίο διατυπώθηκε και η τροπολογία στην κυρία Λόλα Σάλτσες. Η ε, ένδια όχι μόνο βάσει του εισοδήματο. Ε, Βεβαίω, αυτή είναι μία από τις δεσμεύσεις που θέλουμε να συμπεριλάβουμε και θα συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση και θα το δούμε σίγουρα και την Τετάρτη. Αλλά νομίζω ότι αυτή η άποψη ε, σίγουρα δεν θα έχει πρόβλημα. Ίσως να μην ήταν τόσο σαφές όσον αφορά το όριο των λέξεων που υπάρχει στην πρώτη εκδοχή του κειμένου, αλλά στις συμβαστικές λύσεις σίγουρα θα τα ανακλάτε αυτό στην κυρία Χόιμπαχ, η χρηστή διακυβέρνηση, πέραν των όσων είπατε για τη σημασία της ε, κλιματικής αλλαγής, νομίζω ότι η χρηστή διακυβέρνηση θα πρέπει να επισημάνεται και ως παγκόσμια χρηστή διακυβέρνηση. Ε, πολλές φορές αναφερόμαστε στο θέμα αυτό και λέμε και το εξής, χρειάζονται δύο για να τα καταφέρουν. χρειαζόμαστε και από τις δύο πλευρές ε, χρηστή διακυβέρνηση, όχι μόνο στις αναπτυσσόμενες χώρες, διότι συζητούμε και το ρόλο των αναπτυγμένων χωρών εδώ. Και εδώ έρχεται και ο καθολικός χαρακτήρας του νέου πλαισίου. Η χρηστή διακυβέρνηση στην οποία αναφερόμαστε είναι παγκόσμια χρηστή διακυβέρνηση και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το επισημάνουμε. Ο στόχο του 0,7 είναι στι συμβιβαστικές προτάσει. Υπήρχαν πολλέ τροπολογίε προ αυτή την κατεύθυνση, Επομένω πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι και δεν νομίζω ότι θα δημιουργηθεί θέμα. Ω προ ένα μόνιμο εισηγητή, νομίζω ότι είναι έστοχη η παρατήρησή σα. Δεν ξέρω αν αυτό είναι το κατάλληλο έγγραφο για να, γίνει, να ληφθεί συγκεκριμένη απόφαση, διότι αυτή η απόφαση θα πρέπει να ληφθεί από την Επιτροπή. Δεν ε, χρειαζόμαστε όλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποφασίσει κάτι το οποίο μπορούμε να αποφασίσουμε εμεί σε επίπεδο Επιτροπή μας. Αυτή είναι η απόψή μου. Ε, είμαι πολύ ειλικρινής και ανοιχτός ως προς την πρόταση αυτή. Ε, πολύ λογική πρόταση. Αναφερθήκατε, κυρία Χιμένες Μπεχερίλ, στην γνωμοδότηση τη Επιτροπής Γυναικών και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ο ρόλος των γυναικών και ε, κατά πόσον μπορεί να είναι και ενεργός. Ε, δεν ξέρω αν βοηθά μόνο στην ε, πάταξη των διακρίσεων ε, και στα περιστατικά βίας κατά των γυναικών, αλλά υπάρχει και η διαδικασία λήψης απόφασης και νομίζω ότι θα πρέπει να επισημάνουμε και το ρόλο των γυναικών σε αυτή την έκθεση και σε αυτό το τομέα. Στην κυρία Χάουτουλα για τη συνένεση. Σας ευχαριστώ που είστε αισιόδοξοι. Ε, τον, τον αισιοδοξία σας και ελπίζω ότι την Δετάρτη θα έχουμε συνένεση για τα αποτυχημένα κράτη, να σας πω ότι και αυτό ε, περιλαμβάνεται στο κείμενο και θα προσπαθήσουμε να συμπεριλάβουμε και το θέμα των ατόμων με αναπηρία. Όσον αφορά τον αριθμό των στόχων, και με αυτό θα κλείσω, κατά πόσον η συζήτηση θα κινηθεί ε, ως προς την ομαδοποίηση ή στο έγγραφο του Γενικού Γραμματέα πώς θα πάνε οι διακυβερνητικές διαπραγματεύσεις, πρόκειται για ένα θέμα το οποίο τους άλλους μας αφορά. Νομίζω ότι θα πρέπει να πούμε την άποψή μας και γι' αυτό. Δεν θα πρέπει ε, να μην είναι σαφής η άποψή μας. Και νομίζω ότι θα έπρεπε να λέμε ότι ναι, είμαστε ανοιχτοί σε απλούστευση και αναδιοργάνωση και σε ιδανικές συνθήκες ε, ο, ο πρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπε ακόμα και να μειώσουμε. Ε, εμείς δεν είμαστε αντίθετοι σε αυτό. Αυτό το οποίο δεν θα θέλαμε όμως σε καμία περίπτωση είναι να είναι αυτό εις βάρος της προσέγγισης με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι σαφές ως μήνυμα. Και αν μόνο ε, το μήνυμα τελικώς περάσει. Εμείς συζητούμε εδώ τη φιλοδοξία που πρέπει να έχουμε. Αν λοιπόν είναι αυτό το βασικό μήνυμα το οποίο θα ε, απορρέει από αυτή την έκθεση, θεωρώ ότι ούτω ή άλλω θα έχουμε επιτύχει ένα πάρα πολύ σημαντικό στόχο για το έγγραφο αυτό. Βεβαίω δεν λέω ότι αυτό είναι το μόνο μήνυμα, αλλά θεωρώ ότι είναι σημαντικό να είναι τουλάχιστον αυτό το μήνυμα σαφή. Σα ευχαριστώ πολύ για τη συνεισφορά σα. Uh, Σας ευχαριστώ κύριε Στήρη. Θα ήθελα να πω στους συναδέλφους, ξέρω ότι οι σκιώδες συναντιόνται με τον εισηγητή αυτή την εβδομάδα. Ε, προσπαθήστε να βρείτε συμβιβασμού γιατί πρέπει να ψηφίσουμε την άλλη εβδομάδα εάν θέλουμε να επηρεάσουμε την άποψη του, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Κάντε λοιπόν ό,τι μπορείτε. Κλείστε συμβιβασμού για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε μέχρι την άλλη εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα Έχουμε καθυστερήσει, θα κάνουμε την ε, ψηφοφορία για την κλιματική αλλαγή. 10 λεπτά θα πάρει. Αν ε, έχετε την καλοσύνη να δείξετε υπονομή, να ξεκινήσουμε λοιπόν κατευθείαν την ψηφοφορία. Έχετε τις ε, κάρτες σας έτοιμες, συνάδελφοι. Okay. Okay, colleagues. Okay, I, you need, you need to... Okay, colleagues. Μάλιστα λοιπόν συνάδελφοι, όπως ξέρετε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα ανέκρινε τα συμπεράσματα για την αλλαγή του κλίματος και κάλεσε την έγκριση των στόχων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη μείωση του διοξιδίου του άνθρακα και θα ψηφίσουμε λοιπόν ε, το ψήφισμα που θα αποσταλεί στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και μετά θα ε, ψηφιστεί στη δεύτερη ε, ολομέλεια της δεύτερη σύνοδο του Νοεμβρίου και θα ψηφιστεί τελικά πριν από την κόπ του Δεκεμβρίου στη Λίμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για αυτά που συζητήσαμε σε ατεφάτες στόχους ε, της χιλιετίας και το θέμα της δικαιοσύνης σε παγκόσμιο επίπεδο και για θέματα κλίματος. Να περάσουμε λοιπόν κατευθείαν στην πρώτη ψηφοφορία. Τροπολογία 30. Υπέρ. Υπέρ της τροπολογίας 30 παρακαλώ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 29. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία υπαριθμών 2. Υπέρ. Της προφορικής τροπολογίας. Κατά. Άποχες. Να το ελέγξουμε. Ελέγχουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά την ε, προφορική τροπολογία. A check on amendment, all amendment two. Προφορική τροπολογία 2. Έναρξη ψηφοφορία. So EFTD... Από το EFTD έχουμε δύο άτομα παραπάνω που ψηφίζουν. Δύο ψήφοι παραπάνω για την ομάδα του EFTD. Τέσσερις ψηφίζουν. Μα τι γίνεται. Okay, hang Συνάδελφοι, μισό λεπτό. Κάντε λίγο υπομονή γιατί κάτι δεν πάει καλά με το σύστημα. Να κάνουμε έναν έλεγχο, γιατί δύο μόνοι είσαστε. Πώς λοιπόν περισσεύουν δύο. Πώς έχουμε δύο ψήφους υπεράριθμες. Να περιμένουμε λίγο. Should we check, full check? Hmm? we They're checking the system. do show. Ελέγχουμε το σύστημα. Ας κοιτάξουμε για σηκώστε τα χέρια για την προφορική τροπολογία 2. Σηκώστε τα χέρια. Όσοι είναι υπέρ της προφορικής τροπολογίας 2. Okay, Κατά τώρα. Abstentions. Αποχές εγκρίνεται. Άρα ελπίζω την επόμενη φορά να, πάνε καλύτερα τα πράγματα. Να μην έχετε δεκτυμένο κανένα δίδυμο μόνο ψηφίσετε. Okay. Compromise Τροπολογία συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 33. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 3. Υπέρ. Δεν τη θέλει λοιπόν η δική σα η ομάδα, άρα δεν μπορούμε να την υπερψηφίσουμε. Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε την προφορική τροπολογία, συμβαστική τροπολογία 5. Λοιπόν, υπέρ. Συμβαστική τροπολογία 5, υπέρ. Κατά. άποχέ. Εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην τροπολογία τη 40, στα μέσα της σελίδας. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 41. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 42. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 43. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Συμβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 48. Τώρα περνάμε στη 48. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7. Στη σελίδα 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 49 πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 50. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 52 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 53 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Την ψηφίζουμε την 55. 55, ναι, ναι, ναι. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Έγκρινεται. Η 56 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. 57 υπέρ. Κατά. Άποχες. Έγκρινεται. Α, συγγνώμη, απορρίπτεται, λέει η Πρόεδρος. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 60 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Και έτσι περνάμε την 59, Τώρα λοιπόν τι ψηφίζουμε. 61. 61. Τροπολογία 61. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 63. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 64. Υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. 70. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. Στις συντελεγικές σκέψεις τώρα περνάμε. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 2. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 9. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 10. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 11. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Και περνάμε στην 19. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 23. Υπέρ. Κάτα. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τελική ψηφοφορία τώρα ηλεκτρονικά. Έναρξη της ψηφοφορίας. Close the vote. Πέρας ψηφοφορίας. Και τα αποτελέσματα λοιπόν της ψηφοφορίας είναι ως εξής 19 ψήφοι υπέρ, 3 κατά, μία αποχή. Σας ευχαριστώ λοιπόν και όσοι συμμετείχατε στην ψηφοφορία και στους κοιόδης. Και γρήγορα, γρήγορα να περάσουμε στο τελευταίο θέμα της σημερινής διάταξης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα διακόψουμε δύο λεπτάκια για να έρθουν οι ομιλητές μας εδώ στο Προεδρείο. Ε, διάλειμμα λοιπόν για να αλλάξουμε θέση.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 Okay, colleagues, if everyone can settle down now. Παρακαλώ καθίστε συνάδελφοι γιατί ούτως ή άλλως έχουμε καθυστερήσει και το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα ήθελα λοιπόν να καθίσετε όλοι για να ξεκινήσουμε με το σημείο 10, ανταλλαγή απόψεων για την κρίση του έμπολα. Βεβαίως δεν είναι η πρώτη φορά που συζητάμε το ζήτημα, ούτε εδώ στην Επιτροπή ούτε στην Ολομέλεια, αλλά όπως θα γνωρίζετε από τα νέα από τις ειδήσει, η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή και σήμερα το σκεπτικό μας είναι ε, ότι επειδή Στι αρχές Σεπτεμβρίου μιλήσαμε τελευταία φορά εδώ στην Επιτροπή μας για το θέμα. Θα θέλαμε να δούμε τι γίνεται με τη βοήθεια επιτόπου, αν φτάνει η ανθρωπιστική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι έχει να μας πει ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ, τι θέματα θεωρούν ότι προχωρούν, αν έχουμε καταφέρει να έχουμε πρόσβαση μέσω της ανθρωπιστικής μας βοήθεια. Την προηγούμενη εβδομάδα το συζήτησαν το θέμα και αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και λήφθηκε απόφαση ο Επίτροπος Στυλιανίδης να είναι ο υπεύθυνο ε, επιτετραμένος του έμπολα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πάει στη Δυτική Αφρική τις επόμενες εβδομάδες και φαντάζομαι ότι θα έχουμε νεότερα από τον ίδιο μόλις επιστρέψει από την αποστολή του στην Αφρική. Σήμερα όμως πρώτα θα, μιλήσει, θα μιλήσουν ο πρεσβευτής ε, της Γουινέας, ο κύριος Ουας ο πρεσβευτής της Δημοκρατίας Γουινέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρόεδρος Επιτροπής Περισβευτών και στη συνέχεια ο κύριος Μοχάμεντ Μουμούνι, Γενικός Γραμματέας της Ομάδας Κρατών ΑΚΕ. Θα μας πούν ε, για τα συμπεράσματα ενός ειδικού συμποσίου για την κρίση του έμπολα που έγινε στην έδρα της ΑΚΕ στις Βρυξέλλες πριν από λίγες μέρες και θα μας πούν και τα νεότερα από τις χώρες που έχουν πληγεί. Επίσης ε, θα συζητήσουμε και τα μακροπρόθεσμα ζητήματα τα οποία εφήχθησαν και όπως γνωρίζετε συμφωνήσαμε και στην Επιτροπή μας να συντάξουμε μια έκθεση για τα διδάγματα μακροπρόθεσμα από τον ε, έμπολα, ώστε να μην επαναληφθεί ε, το ζήτημα. Έχουμε ορίσει και εισηγητή. Και αφού ακούσουμε λοιπόν τους δύο προσκεκλισμένους μεσομελητές από την ΑΚΕ, θα ακούσουμε και τον κύριο Ζαν Λουί Ντεμπρουγέ, Διευθυντή Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας στη Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ, για να ακούσουμε και την οπτική γωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε επίσης και δύο εκπροσώπους από τη Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης που θα μιλήσουν και αυτοί στο τέλος. Να δώσω λοιπόν πρώτα το λόγο στον κύριο Σίλα για 8 λεπτά για να μας πει δύο λόγια για την κατάσταση στη Γουινέα και ε, να μας πει αν βελτιώνεται η κατάσταση επιτόπου και κατά πόσον κύριε Πρέσβη αν θέλετε να κάνουμε και εμείς κάτι προκειμένου να πιέσουμε ώστε να υπάρξει ε, βοήθεια για τη χώρα σας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω εξ ονόματος ε, της Επιτροπής Πρεσβευτών, της οποίας προεδρεύω επί του παρόντος, για την πρόσκληση εδώ για δεύτερη φορά ε, είχα έρθει και στις 23 Σεπτεμβρίου του 2014 με τη συνάδελφο από τη Σιέρα Λεώνα για να μιλήσουμε για τον έμπολα και επομένω, για άλλη μια φορά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την πρόσκληση. Πράγματι, από τις 23 Σεπτεμβρίου οι χώρε ΑΚΕ αποφάσισαν να διοργανώσουν μαζί με τις ε, ε, τρεις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο, ε, την Σιέρα Λεόνε τη Γουινέα και τη Λιβερία, ένα συμπόζιο το οποίο έγινε στις 17 Οκτωβρίου εδώ στην έδρα των χωρών ΑΚΕ. Και το συμπόσιο αυτό... Ε, διοργανώθηκε με πολύ αποτελεσματικό τρόπο και θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμή εδώ στην κυρία Ρέμοντ, τη Γενική Γραμματέα των Χορονακέ, η οποία διοργάνωσε με τέτοια αποτελεσματικότητα το συμπόσιο σε τόσο σύντομο διά, ε, διάστημα. Είχαμε περίπου 185 ε, συμμετέχοντες. Έγινε το συμπόσιο αυτό ε, και είχαμε συμμετοχή από όλους όσους έχουν πληγεί από τον έμπολα. Ε, είχαμε και ε, έναν ε, ερευνητή από τη Γουινέα που κάνει έρευνες στη Γουινέα όχι μόνο για τον έμπολα αλλά και για το AIDS και για άλλες ασθένειες. Και αυτό ήταν για να αποδείξουμε ότι δεν υπάρχει μόνο επιστημονική έρευνα από ε, ευρωπαϊκή και αμερικανική πλευρά, αλλά και στην Αφρική έχουμε μεγάλους ερευνητές, τις χώρες οι οποίες πλήττονται, που ασχολούνται ε, στο φαρμακευτικό τομέα ε, με τα φαρμακευτικά φυτά ε, και προσπαθούν να βρουν εάν μπορούμε να βρούμε όχι ίσως ένα εμβόλιο αλλά κάποια φάρμακα τα οποία θα μας βοηθήσουν να φροντίσουμε τους ανθρώπους που έχουν έμπολα. Ε, ήρθε λοιπόν ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος μας εξήγησε τον ιό του έμπολα, τα αποτελέσματα της έρευνας και τη συνεργασία που υπάρχει. Δεν γίνονται ε, μόνο ε, έρευνες ε, αυτόνομες, αλλά υπάρχει συνεργασία με ερευνητικά κέντρα σε τροπικές ασθένειες, όπως για παράδειγμα το κέντρο στην Αμβέρσα που είναι πολύ γνωστό, υπάρχει ένα κέντρο στη Γερμανία πολύ γνωστό για ασθένειες αυτής της μορφής και μας έδωσε και κάποιες ελπίδες ο άνθρωπος αυτός, διότι μας είπε ότι ότι ε, δεν γίνεται έρευνα μόνο στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στην Αφρική υπάρχουν μεγάλοι ερευνητές οι οποίοι ήδη έχουν εντοπίσει κάποια φάρμακα τα οποία φαίνεται ότι μπορούν να βοηθήσουν. Ο συγκεκριμένος ε, άνθρωπος ε, έχει ε, αναπτύξει ένα φάρμακο το οποίο αναγνωρίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και έχει προταθεί στη Γενέβη για να δούμε κατά πόσον μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το μόριο το οποίο θα μπορούσε ίσως να καταπολεμήσει τον έμπορο. Αυτό ήταν λοιπόν ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα του συμποσίου, ε, τα αποτελέσματα της έρευνας. Υπήρχαν επίσης και κάποιοι Βέλγοι ε, ερευνητέ, οι οποίοι εξήγησαν τι γίνεται στο Βέλγιο, έρευνα για εμβόλιο αλλά και φάρμακα. Ξέρετε ότι ο ιός του έμπολα ε, έχει ανακαλυφθεί από έναν μεγάλο Βέλγο ερευνητή, το 1976. Και επίσης ε, ε, μας μίλησαν και για την κατάσταση επιτόπου και εκεί φυσικά είχαμε την τύχη να έχουμε τους γιατρούς χωρίς σύνορα, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τη UNICEF ε, τον ε, Διεθνή Ερυθρό Σταυρό που ε, έκαναν παρουσιάσεις για την εμπειρία τους επιτόπου στις τρεις χώρες. Και θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι μέχρι σήμερα βρισκόμαστε πλέον στους 5.000 νεκρούς. 5.000 νεκρούς στις τρεις χώρες και περίπου 10.000 ανθρώπους που έχουν νοσήσει. Το ποσοστό θνησιμότητας ποικίλει από 50 μέχρι και 100% σε κάποιες περιοχές. Όπω μα είπε ο Υπουργό Υγεία τη Λιβερίας και οι τρει αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων που ήταν εκεί, ε, το ε, έμπολα, ο έμπολα είναι για μα σαν ένα δαδί το οποίο αρχίζει να κάνει πολύ μεγάλες, προκαλεί πολύ μεγάλε πυρκαγιέ. Επομένω θέλουμε να δράσουμε αποτελεσματικά επιτόπου προκειμένου να βελτιώσουμε τα συστήματα υγεία μα, τα οποία φυσικά πάσχουν στις χώρες μας. Ε, δεύτερον, θα πρέπει να ενημερώσουμε του ιατρού μα και του νοσοκόμου μα για την θεραπεία του έμπολα και τρίτο, κατεπηγόντως, κατάλληλος εξοπλισμός. Κυρία Πρόεδρε, με ρωτήσατε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς εδώ και τώρα. Η έκκλησή μου λοιπόν προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι, αφού καταρχάς ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, όλα τα τμήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την Επιτροπή σας, αλλά και όλους όσοι κινητοποιήθηκαν. Η κινητοποίηση ήρθε με ε, κάπως καθυστερημένα, αλλά δεν ήρθε κατόπιν εορτής. Και ελπίζουμε ότι με αυτή τη μεγάλη κινητοποίηση θα υπάρξει μια πολύ ε, γρήγορη ανταπόκριση στον πυρετό αυτό. Και επίσης ε, ε, όταν συζητήσαμε και τους εταίρους μας από τη Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟΥ ε, χρειαζόμαστε μία άμεση βοήθεια στη χώρα μας. Συναντηθήκαμε στη Νέα Υόρκη και με την Παγκόσμια Τράπεζα η οποία έκανε και μία πολύ μεγάλη διάσκεψη. Στα Ηνωμένα Έθνη το Σεπτέμβριο υπήρξαν πολλές δεσμεύσεις. Βρισκόμαστε στα 2 με 3 δισεκατομμύρια δεσμεύσεων αλλά γνωρίζετε ότι μεταξύ της δέσμευσης, της εκταμίευσης και της υλοποίησης επιτόπου υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση. Σας ευχαριστούμε για δεσμεύσει στη Νέα Υόρκη, αλλά χρειαζόμαστε άμεσε ταχύτατες αποτελεσματικέ ενισχύσει αυτή τη στιγμή και χαιρόμαστε που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, Ένωση αποφάσισε να έχει έναν υπεύθυνο για τον έμπολα για να συντονίζει όλε τις εργασίες, γιατί ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ακριβώ αυτό ο συντονισμό τη βοήθεια. Ε, θυμάστε τι έγινε στο σεισμό στην ΑΕΤ. Υπήρξαν όλε αυτέ οι υποσχέσει για την ΑΕΤ και μετά, επειδή ακριβώ δεν υπήρξε συντονισμό, ακόμα και σήμερα δεν έχουν επιληθεί τα πολύ σοβαρά προβλήματα τα οποία προέκυψαν από αυτό το σεισμό. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε αυτά τα προβλήματα, διότι και στη Γουινέα και στη Σιέρα Λεόνε και στη Λιβερία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις ευρωπαϊκές χώρες που μας βοηθούν. Είναι εδώ και η Κίνα, η Ρωσία, η Κούβα, πολλές χώρες μας βοηθούν. Θα πρέπει να υπάρξει κάποιο συντονισμός, διότι δίχως συντονισμό θα χαθεί η βοήθεια, θα, ε, ε, θα είναι διάσπαρτη παντού και θα έχουμε αποτυχία. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι καταφέραμε να μελετήσουμε την οικονομική κατάσταση. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο η θεραπεία της νόσου, αλλά και οι συνέπειες της ε, ε, νόσου στην οικονομία των χωρών μας. Οι χώρες μας ε, αυτή τη στιγμή έχουν οικονομικά προβλήματα λόγω της απομόνωσης, είμαστε στιγματισμένοι, αρκεί κάποιος να πάει σε κάποιο αεροδρόμιο και να δει ότι μόλις εμφανιστεί κάτοχος διαβατηρίου από Νέα Λιβερία και Σιέρα Λοένα, αμέσως ε, υπάρχει το στίγμα. Και επομένω, είπα σε πολλές συναντήσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, χρειαζόμαστε, ε, και είναι και λίγο φιλόδοξες από πλευρό μας, χρειαζόμαστε ένα σχέδιο Μάρσαλ μετά τον έμπολα. Διότι μετά τον έμπολα υπάρχει ανοικοδόμηση των οικονομιών μας. Η γεωργία δεν λειτουργεί πλέον, ο τουρισμό δεν λειτουργεί πλέον, οι επενδύσεις ε, στον τομέα των εξορίξεων έχουν σταματήσει, ε, τα ξενοδοχεία είναι άδεια και η ζωή έγινε πάρα πολύ δύσκολη στις χώρες μας. Υπάρχει λοιπόν η περίοδος μετά τον έμπολα, την οποία θα πρέπει να προετοιμάσουμε και θα πρέπει να μας βοηθήσετε να ανεκοδομήσουμε τις οικονομίες μας. Διότι με την παγκόσμια κινητοποίηση που έχουμε, θεωρώ ότι δεν υπάρχει πλέον αμφιβολία, θα την αντιμετωπίσουμε τον έμπολα. Αλλά από εκεί και πέρα ε, ε χρειαζόμαστε... Ε, και το είπε και ο πρόεδρο τη Λιβερία ότι αυτή τη στιγμή αρχίζει να σταθεροποιείται η κατάσταση. Έχουμε και στοιχεία από τον ΠΟΗ και υπάρχει και μία ψύχωση με τα στατιστικά στοιχεία, αλλά δούμε τι γίνεται επί τόπου. Πραγματικά ε, να πούμε στη διεθνή κοινότητα ότι ε, σιγά σιγά αρχίζουμε να ε, σταθεροποιούμε αυτό τον αιμορραγικό πυρετό και να ε, περιορίζουμε την ασθένεια. Ελπίζουμε ότι όλα τα πειράματα τα οποία έχουν ξεκινήσει θα μας επιτρέψουν να έχουμε ένα εμβόλιο στις αρχές του 2015 και ε, υπάρχουν φάρμακα, υπάρχει μεγάλη εμπειρία αυτή τη στιγμή και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην ίδια την Αφρική και επομένως ότι ελπίζουμε ότι σε μερικούς μήνες θα μπορέσουμε να έχουμε ένα εμβόλιο το οποίο θα μας βοηθήσει αλλά κυρίως φάρμακα τα οποία θα μας επιτρέπουν να θεραπεύσουμε την ασθένεια. Αυτά λοιπόν συνοπτικά για τα όσα συνέβησαν στο συμπόσιο. Το συμπόσιο ολοκληρώθηκε με μία έκκληση και αυτή είναι μία έκκληση προς την Αφρικανική Ένωση και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρία Πρόεδρε, θα θέλαμε την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτή την έκκληση και θα θέλαμε να μας βοηθήσετε να διοργανώσουμε το συντομότερο δυνατόν μια διεθνή διάσκεψη αλληλεγγύη για τον έμπολα εδώ στις Βρυξέλλες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, το έκανε και με την ε, Αφρικανική ε, Ένωση όταν υπήρξε επίθεση των τρομοκρατών στο Μάλι και ελπίζουμε ότι θα υπάρξει μια αντίστοιχη πρωτοβουλία με την ε, Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Επιτροπή της Αφρικανικής Ένωσης ώστε να διοργανώσουμε το συντομότερο δυνατόν μια μεγάλη ε, διάσκεψη για τον έμπολα διότι ο έμπολα πλέον δεν είναι μια ασθένεια της Αφρικής αλλά είναι μια παγκόσμια απειλή και θα πρέπει να απαντήσουμε με παγκόσμια κινητοποίηση εδώ στις Βρυξέλλες και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι όλους και όσους μας βοήθησαν και όσους συνεχίζουν να μας βοηθούν, ιδίω την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και περιμένουμε ότι θα έχουμε και μια επόμενη παγκόσμια ε, ε, σημαντική διάσκεψη για να, και να έρθει και ο νέος απεσταλμένος για να δει τι γίνεται στην, στη χώρα μας επιτόπου. Σε ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. much, us... Σας ευχαριστώ που ήρθατε για να μας ενημερώσετε εκ νέου και ακολουθούμε και παρακολουθούμε θα την έκκληση που κάνετε για τη διεθνή διάσκεψη. Κατόπιν έχουμε καλέσει τον κύριο Μουχάμεντ Μούνι, ο οποίο είναι Γενικό Γραμματέα τη Ομάδα Κρατών ΑΚΕ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι πραγματική ευχαρίστηση για μένα που με καλέσατε να παρευρεθώ εδώ στη συνεδρίαση της Επιτροπής σας και να έχουμε ανταλλαγή απόψεων για την επιδημία του εμπολά στη Δυτική Αφρική. Ευχαριστώ την Πρόεδρο και τα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως ε, περιέγραψε ο Δ. Μακρατσάπα, ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΕ, αυτή η επιδημία του εμπολά στη Δυτική Αφρική είναι οπωσδήποτε η πιο οξία ε, κρίση υγείας των σύγχρονων καιρών αποτελεί απειλή στην παγκόσμια ασφάλεια και υγεία και είναι ένας κινδυνός τεράστιων διαστάσεων ε, για την υγεία, κυρίως στη Λιβερία, στη Σιέρα Λεόνα και στη Γουινέα. Ε, έχουμε ήδη περίπου 5.000 νεκρούς και η νόσος απειλεί περισσότερους. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνετε τι μπορεί να γίνει όταν τα συστήματα υγείας ευάλωτων χωρών δεν είναι αρκετά ανθεκτικά για να αντιμετωπίσουν μια τέτοια κρίση οι ελλείψεις στα συστήματα υγείας ε, των πληγέντων κρατών μας υπενθυμίζουν ότι παρά την πρόοδο που έχει παρατηρηθεί καθολικά και σε πολλές ε, χώρες ΑΚΕ ε, δεν ε, μπορούν πολλές χώρες να πετύχουν τους στόχους της χιλιετίας, δηλαδή μείωση της θνησιμότητας, η καταπολέμηση του AIDS, της ενωσίας και άλλων νόσων πρέπει να αναπτυχθούν έγκαιρες παρεμβάσεις και να εφαρμοστούν από τις χώρες αυτές που δεν μπορούν να πετύχουν τους στόχους κυρίως της ατζέντα μετά το 2015. Πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η ενδυνάμωση των ανθρώπινων πόρων για την υγεία καθώς ε, και να υπάρχει κατάλληλη αναλογία ε, εργαζομένων στην υγεία με τον πληθυσμό. Επιπρόσθετα, η πρόσβαση ε, σε ποιοτικά και φτηνά φάρμακα παραμένει ένα πρόβλημα και ε, αυτό οδηγεί σε μη πλήρη θεραπεία και σε πάρα πολλά έξοδα για τους ασθενείς η ανανεωμένη εταιρική ε, σχέση ε, του ΠΟΕ έχει βελτιώσει ε, την προμήθεια φαρμάκων σε αυτές τις χώρες και φυσικά και το θέμα της, των τροφίμων είναι μεγάλη πρόκληση σε πολλές χώρες και πρέπει να υπάρχουν, υπάρχει συμπερίληψη των δικτών ε, επισητισμού στα προγράμματα. Η Δημοκρατία της Γουινέας με τις άλλες χώρες οργάνωσε το συμπόσιο στο οποίο αναφέρθηκε και ο Δ. Σίλα. Στο συμπόσιο τονίστηκαν τα εξής. Ο αιμορραγικός πυρετός του έμπολα συνεχίζει να ε, εκτίθεται στην Γουινέα, στη Λιβερία και στη Σιέρα Λεόνε συνεχίζει να αναπτύσσεται κάθε τρει εβδομάδες. Η διεθνής κοινότητα και ιδίω οι εθελοντές επιτόπους, τα πληγέντα κράτη, ε, θα πρέπει ε, να ε, δεχτούν την ευγνωμοσύνη μας για τη συνεισφορά τους. Υπάρχει ανάγκη να ενδυναμωθούν τα συστήματα υγείας στα πληγέντα κράτη και πρέπει να υπάρξει και κατάρτιση του ιατρικού προσωπικού. Θα πρέπει η διεθνή κοινότητα να παράσχει βοήθεια στις πληγήσει χώρες, ε, Κυρίω όταν μιλάμε για προσωπικό και για εργαζομένου στην υγεία. Η διεθνή κοινότητα θα πρέπει να αποφύγει να ταξινομήσει όλη την περιοχή της Δικής Αφρικής σε μια μεγάλη χώρα παρία και να περιορίσει την κινητικότητα ε, των ανθρώπων από την περιοχή της Δυτικής Αφρικής. Υπάρχει ανάγκη για κατάλληλο συντονισμό των προσπαθειών απάντησης σε όλα τα επίπεδα για να αποφύγουμε τις επικαλύψεις. Πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους και που, αυτούς που παρέχουν βοήθεια και αυτούς που βοηθούν ε, και να βελτιώσουμε την επιμελητή όχι μόνο στις πληγήσεις χώρες αλλά να λάβουμε και κάποια μέτρα για τις χώρες που είναι σε κίνδυνο. Πρέπει να υποστηρίξουμε τις προσπάθειες ετοιμότητας ε, σε όλες τις γειτονικές χώρες, ε, κυρίως στις χώρες όπου υπάρχουν χερσαία σύνορα. Επίσης, η διακοπή κάποιων εμπορικών πτήσεων στις πληγήσεις χώρες έχει οδηγήσει σε μείωση της δραστηριότητας του τουρισμού και έτσι επιδεινώνεται και το παραγωγικό σύστημα των χωρών. Στο συμπόσιο τονίστηκε ότι τρεις πληγήσεις χώρες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τεράστιες προκλήσεις για να κατεπολεμήσουν τον έμπολα. Καταρχήν, δεν υπάρχουν επαρκείς ομάδες έρευνας ε, ε, λόγω πάρα πολλών ε, θανάτων και κρουσμάτων στην περιοχή και στις πληγήσεις χώρες. Πολλές από τις επαφές χάνονται. Δεύτερον, υπάρχει μια καθυστέρηση στην ταφή ε, των πτωμάτων ε, και μπορεί να εκτίθενται περισσότεροι άνθρωποι σε επίπεδο κοινότητας. Τρίτον, η ε, αξιοπρεπής ε, ταφή και η απολύμαση των σπιτιών. Τέσσερα, υψηλή έκθεση των εργαζομένων στην υγεία ως αποτέλεσμα κάποιων αδύναμων μέτρων προστασίας και μη επαρκών ε, υλικών προστασίας, επίσης άρνηση, έλλειψη εμπιστοσύνης ε, που προκαλείται από παρεξήγηση της αιτία αυτής της νόσου και ε, οδηγεί ε, στο να καταλήγουμε και σε υψηλούς θανάτους στην κοινότητα. Επίσης, παροχή πληροφοριών, πρόληψη του στοίγματος και 7 ε, γίνεται μια απεύθυνση στα παιδιά και στις γυναίκες ε, και αναφέρεται και το θέμα της οικονομικής καταστροφής συνολικά. Αυτές οι προκλήσεις δείχνουν ότι η πολύπλοκη φύση και οι διαδικασίες ε, της διάδοσης της επιδημίας χρειάζονται να υπάρχουν αποτελεσματικά συστήματα υγείας ο έμπολα μας έχει δείξει την ανάγκη που χρειάζεται να υπάρχει πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας για όλους. Επομένως, οι δωριστές καλούνται να χρηματοδοτήσουν το πλήρες φάσμα των δραστηριοτήτων που χρειάζεται για να αναχαιτιστεί η επιδημία του έμπολα. Επειδή τα πληγέντα κράτη ήδη έχουν επιβαρυνθεί από ε, πολύ μεγάλα ποσοστά θνησιμότητας στις μητέρες και τα παιδιά. Έχουμε επίσης επιδημία μηνυγκίτιδας και χολέρας. Ε, έχουμε υποσυτισμό ε, έχουμε νοσοκομεία χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και πολύ περιορισμένους ανθρώπινους σπόρους. Και όλα αυτά αυτά ε, καταλήγουν στο εξή. Το με έθεσε τη σκηνή για να υπάρξει μία διεθνής διάσκεψη για τους δωρητές του έμπολα, για τους δωρητές, λοιπόν, όπως είπα, κυρίως εδώ στις Βρυξέλλες, που ολιστικά να αντιμετωπίσει τον αντίκτυπο της νόσου και στην συγκεκριμένη περιοχή αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Επίσης, αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας για τη συγκράτηση του μερογικού πυρετού το έμπολα στη Δυτική Αφρική, το συμπόσιο επανέλαβε την συνένεση ε, ότι η απάντηση της διεθνούς κοινότητας ε, δεν σέβεται ε, την ταχύτητα, δεν ανταποκρίνεται στην ταχύτητα εξάπλωσης του ιού. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής λοιπόν είναι ο κύριος Ντεμπρουγέρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα μας παρουσιάσει, κύριο Ντεμπράουερ, την ε, δική του άποψη για την τρέχουσα κατάσταση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίε και σας ευχαριστώ που μου καλέσατε εκ νέου εδώ. Είχα... Δεν δεν να σας επενθυμίσω ότι ήταν στη διάθεσή μας οι υπηρεσίες σας για να σας ενημερώσουν και μας δώσατε την ευκαιρία. Εγώ όλη την πρεσμένη εβδομάδα ήμουν στην περιοχή και ήμουν στο Κονακρή, στη Γουινέα, στη Σιέρα Λεόνη και στη Λιβερία και αυτό μου επιτρέπει να έχω μια αρκετά φρέσκια εικόνα ενωμένοντας ε, και τη μεταβάση του κυρίου Στυλιανίδη εκεί. Και σας ευχαριστώ που με καλέσετε εδώ για να σας μεταφέρω τις κυρίες μου εντυπώσεις. Ε, ήταν μια διατομιακή αποστολή όλοι εκπροσωπούνται στην αίθουσα εδώ. Είχαμε συναδέλφου από την Ευρωπαϊκή Περισσία Εξωτερική Δράση, από τη Γενική Διεύθυνση ανάπτυξη και από τη Γενική Διεύθυνση για τη Δημόσια Υγεία. Και τώρα που μιλάμε ολοκληρώνουμε μία έκθεση η οποία έχει μία ολοκληρωμένη εικόνα για την κατάσταση της εξέλιξη της επιδημίας και για το ποιε είναι οι προκλήσεις για μας. Λοιπόν, θα κάνω κάποιες ε, γενικές σκέψεις λοιπόν για την επιδημία είναι αλήθεια ότι μπορούμε να παρατηρήσουμε εδώ και εκεί κάποια σημάδια που μας κάνει να σκεφτόμαστε ότι είμαστε στην αρχή μιας φάσης, ενός σταδίου που αποκοινούμε όλους ε, όσους δραστηριοποιούνται και τις κυβερνήσεις στην περιοχή, στην περιοχή θα αρχίσουμε να ελέγχουμε την επιδημία. Έχω κατά νου στατιστικά στοιχεία που μόλις δημοσιεύτηκαν σε ό,τι αφορά την κατάσταση στη Λιβερία και που μας κάνουν να σκεφτούμε ότι σε κατέργαστος ε, αριθμούς ο αντίκτυπος της επιδημίας στη Λιβερία θα μπορούσε ίσως να είναι κάπως λιγότερο βίος σε σχέση με το παρελθόν. Και θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η Λιβερία στο τέλος της Άνοιξης είχε κηρυχθεί μια πρώτη φορά εμπολαφρή, ότι δεν είχε εμπολαμβανθεί και τώρα έχει τα πιο δραματικά στατιστικά στοιχεία. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Τι μας μαθαίνει αυτό το φαινόμενο. Καταρχήν νομίζω ότι πρέπει να είμαστε σαφείς ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποκτήσουμε πληροφορίες και αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία. Απλώς ε, γιατί ακόμη αντιμετωπίζουμε ε, κάποια ε, φαινόμενα που έχουν να κάνουν με πολλαπλές ταυτοποίησεις ε, του ίδιας περίπτωσης και η βάση των αστικών στοιχείων από την οποία, τις οποίες εργαζόμαστε δεν είναι σταθερή. Δεύτερον, ο ιός, η επιδημία, είναι ένα φαινόμενο ζωντανό, ένα εξελίξη, συνεχώς αλλάζει. Αυτό είπε είναι η εικόνα της επιδημίας σήμερα, δεν θα είναι απαραίτητα η φωτογραφία της επιδημίας αύριο και τα λοιπά Δύο παραδείγματα. Στη Σιέρα Λεόνε οι αρχές ανησυχούν για το εξή, αφού επικεντρώθηκαν ε, για πολύ καιρό στις ε, περιφερειακές ε, και στην στις περιφερειακές περιοχές, επανέρχεται η νόσος και είναι πάρα πολύ διαφορετικά ο τρόπος που ξεσπάει η επιδημία στις πόλεις παρά στην Υπεθρό. Στη Γουινέα υπήρχε μια πολύ ενισχυτική κατάσταση σε μια και περιοχή, δηλαδή στα δάση της Γουινέας. Εκεί έχουμε πολύ λίγες πληροφορίες για το πώς αναπτύσσεται, πώς εξελίσσεται η επιδημία και πρέπει κατεπηγόντως να ενισχύσουμε την παρουσία μας. Τέλος, στη Λιβερία αν ε, πράγματι εξακολουθεί να είναι ισχυρή κατάσταση στη Μονοροβία. Τα νούμερα ίσως σημειώνουν κάποια μείωση, αλλά και η Λιβερία όπως και η Σιέρα Λεόνε γνωρίζουν πλήρως ότι θα πρέπει πολύ γρήγορα μαζί με τους εταίρους τους ε, και ε, με όσους δρούν στην περιοχή να βρουν μια νέα διαφορετική στρατηγική προσέγγισης και καταπολέμησης της επιδημίας. Να αναφέρω κάποια λόγια για τις εναλλακτικέ. Μέχρι τώρα είχαμε εστιάσει τις προσπαθίες μας κυρίως στο στάδιο της θεραπείας. Εξού και η δημιουργία υποδομών και πάλι σήμερα συνομίλησα με τους γιατρούς χωρίς σύνορα από το Βελγικό τμήμα κάποιον εκπρόσωπο του βιβλικού τμήμα που έχει πολύ μεγάλη εμπειρία και μου είπε ναι είναι αλήθεια, του είδα, ποτέ δεν ε, είχαν τόσο ευρείες υποδομές. Δηλαδή μιλάμε για εκατοντάδες κρεβάτια στη Γουινέ και στη Λιβερία. Αυτή ήταν ε, η πρώτη αντίδραση. Δηλαδή να αναπτύξουμε κάποια κέντρα θεραπείας, βαριές, δαπανηρές δομές, εξορισμού ολιγάριθμες που απαιτούν πολύ προσεκτικό σχεδιασμό, δηλαδή πώς ε, θα υπάρχει και κένωση των απαρημάτων κτλ. Χρειάζεται πάρα πολλής χρόνος να εγκαθιστηθούν, να δημιουργηθούν και γίνεται αυτό διαπαντός. Όπως ε, σας είπα, η επιδημία αλλάζει συνεχώς πρόσωπο και μπορεί να εξελιχθεί πολύ γρήγορα από μια γεωγραφική περιοχή σε μια άλλη. Και ανοίγω μια μικρή παρένθεση, Πρόεδρε, για να φυστήσω την προσοχή σας στο ότι φτάνουμε ε, τώρα στις χώρες το τέλος της ε, περίοδου των βροχών. Και το πρόβλημα που συνδέεται με τις μετακινήσεις των πληθυσμών θα θεθεί όχι μόνο για τις τρεις πληγήσεις χώρες σήμερα, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος να αρχίσει να τίθεται και για τις όμορες χώρες. Και κλείνω αυτό που είναι μια υποσημείωση προς τη στιγμή, αλλά μπορεί να γίνει μια συγκεκριμένη ανησυχία για μας. Είμαστε πολύ ανησυχοί όταν παρατηρούμε τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται ε, η περίπτωση στο Μάλι χρειάστηκαν ώρες ε, για να ταυτοποιηθεί το παιδί ε, που νοσούσε από την έμπολα ενώ είχε όλα τα συμπτώματα και δεν μπόρεσαν παρά να εντοπίσουν πολύ λίγους ανθρώπους με τους οποίους ήρθε σε επαφή. Και δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει στην Μπουργκίνα Φάσο. Φανταστούμε μια στιγμή ότι αν ανοιχνευτεί ένα κρούσμα έμπολα στην Μπουργκίνα Φάσο, τι θα γίνει. Μπορείτε να φανταστείτε τις συνέπειες ε, ως προς τις θεραπείες. Όταν μάθαμε ότι η Νιγερία ε, είχε πληγεί, όλοι πραγματικά να τριχιάσαμε, θα μπορούσαμε να φανταστούμε τι μπορεί να γίνει ε, αν αναπτυχθεί η επιδημία του έμπολα σε μια πόλη όπως το Λάγκος. Όμως ελήφθησαν ταχείες, ταχεία μέτρα και μπορούσαμε τελικά να κηρύξουμε την Νιγερία ως μια χώρα χωρίς έμπολα. Όμως ε, τώρα το ότι είμαστε στο τέλος ε, της περιοχής των λογών και θα υπάρχουν μετακινήσεις του πληθυσμού σημαίνει ότι θα πρέπει να επαγρυπνούμε σε ό,τι αφορά τις όμορες χώρες. Και κλείνω την παρένθεση και επανέρχομαι τώρα στην κατάσταση της τρεις χώρες. Η επιδημία λοιπόν θα κινηθεί και σίγουρα θα αλλάξει και πρόσωπο, θα αλλάξει και εικόνα. Εξού και μια όλο και μεγαλύτερη προσοχή που ε, θα πρέπει να δοθεί σύμφωνα με τις κυβερνήσεις και τους παίκτες της περιοχής ότι αφορά ε, την θεραπεία ανάντι και κατάντι. Ανάντι να εντοπιστούν στην πηγή ε, τα κρούσματα και να απομονωθούν ως δυνατόν ταχύτερα. Και αυτό δεν συνάδει πάντα με την αναγκαιότητα να μεταφερθεί κάποιος σε ένα κέντρο που μπορεί να είναι δεκάδες χιλιόμετρα μακριά. Έτσι λοιπόν πρέπει να υπάρχει ανάγκη να έχουμε πιο ελαφρές υποδομές, πιο κοντά στις κοινότητες και ε, πρέπει να αλλάξει και η νοοτροπία ε, για να δώσουμε μεγαλύτερο ρόλο στις βασικές συλλογικότητες. Ο ε, Ποργός της μου έδωσε κάποια στατιστικά στοιχεία. Όταν ανοιχνεύεται ένα πρώτο κρούσμα έμπολα σε μια οικογένεια, η αλυσίδα μετάδοσης είναι τέτοια, ε, στην ίδια οικογένεια ανακαλύπτεται ένα πλέον κρούσμα τη βδομάδα. Πρέπει λοιπόν να διακόψουμε αυτή την αλυσίδα μετάδοση στο συντομότερο και πώς θα το κάνουμε αυτό εντοπίζοντας και απομονώνοντας το συντομότερο τους ασθενείς πριν να τους μεταφέρουμε ίσως ε, σε ένα κέντρο θεραπείας όπου επιδεινώνεται η κατάσταση του ασθενή. Πρέπει λοιπόν σήμερα αυτά να τα σκεφτούμε ανάντι. Πριν το χάρη οι Ηνωμένε Πολιτείε, ω στην τη Λιβερία, είχαν αρχικό σχέδιο να κατασκευάσουν ένα μεγάλο αριθμό υποδομών με εκατοντάδε κρεβάτια και τελικά αναθεώρησαν για να ε, πολλαπλασιάσουν τις ε, μικρές ε, δομές με 10 κρεβάτια. Τώρα, Κατά αντιπρεσβευτές ε, φέρθηκαν φέρθηκαν ε, στις ε, ταφές, στις ασφαλείς ταφές. Η Διεθνή Ομοσπονδία του Ερυθρού Σταυρού έχει πολύ μεγάλη εμπειρογνωμοσύνη στο θέμα και όλοι αναγνωρίζουν ότι ο αντίκτυπος της παρέμβασης του Ερυθρού Σταυρού σε ό,τι αφορά την πρόληψη της διάδοσης, της μετάδοσης της νόσου κατά την ταφή είναι κάτι πολύ σκόπιμο. Δεν, ε, η διαδικασία που πρέπει να ακολουθεί κατά την ταφή δεν συνάδει με τα ντόπια έθιμα, ε, όμως ε, πρέπει να προσέξουμε εκεί για να μην βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου ένας ε, άνθρωπος φεύγει από ένα κέντρο θεραπείας, κανένας δεν έχει νέα του και αν τελικά ε, κάποιος από την οικογένεια πάρει τηλέφωνο στο κέντρο, λέει ότι πέθανε αυτός ο άνθρωπος ε, και τελικά έχει ε, αποτεφρωθεί. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να εργαστούμε από αυτό και πρέπει να κάνουμε μια αποτελεσματική δουλειά, δηλαδή στο στάδιο μετά το θάνατο. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά παραδείγματα, αλλά τι σημαίνει αυτό. Όποια και αν ε, είναι η μορφή που παίρνει η επιδημία, όποιε ε, και αν είναι οι αριθμητικέ ενδείξει που μπορεί να έχουμε σήμερα, Όποιε και αν είναι οι στρατηγικές που αναπτύσσονται, η ανάγκη για τους πόρους δεν θα μειωθεί. Μην πιστεύετε ότι οι επικεντρωμένες στρατηγικές ε, είναι λιγότερο δαπανηρές από ότι το να επενδύουμε σε μεγάλε δομέ. όπως κάναμε μέχρι σήμερα. Τώρα για ποιους πόρου μιλάμε. Πρόκειται για υλικού πόρου, οικονομικούς πόρου και σε είδου, αλλά και για ανθρώπινους πόρου. Θα σα ε, αναφέρω μία φράση ενός ανθρώπου που συνάντησα σε μία από τις τρεις χώρες. Τότε με αυτό μου είπε οι πιστώσεις και οι υποδομές δεν είναι τίποτα αν δεν έχουμε τους ανθρώπους για να τα χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά. Και δεν έχουμε ανθρώπινο δυναμικό. Έτσι λοιπόν η πρώτη προτεραιότητα είναι να καταφτάσουν στην περιοχή ανθρώπινοι πόροι ε, που θα έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση και τα κατάλληλα προσόντα. Οι πόροι αυτοί θα μπορούσαν να προέρχονται από την Ευρώπη. Και επιμένω στο θέμα της κατάρτισης και των προσόντων. Θα είμαι κάπως σκληρός, ε, Πρόεδρε, αλλά ούτε γουινέο της Σιέρα Λεόνε ούτε η Λιβερία δεν είναι ε, κάποια παιδεία για ανθρώπους που έχουν αυτοκτονικές τάσεις. Εδώ ε, πρέπει να οργανωθούμε όχι μόνο στο θέμα της δημόσιας υγείας αλλά και στο θέμα της επιμελητίας. Ξέρετε, ως προς την επιμελητία είναι πάρα πολύ δύσκολη οργάνωση, δηλαδή να μεταφερθούν τα υλικά, ε, να συντηρηθούν ε, τα υλικά και τα λοιπά. Έχουμε ε, αυτούς τους ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση απλώς μέσω της ε, δημιουργίας ενός clearing house και έχει ληφθεί μια παρόμοια πρωτοβουλία από τη Γερμανία. Μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί από όσο ήμασταν μέχρι τώρα σε ό,τι αφορά στο να συνδέσουμε την ευρωπαϊκή προσφορά με τη ζήτηση και έχουμε προγράμματα κατάρτισης από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, καθορίζονται τα ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων, ε, προγράμματα κατάρτισης ε, που θα μπορούσαμε να θέσουμε σε εφαρμογή πριν ε, από την αναχώρηση από την Ευρώπη. Έτσι λοιπόν είναι προτεραιότητα όταν έχουμε το κατάλληλο προσωπικό. Μπορούμε να εργαστούμε και με άλλους εταίρους. Όταν ήμουν επιτόπου εγώ γνώρισα κάποιον ε, που εκπροσωπούσε ε, τους κουβανούς γιατρούς. Είναι 150 άτομα, δεν είναι πολλοί, αλλά είναι άνθρωποι με μεγάλη εμπειρία που έχουν εργαστεί αλλού για άλλες επιδημίες, γνωρίζουν καλά ε, την περιοχή και το πεδίο και υπάρχουν ε, κάποια κέντρα όπου θα εργαστούν και μιλάμε για τα κέντρα που μόλις εγκαινιάστηκαν από το USAID στη Λιβερία. Και εκεί θα εργαστούν κουβανοί γιατροί. Υπάρχει και άλλη μία πρωτοβουλία που αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή της ε, Αφρικανική Ένωση, μία αποστολή Ένωσης, μία αποστολή που υποστηρίζουμε. Θα είναι μία αποστολή με 2.000 άτομα που θα καταναμηθούν στις τρεις χώρες οι πρώτοι έχουν ήδη φτάσει, η μπροστοφυλακή αν θέλετε, η, Ευρωπαϊκή, συγγνώμη, η Αφρικανική Ένωση μας είπε ότι έχει κατορθώσει να καταρτήσει χίλια άτομα, λείπουν ακόμη χίλια άτομα, πρόκειται για άτομα που γνωρίζουν πώς να εργαστούν σε αυτές τις περιοχές. Και ξέρετε, τον εργαστεί κάποιο εκεί επί τόπου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εμεί δεν μπήκαμε ε, στα κέντρα θεραπείας. Είδα όμως ανθρώπους να βγαίνουν από τις κεντρικές μονάδες, όπου είναι τα βαριά περιστατικά και μπορώ να σας πω ότι ένας γιατρός που εργάστηκε μία ώρα σε αυτά τα κέντρα είναι εξαντλημένο. Είναι σαν να έτρεξε μαραθώνιο. Του είδαμε λοιπόν να βγαίνουν και πρέπει να ξέρουμε ότι η δουλειά σε αυτά τα κέντρα είναι ιδιαίτερα απαιτητική, χρειάζεται σοφροσύνη, τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, φυσικές αντοχές, σωματικές αντοχές και άνθρωποι που θα εργαστούν εκεί θα πρέπει να έχουν την κατάλληλη κατάρτιση και εκπαίδευση. Αυτά για το πώς θα απαντήσουμε στην κρίση του έμπολε. Τώρα, γενικά. Εν τω μεταξύ, οι αποφάσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ελήφθησαν για την ε, προετοιμασία του Ευρωπαίου Συντονιστή. Και ξέρετε, ως Ευρωπαίος Συντονιστής ο κύριος Τηλιανίδης θα έχει κάποιες ε, αρμοδιότητες που θα ξεπερνούν τις αρμοδιότητες του Επιτρόπου ανθρωπιστικής ε, βοήθειας. Ε, ουσιαστικά θα αναλάβει κάποιες αρμοδιότητες που σήμερα ανήκουν σε άλλες υπηρεσίες. Ο κύριος Πρεσβευτής αναφερθήκε στο θέμα του συντονισμού και συμφωνώ απόλυτα μαζί του, είναι κατεπήγον και πρέπει να αποφύγουμε τώρα που η διεθνή κοινότητα ξυπνάει, αφυπνίζεται, να ξαναβρεθούμε σε μια κατάσταση όπως αυτή είδαμε τότε στην Αιτή. Και εγώ θεωρώ ότι τότε είχαμε τη δράση πάρα πολύ αργά. Πρέπει λοιπόν να είναι καλό ο συντονισμό, είναι σαφέ. Υπόθηκε αυτό και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ότι διασφαλίζουμε έναν ευρωπαϊκό συντονισμό στο πλαίσιο ενό παγκόσμιου συντονισμού και υπό την ευθύνη του συστήματο των ΗΠΑ. εμεί. χαιρετήσαμε τον διορισμό του κυρίου Ναβάρο από τα Ηνωμένα Έθνη και χαιρετήσαμε την απόφαση της ε, ε, δημιουργίας της NMR, e της αποστολής για να αντιμετωπίσει τον έμπολα. Τώρα φτάνουν οι ε, ε, πρώτοι άνθρωποι εκεί. Εγώ συνάντησα ηθήνοντες από τις τρεις χώρες. Ε, ο πιο παλιός ε, της NMR e ήταν εκεί εδώ και ένα μήνα. Πρέπει λοιπόν ε, να, δώσουμε και κάποιο χρόνο, όχι υπερβολικό όμω, αλλά θα πρέπει να αφήσουμε χρόνο στην ΕΝΜΗΡ για να αναπτυχθεί και να παίξει το ρόλο τη. Ποιο θα είναι ο ρόλο τη τώρα. Αυτό θα καθοριστεί ανάλογα με τι χώρε, αλλά κάθε φορά επιμείναμε στο να αναλαμβάνουμε δράση πολύ γρήγορα θα υπάρχει και ένα επιχειρησιακό έγγραφο που θα βγει πολύ σύντομα και τα λέει αυτά για να καλύψουμε τα κενά και να διασφαλίσουμε τον απαραίτητο συντονισμό μεταξύ όλων των ε, οργανισμών των Εθνών και των stakeholders. Πρόκειται λοιπόν για ένα ευρωπαϊκό συντονισμό που έχει σκοπεύει να δώσει μια ολοκληρωμένη και με μία απάντηση στα πλαίσια μιας παγκόσμιας προσπάθειας ε, που όμως την ευθύνη την έχουν τα Ενωμένα Έθνη. Και κάτι ακόμη και κλείνω, συγγνώμη μακρηγόρησα. Και εδώ θέλω να επανέλθω σε αυτά που τέθηκαν από τις δύο πρεσβευτές της ε, παρεμβάσεις τους. Ακόμη κι αν σήμερα έχουμε ενώπιόν μας ε, μια πρωτοφανή κατάσταση, δεν μπορούμε να λέμε το ένα και μετά το αντίθετο, δηλαδή ε, δεν μπορούμε να λέμε ότι πρόκειται για μια πολυδιαστή κρίση και ταυτόχρονα μην ενδιαφερόμαστε για τις άλλες διαστάσεις της κρίσης. Οι από τους τρεις προέδρους της Σιέρα Λεόν και της Λιβερίας ε, και είχα την τιμή να τη συναντήσω μου είπαν ε, και χρησιμοποίησαν την ίδια διατύπωση ότι πρέπει σήμερα να αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε για μετά τον έμπολα. Οι κυβερνήσει αυτές ε, γνωρίζουν πλήρως το αν έχουμε μια μερική προσέγγιση πρώτα έμπολα και τα υπόλοιπα μετά θα βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου την ημέρα που θα κηρυχθούν ε, απαλλαγμένες από τον έμπολα οι χώρες, θα εγκαταλειφθούν από όλο τον κόσμο και θα βυθιστούν στην κρίση. Πρέπει αυτό να το αποφύγουμε με κάθε τίμημα. Έτσι λοιπόν είναι η ευθύνη των δωρητών να δεσμευτούν σήμερα σε αυτή την προσέγγιση που αποκαλείται resilience based, δηλαδή που βασίζεται στην ανθεκτικότητα και να μας επιτρέψει στον τομέα της υγείας, ε, του επισητισμού, της εκπαίδευσης στη Σιερέ Λεόνε. Έχουμε και μια μεγάλη επισητιστική κρίση επειδή διεκόπησε ο εφηδιασμός και λειτουργούν άσχημα, δεν λειτουργούν καλά οι αγορές, να υπάρχει ε, μία ανάληψη πρωτοβουλίας για να υπάρξει ανοικοδόμηση και να βρεθούν οι χώρες πέραν από την επιδημία του έμπολα σε μια κατάσταση που δεν θα είναι χειρότερη, αλλά τουλάχιστον να είναι στην κατάσταση παρόμοια με την κατάσταση που βρίσκονταν στην αρχή. Πρέπει να αναβιώσουμε λοιπόν, να δώσουμε όθηση σε αυτές τις οικονομίες που έχουν πληγεί από την επιδημία. Αυτά από μένα, Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που μας παρουσιάσατε τι σημαίνει επί Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η παρουσίαση και νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει και μια φάση μετά την αντιμετώπιση της κρίσης του έμπολα. Είναι σημαντικό λοιπόν να διδαχτούμε από τα διδάγματα του παρελθόντας σε ό,τι αφορά τώρα την ε, φάση που βρισκόμαστε τώρα. Αυτό που προέχει είναι η άμεση αντιμετώπιση του ιού. Και γι' αυτό λοιπόν θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση από τους συναδέλφους. Έχουμε εδώ και τους συναδέλφους από την Επιτροπή DG ε, DEFCO, από την Επιτροπή ε, ΟΠΗ. Θα μπορείτε να πάρετε το λόγο στο τέλος, αν το επιθυμείτε να προσθέσετε κάτι, αλλά θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση από τα μέλη της Επιτροπής, ο κύριος Γκιόρενς, ο οποίος θα είναι και ο εισηγητής της Επιτροπής μας για τον εμπόλα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να πατήσω φοροτιμή ε, στους γιατρούς χριστιανών που κάνουν εξαιρετική δουλειά. Ήδη έχουν λάβει το βραβείο Νόμπελ και νομίζω το αξίζουν για δεύτερη φορά για τη δουλειά που κάνουν στην ε, Αφρική. Θα ήθελα επίση να αποτύσσω φορά τιμή στον κύριο Ντεμπράουρ. Δεν ε, είναι προφανέ να μεταβαίνει κάποιο σε αυτέ τι χώρε και να εκτίθεται στον κίνδυνο και να επανέρχεται με μια ιδιαίτερα διαφωτιστική ανάλυση. Σα ευχαριστούμε για αυτή τη διαφωτιστική ανάλυση και ευχαριστούμε και του δύο προσευχητές. Όμως θα είμαι λίγο πιο επικριτικός για τους δύο πρώτους ομιλητές και να πω δύο λόγια για την έκθεση. Ε, ε, έχουμε δύο χρόνους. Καταρχήν έχουμε το κατεπήγον, ε, δεύτερον έχουμε τα διδάγματα της επιδημίας και νομίζω ότι εδώ πρέπει να εξετάσουμε και το θέμα της διακυβέρνησης σε καθολικό επίπεδο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, επίπεδο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, πολύ ε, γρήγορα υπήρξαν αντιδράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση από το Μάρτιο εκταμιεύτηκαν ε, καταμία. όμως το ίδιο δεν ισχύει για τα κράτη-μέλη αυτό το βλέπουμε. Υπήρξαν πολλές προφάσεις που εφευρέθηκαν από τα κράτη-μέλη για να μην κάνουν τίποτα. Η κρίση αυτή στις αρχές Μαρτίου ξέσπασε στην Αφρική και κάνω αυτή τη γεωγραφική αναφορά γιατί ε, όταν ε, υπάρχουν ε, μόνο οι μαύροι που πεθαίνουν ε, σε αυτή την περιοχή ε, δεν είναι οι δικές μας αντιδράσεις όπως θα έπρεπε. Ο Παγκόσμιος Οργανικό Υγείας ήδη αναφέρθηκε στο μέα κούλπα του και αναγνώρισε τα λάθη του σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης και είναι συγχώρητα τα λάθη αυτά. Η κατάσταση στην οποία ε, βρισκόμαστε σήμερα δεν είναι ένα status quo, αλλά status quo ενεξελίξει. Χαίρομαι που είπατε ότι ίσως μπορούμε να αμφισβητήσουμε τις πτυχές, τις εκθετικές πτυχές της κρίσης. Ελπίζω να έχετε δίκιο. Θα πρέπει να το ευχόμαστε τουλάχιστον, γιατί είμαστε πάρα πολύ απογοητευμένοι για την αντίδραση που θα έπρεπε να υπάρχει απέναντι σε αυτήν την κρίση. Μια άλλη πτυχή που θέλω να αναφέρω είναι η κρίση μέσα στην κρίση. Στη Λιβερία το σύστημα υγείας κατέρεε ήδη από το Δεκέμβριο. Υπήρχε κενό ως προς τους γιατρούς και όλοι όσοι θρέπευσαν τους ασθενείς ε, τελικά κατέληξαν. Κατέρευσε λοιπόν το σύστημα και διώχθηκαν ε, οι άνθρωποι από τα κέντρα θεραπείας ε, γιατί δεν χωρούσαν πλέον. Εσείς περιγράψατε πολύ καλά την κατάσταση για τις ταφές. Ε, υπήρξαν κάποιες αφρικανικές παραδόσεις και αυτό ήταν ένα ακόμα εμπόδιο που έπρεπε να υπερβούμε. Η Κομισιόν, όπως είπα, αντέδρασε αρκετά γρήγορα. Η αντίδραση των ε, κρατών μελών δυστυχώς δεν ήταν η αρμόζουσα η κατάσταση στην Αφρική ήταν εξή. Έλειπαν οι γιατροί ε, και ιατρικό προσωπικό και θα έπρεπε ε, γιατροί από τις βόρειες χώρες να μεταβούν εκεί. Χρειάζονται ανθρώπινοι πόροι. Εγώ πραγματικά θαυμάζω του ανθρώπου που κάνουν αυτή τη χειρονομία. Για να μπορούν να γίνουν τέτοιε χειρονομίε χρειάζεται κάτι. Ζητούν να υπάρχει μια ικανότητα εκένωσης και αυτή η ικανότητα εκένωσης ε, συζητείται για μήνες. Η Γαλλίδα νοσοκόμος έπρεπε να περιμένει τρεις μέρες. Ευτυχώς που είχε καλή έκβαση, αλλά αν θέλετε οι άνθρωποι να μεταβούν σε αυτές τις περιοχές για να βοηθήσουν θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός εκένωσης. Έχουμε και ένα νόμιμο συμφέρον ε, να δώσουμε κάποιες εγγύησεις στους ανθρώπους που μεταβαίνουν στην περιοχή για να μπορούν να θεραπευτούν. Να πω κάτι για την απόφαση του Συμβουλίου να διορίσει τον κύριο Στυλιανίδη ως συντονιστή για ε, τον έμπολα. Πολύ καλό είναι να διορίζουμε ένα συντονιστή και θαυμάζω τον κύριο Στυλιανίδη, ο οποίος ε, έκανε και μια εξαιρετική ακρόση. Θα δώσει το παράδειγμα σε αυτήν την περιοχή, αλλά θα δώσει και, θα παροτρύνει και άλλους γιατρούς, είναι και ο ίδιος γιατρός. για να βοηθήσει να καλυφθεί αυτό το κενό στο οποίο αναφέρθηκα. Το θέμα δεν είναι μόνο να ξέρουμε να έχουμε ένα, ένα συντονιστή, αλλά αν τα κράτη-μέλη είναι έτοιμα να δεχτούν τον συντονισμό. Έχω σοβαρές επιφυλάξεις. Ή είναι έτοιμα, επομένως πρέπει να ρωτήσουμε γιατί δεν ήταν έτοιμα πιο πριν. Και εδώ υπάρχουν ευθύνες να καταλογιστούν και σας διασφαλίζω, εγώ θα είμαι αρκετά σκληρός απέναντι σε όλες αυτές τις ελλείψεις που είναι σχεδόν ασυγχώρητες και δεν θα ήθελα να υπάρχει ούτε ένα εμπόδιο πίσω από το οποίο να μπορούσαμε να κρυφτούμε ή να βρούμε προφάσεις για να κάνουμε τίποτα. Ω Κομισιόν, μα κάνετε τον κατάλογο όλων των εμποδίων που τίθενται εφ' για να σταλούν γιατροί επιτόπου ε, μια πλήρη λίστα, ένα πλήρη κατάλογο και εμείς θα είμαστε πάρα πολύ σκληροί με αυτούς που δεν είναι έτοιμοι να άρουν τα εμπόδια αυτά. Αν αυτά τα εμπόδια είναι δημοσιονομικής φύσης θα πρέπει να τα υπερβούμε. Αν αφορούν τη χρηματοδότηση θα πρέπει να τα υπερβούμε. Δεν θα πρέπει να μπορούμε να κρυφτούμε πίσω από τέτοιες δυσκολίες. Και χρειαζόμαστε και ένα master plan. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το master plan ακόμη δεν υπάρχει, δεν έχει συσταθεί. Πολύ ωραία να εγγράφονται αυτά υπό την ευθύνη της διεθνούς κοινότητας. Νομίζω ότι η διεθνή κοινότητα ε, δυστυχώς δεν αντέδρασε όπως έπρεπε. Ο κύριος Ματιέ μίλησε για την παγκοσμιοποίηση της αδιαφορίας. Νομίζω ότι πρέπει να ξεπεράσουμε το στάδιο αυτό, ότι έχουμε ξεπεράσει το στάδιο αυτό για το μέλλον θα πρέπει να συγκρατήσουμε ότι όλες οι επενδύσεις που ζητάμε εδώ και χρόνια, τουλάχιστον η επένδυση του 20% των δαπανών για την παγκόσμια αναπτυξιακή βοήθεια στους βασικούς κοινωνικούς τομείς είναι μια μακροπρόθεσμη επένδυση. Και τώρα αποδεικνύονται όλα αυτά. Είδαμε τι έγινε στην, στην Ιγυρία. Στην Ιγυρία δεν έγινε μεγαλύτερο κακό από ό,τι στη ΣΥΠΑ. Δεν ε, υπήρξαν ε, θάνατοι σε επίπεδο γιατρών ή ιατρικού προσωπικού. Αν λοιπόν υπάρχουν τα μέσα, αν δοθούν τα μέσα στους Αφρικανούς, θα μπορέσουν και αυτοί να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Από αυτή τη σκοπιά, λοιπόν, ε, εκ των υστέρων αυτό αποτελεί μια εξήγηση Πρέπει να διεκδικήσουμε την υλοποίηση αυτής της μεγάλης διάσκεψης και πρέπει όλοι να συνεισφέρουμε στην οργάνωσή της. Αυτές τις σκέψεις είχα να κάνω σε σχέση με τις τρεις παρεμβάσεις που ακούσαμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και άλλοι πέντε έχουν ζητήσει το λόγο και έχουμε μόνο λίγα λεπτά στη διάθεσή μας. Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό. 90 λεπτά στον καθένα, λοιπόν, μια μισή 1,5 λεπτό για να κάνετε την ερώτηση και ξεκινάμε με τον κύριο Ντομπρόφσκι. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Πάρα πολύ σύντομα να πω δύο λόγια ε, συντονισμός και επικοινωνία. Για τον συντονισμό συμφωνώ με τον εισηγητή μας ότι παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή ήταν εκεί, τα κράτη-μέλη υστερούν και τώρα το θέμα είναι κατά πόσον θα αποδεχτούν τον συντονισμό αυτό. Είναι όμως πραγματικά κατεπήγον το θέμα. Όταν υπήρξε η πρώτη ανταπόκριση, υπήρξε μια κατανομή των εργασιών που προφανώς δεν ανταποκρινόταν ε, στις καλύτερες δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Γαλλία, στη Ρουμανία, η ΕΠΑ, στη Λιβερία. Πού ήταν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της στην στιγμή εκείνη. Συντονισμός λοιπόν. Εξακολουθεί να παρατελεί θέμα κλειδί. Και χαίρομαι που βλέπω ότι επενέθηκε ο κύριος Τηλιανίδης και προφανώς και προσβλέπουμε στη δουλειά που θα κάνει σε ό,τι αφορά το συντονισμό. Και η επικοινωνία θεωρώ ότι αποτελεί ένα θέμα κλειδί για να βρεθεί η ισορροπία, για να υπάρχει η δέσμευση του Κοινούργιου Επιτρόπου στη Δυτική Αφρική Αυτό βοήθησε με δύο τρόπους, ότι καταρχάς θέλουμε να απομονώσουμε τον έμπολα, αλλά όχι τις χώρες, αλλά και αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση στην Ευρώπη με σόφρονα τρόπο, χωρίς να σπείρουμε πανικό. Διαδίδοντας το σωστό μήνυμα και το πώς λοιπόν μπορούμε να βρούμε αυτή την ισορροπία. Αυτό είναι το ερώτημά μου και δεν μπορώ να μιλήσω παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Σγκυρέρο. Ευχαριστώ. Ο κ. είπε ότι κάποιος ε, του είπε ότι αν μετά το τέλος του έμπολα ε, θα εγκαταλείπαμε τις χώρες που είναι τώρα σε κρίση. Και η ερώτησή μου είναι αν σε κάποιο βαθμό δεν τις έχουμε ήδη εγκαταλείψει στην κοινή γνώμη των δυτικών χωρών. Γιατί μετά από τη στιγμή της κρίσης ε, με κρούσματα στις Ηνωμένες και στην Ισπανία, ήταν μια στιγμή όπου αυξήθηκε η παγκοσμία ανησυχία για τον ομολογικό πυρετό του έμπολα. Από τη σκοπιά των μέσων μαζικής ενημέρωσης εξαφανίστηκε ή μειώθηκε το ενδιαφέρον. Αυτό αναμειγνύεται με ένα στιγματισμό, στο οποίο αναφέρθηκαν και οι πρεσβευτές. Ένα στιγματισμό που καταγγέλθηκε από τους γιατρούς χωρίς σύνορα. Επισήμεναν ότι και αυτοί έχουν προβλήματα, γιατί στιγματίζονται <laughs> επειδή πάνε στην Αφρική. και υπάρχει ένα σύμβολο που δεν είναι δευτερεύον. Χθες στο μαραθώνιο της Νέας ε, Υόρκης, ο μαραθώνιος της Υόρκης έγινε χωρίς ε, την παρουσία αθλητών από χώρες ε, της Αφρικής με έμπολα και αυτό μεταφέρθηκε στην κοινή γνώμη ως ένα κόσμο στοιχείο στιγματισμού. Οι προσβευτές αναφέρθηκαν στην άμεση βοήθεια στις χώρες. Δεν ξέρω αυτό σχετίζεται με αυτό που λέμε budget support, δημοσιονομική σύρρηξη, δηλαδή να μεταφέρουμε άμεσα τους φόρους στις κυβερνήσεις. Όμως, αυτό θα ήταν δύσκολο σε ό,τι αφορά την ταχεία απάντηση που πρέπει να δώσουμε στο πρόβλημα. Αν έχουμε 30 δευτερόλεπτα στη θέση μας, θα θέλω να μου πείτε πώς συνδυάζουμε την άμεση βοήθεια στις χώρες με το συντονισμό της βοήθειας που θα έρθει από διάφορους δωρητές ή διεθνείς οργανισμούς. Ευχαριστώ. Ο ο είναι ο Αντιπρόεδρος Βοσγίνεβα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερως που συμμετείχα στη συζήτηση αυτή που περιέχει πολλά καλά στοιχεία για την Επιτροπή μας. Πολύ καλή ενημέρωση. Εξαιρετική. Νομίζω ότι θα πρέπει να κοιτάξουν το θέμα συνολικά. Είναι σαφές ότι ο κύριος Ήλα και το έθεσαν το θέμα αυτό άλλωστε, ότι πολλά θα πρέπει να γίνουν εκ παραλλήλου. Καταρχάς, περιορισμός. Δεύτερον, εφαρμογή των τοπικών δυνατοτήτων, χρήση των ε, τοπικών δυνατοτήτων, αναγνώριση των παραγόντων οικονομικής ύφεση. Τέταρτον, μία σύμβαση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών που πλήττονται από τον έμπολα για βοήθεια. Δεν χρειάζεται να το λέμε σχέδιο Μάρσαλ κάθε φορά. Κάποια συμφωνία μεταξύ ημών, εν και των χωρών που έχουν πληγεί από τον έμπολα, ότι θα τις βοηθήσουμε να αναδομήσουν ό,τι έχει γίνει στην οικονομική του σφαίρα. Το ενδιαφέρον όμως που άκουσα από τον κύριο Ντεμπράουερ είναι ότι ψάχνουμε άτομα εκπαιδευμένα που μπορούν να αναλάβουν θέματα επιμελητίας, που μπορούν να μεταφέρουν και να τα μετακομίσουν ασθενείς, που έχουν πειθαρχία και το καθεξής. Όταν έκανα μία πρόταση στην Ολομέλεια ότι θα πρέπει να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη μας να ζητήσουν κάποια από τη βοήθεια που έχουν στο συστητικό ιατρικό προσωπικό τους που κάθονται και περιμένουν με χτύπησε στα δάχτυλα η αριστερά. Αλλά ας ξεχάσουμε την πολιτική. Εδώ μιλάμε για να σώσουμε ζωές. Αν έχουμε λοιπόν κόσμο που έχει την ικανότητα επιμελητίας, με πειθαρχία, με ιατρική εκπαίδευση και που δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει, θα πρέπει να τους αξιοποιήσουμε. Θα πρότεινα λοιπόν να πάτε στο Συμβούλιο ότι βουαλά το Κοινοβούλιο έχει μία λύση. Να κοιτάξουμε το ιατρικό προσωπικό του στρατιωτικού, των στρατιωτικών σωμάτων των χωρών μας. Και έτσι πολλοί κόσμος θα μπορούσε να αποσταλεί εκεί και να κάνει πραγματικά καλό. Ευχαριστώ. Κάποια κρατημέλη νομίζω το κάνουν αυτό. Το Ηνωμένο Βασίλειο και είπα, ΕΕ, νομίζω και κάποιες άλλες χώρες αποστέλουν εκεί ιατρικό προσωπικό. Η κυρία Σάντσες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγεία, το 5% των νεκρών στι χώρε τη Δυτική Αφρική ε, σε σχέση με το κρούσμα του έμπολα είναι το προσωπικό υγεία, το ιατρικό προσωπικό και αυτό μα δείχνει ότι υπήρχε έλλειψη πόρων, ε, πόη συστήνει να υπάρχουν 41 ε, ε, άτομα του προσωπικού για 3.000. Ε, Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη έλλειψη για επένδυση στον τομέα της δημόσιας υγείας και σε τέτοιες περιπτώσεις δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Εγώ θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κοινοβούλιο και συγκεκριμένα αυτή η Επιτροπή, η Επιτροπή Ανάπτυξης, να το σημειώσει αυτό, έτσι ώστε να το έχουμε κατά νου για την επόμενη φορά. Δηλαδή πόσο σημαντικό είναι να αναπτύσσουμε ένα δημόσιο και καθολικό σύστημα υγείας που να είναι ισχυρό με τους απαραίτητους πόρους. Θα ήθελα επίσης η έκθεση που περιλαμβάνει η έκθεση να συμπεριλαμβάνει και αυτή την ανησυχία θα ήταν πολύ καλό ο κύριος Στυλιανίδης ε, να έρθει σε επαφή και με τους ντόπιου εργαζομένους στον τομέα της υγείας και όχι μόνο ε, με τους εργαζομένους που έρχονται από άλλες χώρες και θα ήθελα η Κομισιόν ε, να σημειώσει όλα αυτά, συγγνώμη, Επιτροπή να σημειώσει όλα αυτά τα θέματα για να μην τα επαναλάβουμε. Ευχαριστώ τελευταία ομιλήτρια, κυρία Χόιμπαχ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και για την ε, παρουσίαση αυτή που κατέστησε σαφέ που βρίσκονται οι ελλείψεις μα και ο κύριος Γκούρεν ε, επισήμανε που κάναμε σφάλματα. Πολλά λοιπόν έχουμε να διορθώσουμε. Ας ε, στραφούμε τουλάχιστον και στην οικονομική αναδόμηση των χωρών αυτών. Τώρα το πιο σημαντικό είναι να διδαχθούμε από τα παθήματα τη κρίση αυτή. Γιατί δεν πρόκειται να είναι η τελευταία κρίση. Πολλέ άλλε ασθένειε απειλούν την ανθρωπότητα. Και είπατε, κύριε Ντεμπράουερ, ότι θα πρέπει να κάνουμε τώρα εκπαίδευση του προσωπικού. Τώρα είναι πάρα πολύ αργά. Τώρα βρισκόμαστε ήδη σε φάση κρίσης. Χρειαζόμαστε σχέδια για τις κρίσεις του μέλλοντος, χρειαζόμαστε σχέδια στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του ΟΗΕ, προκειμένου να είμαστε σε θέση άμεσης ανταπόκρισης σε τέτοιες ε, κρίσεις. Και τέτοιες ε, Μορφέ ανταπόκριση σε κρίσει μπορεί να περιλαμβάνουν και στρατιωτικό προσωπικό και στρατιωτικό υλικό. Αλλά αυτό θα πρέπει να ορίζεται εκ των προτέρων, προκειμένου του, τουλάχιστον να έχουμε μία προετοιμασία επί της αρχής σε τέτοιες περιπτώσεις κρίσεων. Να έχουμε κάποια βασική, κάποιο βασικό εξοπλισμό για να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε πιο γρήγορα, πολύ πιο γρήγορα. Και κάτι άλλο που με απασχολεί ιδιαίτερα και το οποίο το ακούσαμε είναι τα συστήματα υγεία που έχουν καταληθεί πλέον. Είναι σημαντικό τα συστήματα υγείας να σταθούν πάλι στα πόδια τους και να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό δεν είναι μόνο ευθύνη των χωρών αυτών, είναι ευθύνη όλων των κρατών, της διεθνούς κοινότητας και των βιομηχανικών κρατών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος, και τώρα θα δώσω το λόγο στους πρεσβείς και στον κύριο Ντεμπρούγερ, αλλά θα ήθελα να κάνω και εγώ μια ερώτηση στον κύριο Ντεμπρούγερ. Ο κύριο Τουλιανίδη πλέον είναι ο απεσταλμένο από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι επίτροπο. Είπατε δε ότι θα συντονίσει από πλευρά των κρατών μελών τι δράσει. Ξέρουμε τι σημαίνει αυτό για να απαντήσουμε στην ερώτηση του κύριου Γκούρεντ. Τι διαφορά έχει ε, η ιδιότητά του ω επίτροπο ή ως ε, ειδικός ταπεζαλμένος. Έχετε κάποια σχόλια να κάνετε παρακαλώ, κύριε Πρέσβη. Ε, δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσου πήραν το λόγο και εσά Να επανέλθω στο θέμα του συντονισμού. Οι τρεις προεδρευτές ε, πήγαμε στο Λουξεμβούργο και τα κάνουμε όλα μαζί ως πληγήσεις χώρες. Πήγαμε και στις κατοχώρες θα συναντήσουμε και την Βελγική κυβέρνηση σύντομα. Αλλά αυτό που σημειώσαμε είναι ότι κάθε μία από αυτές τις χώρες έχει ένα απεσταλμένο για τον έμπολα. Οι χώρε μόλις ε, διόρισαν το δικό τους πρεσβευτή, το Λουξεμβούργο το ίδιο. Και η Γερμανία διόρισε έναν απεσταλμένο. Όλοι αυτοί οι απεσταλμένοι ήρθαν στι χώρε μου, του δέχτηκαν ε, οι αρχηγοί κρατών μα και τώρα διόρισε έναν και Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό να υπάρχει ένα απεσταλμένο επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορεί να συντονίσει του υπόλοιπου και να υπάρχει ένα ενίο συντονισμό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι θα ήταν πολύ θετικό. Και πάλι σα ευχαριστώ πολύ. Εδώ πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω τη Ρογγελέρ Μαρόκ, τη Brussels Rice και την Air France, οι τρει εταιρείε που αποφάσισαν να μην μα απομονώσουν. Όλε οι άλλε μα μποϊκοτάρουν. Είμαστε ε, πραγματικά <laughs> σαν ε, πολίτες δεύτερη κατηγορίες, αλλά αυτές οι εταιρείες συνεχίζουν να έρχονται στις χώρες μας και τις ευχαριστούμε ειλικρινώς και ελπίζουμε ότι το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσουν να ενθαρρύνουν αυτές τις ε, εταιρείε να μην σταματήσουν τις πτήσεις. Και κάτι ακόμη για να κλείσω, τα μέσα μας και σε Έχουμε την εντύπωση ότι υπάρχει μια ιστερία, ένας φόβος, ένας πανικός που εγκαθίσταται. Είναι πολύ μεγάλο κρίμα. Νομίζω ότι τα ΜΜΕ θα πρέπει να προβούν σε αντικειμενική εξήγηση των πραγμάτων. Είναι καλό να μπορούν να μιλούν, να μπορούσαμε να μιλήσουμε και για τα μέτρα που έχουν ληφθεί για να αποφύγουμε τη διάδοση της επιδημίας σε άλλα μέρη του πλανήτη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριος Μουμάνη. Thank Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ αναζωογονητικό και πάρα πολύ ενθαρρυντικό το ότι ακούμε τις δηλώσεις ε, της Επιτροπής σας. Το θέμα του έμπολα έχει περάσει πλέον τα όρια του, της κατεπίγουσας κατάστασης για θέματα υγείας. Έχει καταστεί ένα θέμα αναπτυξιακό πλέον. Και οι χώρες που πλήττονται, οι τρεις χώρες της Δυτικής Αφρικής που πλήττονται, αποτελούν ε, χώρες που απειλούνται σημαντικά. Και θα πρέπει σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν να συζητήσουμε την πανδημία αυτή. Θα πρέπει σε αυτό το πλαίσιο να δημορφωθούν οι πολιτικές και οι απαντήσεις και οι στρατηγικές που χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό σε αυτή την κλίμακα. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερως. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να πω ότι συμφωνώ σε ό,τι αφορά την αποστολή πρέσβεων. Και χαιρόμαστε λοιπόν που είναι ο Επίτροπος ε, υπεύθυνο και δεν είναι κάποιος ε, άλλος ανεξάρτητος. Θέλω να είναι καλά σημαντικό το ότι επικεντρωνόμαστε σε αυτά. Ευχαριστώ. Τέθηκαν πολλές ερωτήσεις και θέλω να απευθυνθώ στον αδελφό από την Γενική Διευθυνσία Ανάπτυξη ότι θα του αφήσω την ερώτηση για το θέμα τη συμβατότητα με την δημοσιονομική στήριξη, γιατί αυτό είναι κάτι που έχει να κάνει με την αναπτυξιακή πολιτική και θα είναι οι συνάδελφοι που θα σας απαντήσουν για αυτό το θέμα. Κάποιες λέξεις κλειδιά που αναφέρθηκαν. Προβολή, συντονισμός, επικοινωνία, συντονισμός. Προβολή. Πρόκειται για μια πολλωστή κρίση και βλέπουμε ότι υποφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση από μεγάλο έλλειμμα προβολής. Ε, μία απόφαση που λήφθη από το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο ήταν να αυξηθεί το ποσό των δεσμεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή του κοινοτικού προϋπολογισμού και των κρατών μελών, προς υποστήριξη χωρών και πληθυσμών της περιοχής και από τα 600 εκατομμύρια ευρώ που ήταν ε, το ποσό πριν από το Συμβούλιο στο 1 δισεκατομμύριο στο τέλη του έτους. Σύμφωνα με τους τελευταίους υπολογισμούς που έγιναν την Παρασκευή ήδη Έχουμε φτάσει στα 900 εκατομμύρια σήμερα κοινοτικός προπολογισμό και κρατών μελών. Ποιος είναι ο αντίκτυπος ως προς την προβολή, πολύ μικρός. Πρόκειται για ένα διαρθρωτικό πρόβλημα που επανέρχεται. Δεν μπορώ να, θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερα από όσα είπαν οι κύριοι Γκέρενς και στη Πρέπει να βρούμε μια απάντηση και ίσως ο συντονιστής ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποτελεί μια αρχή επικοινωνία. Ο κύριος Πρεσβευτής αναφέρθηκε στην έννοια της ιστερίας. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ήρεμες, σοβαρές, ισορροπημένες πληροφορίες. Πρόκειται για ένα ανησυχητικό πρόβλημα, όμως ε, το έχουν αντιμετωπίσει οι μεγάλοι επαγγελματίε στην περιοχή αλλά και στις ευρωπαϊκές χώρες. Ε, αυτή ε, υπάρχει μια άλλη συζήτηση για τον έλεγχο στην είσοδο και στην έξοδο. Δεν έχω χρόνο, όμως όλα αυτά μας δείχνουν την κατάσταση. Θα πρέπει να πείσουμε τους επιβάτες ότι η έλεγχη ε, δεν είναι ένας τρόπος να προστατεύσουμε το φρούριο Ευρώπης, αλλά να προστατεύσουμε τους ίδιους τις οικογένειές τους, τα άτομα που συναντούν και ο καλύτερος τρόπος να εμποδίσουμε την έλευση του ιού εδώ είναι να το καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά στην πηγή και στις χώρες που έχουν πληγεί. Σε ό,τι αφορά το συντονισμό, να επενθυμίσω ότι ο κ. Τηλιανίδης διορίστηκε ε, ως απεσταλμένος από τους αρχηγούς ε, κρατών και κυβερνήσεων, όχι από την Κομισιόν. Δηλαδή το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον διόρισε απευθεία και όταν θα επιστρέψει θα μπορέσετε να συζητήσετε μαζί του. Νομίζω ότι είναι αυτό κάτι ε, που ε, θα βοηθήσει στο εγχείρημα του συντονισμού. Το είπε και ο κ. Στυνίδης. Είναι ένα εγχείρημα συντονισμού, όχι ελέγχου command and control. Για τα δημοσιονομικά δεν ξέρω Συγγνώμη, δεν πρόκειται να προλάβουμε, γιατί οι διερμηνείς μας έδωσαν 10 λεπτά παραπάνω. Είμαστε ήδη στα 10 λεπτά. Δεν ξέρω αν θέλετε να απαντήσετε στο κύριο Γκρέντς. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο. Δυστυχώς, πολύ, πολύ λυπάμαι, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Πολύ, πολύ λυπάμαι. Θα πρέπει να πάρετε το λόγο κάποια άλλη στιγμή. Αν θα μπορούσατε να απαντήσετε απευθεία για το θέμα αυτό, Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήλθατε και πολύ λυπάμαι που δεν πήρατε το λόγο. Θα κλείσω λοιπόν το θέμα, συνάδελφοι. Έχουμε στα διάφορα τα πρακτικά μια συνεδρίαση συντονιστών 7 Οκτωβρίου λοιπόν. Θα αναπευθεί στους συντονιστές και αυτό δούμε στην επόμενη συνεδρίαση. Η επόμενη συνεδρίαση είναι στην επόμενη εβδομάδα, 10-11 Νοεμβρίου. Σας ευχαριστώ, ευχαριστή ευγενικά η Πρόεδρος τους δερμηνείς και ζητώ συγγνώμη προς τους ε, συναδέλφους από την Γενική Διεύθυνση ΤΕΦΚΟ που δεν είχαμε χρόνο να τους ακούσουμε.